Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί συνάδελφε. Θα θέλαμε να αρχίσουμε στην ώρα μας και μάλιστα πρέπει να αρχίσουμε και στην ώρα μας γιατί αν είδατε την ημερήσια διάταξη θα είδατε ότι έχουμε να συζητήσουμε με διάφορους ε, επιτρόπους και με έναν γενικό γραμματέα που έχουν τόσο πολλά να μας πούνε που είμαι σίγουρη ότι θα έρθουν σοριδών οι συνάδελφοι και θα θέλουν να θέσουν ερωτήματα οπότε νομίζω ότι πρέπει να είμαστε τυπικοί με το χρονοδιάγραμμά μας. Θα έχετε λάβει την ημερήσια διάταξη. Υποθέτω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και να την εγκρίνουμε έτσι όπως είναι. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιος αντίρρηση. Σωστά. Ωραία. Οπότε πάμε στα πρακτικά. Τα εγκρίνουμε όπως πάντα. Εάν κάποιος δεν έχει πρόβλημα μέχρι, την μέχρι το τέλος της συνεδρίασης θα εγκριθούν. Δεύτερον, η συνεδρίασή μας και σήμερα το πρωί και σήμερα το απόγευμα θα, παρουσια... θα μεταδίδεται στο ίντερνετ οπότε να ξέρετε ότι τώρα ακούγεστε και σας βλέπει όλη η Ευρώπη ίσως και παρά έξω. Εάν προχωρήσει λίγο η συνεδρίαση και έρθουν όλοι οι συνάδελφοι και αν κάποιος που ενδιαφέρεται στις, για τις εργασίες της Επιτροπής μας αλλά δεν είναι ε, συνάδελφος και αν έρθουν τόσοι πολλοί που δεν έχουμε ε, άλλο χώρο εδώ μέσα Καλημέρα σας πείτε του να πάει στο 3G2. Υπάρχει ειδική αίθουσα και, για, και σήμερα, το απόγευμα, σήμερα το πρωί είναι ε, αυτή που σας είπα και σήμερα το ε, απόγευμα ε, θα είναι στον, ε, στον πρώτο όροφο για το απόγευμα, στον τρίτο όροφο και σήμερα το πρωί. Tagesordnung. Η ημερήσια διάταξη είναι πλήρης. Έχουμε να ακούσουμε τες, τρεις επιτρόπους, μία επίτροπο. Οπότε να είμαστε και συνεπείς. Και επιθαρχημένοι. Να σας πω πώς θα προχωρήσουμε. Δεν γίνεται να χαλάσουμε το πρόγραμμα, θα πρέπει να το τηρήσουμε όσο έχει. Λοιπόν, 5 λεπτά εισαγωγή από τον εισηγητή, 10 λεπτά δήλωση και όταν λέω 10 λεπτά εννοώ 10 λεπτά για τον κάθε επίτροπο και μετά 35 λεπτά για τις πρώτες ε, δηλώσεις από, τους, από τις ε, ομάδες. Μετά θα δούμε πόσους ομιλητές θα έχουμε στον κατάλογο των ομιλητών. Θα δούμε πόσοι μπορούν να μιλήσουν. Βέβαια δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο σήμερα. Και τέλος θα ξαναλάβει το λόγο ο Επίτροπος για 5 ή 10 λεπτά για να μπορέσει να απαντήσει ή να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Είναι σαφές και μας το, υποσχέθηκε, μας το υποσχέθηκαν όλοι οι επίτροποι, εάν υπάρξουν κάποιες ερωτήσεις που πρέπει να τεθούν και δεν προλάβετε να τις θέσετε ή να απαντηθούν στη σας σήμερα, θα απαντήσουν γραπτός. Αυτά για τα τυπικά της συνεδρίασης. Η επόμενη συνεδρίαση είναι στις 10 Φεβρουαρίου. Θα είναι ο Επίτροπος Χάν και ο Επίτροπος Άντρος μαζί μας. Σε εκείνη τη συνεδρίαση χαιρόμαστε ιδιαίτερος. Θα είναι μισή μέρα εκείνη τη συνεδρίαση για να μπορέσουμε να συζητήσουμε με τους δύο αυτούς επιτρόπους. τα υπόλοιπα μπορεί να έχετε λάβει, μπορεί και να τα λάβετε σήμερα. Έχουμε, ε, έχει ζητηθεί από τους προέδρους των επιτροπών, έχει σταλεί μάλλον μια πρόσκληση από, τους, ε, από την διάσκεψη των προέδρων προς τον ε, πρόεδρο, να, προς εμένα δηλαδή, να κάνουμε μια παρέμβαση για την Σύνοδο Κορυφής Το συζητήσαμε και με τους συντονιστές και στείλαμε το σχέδιο στις ε, ομάδες. Νομίζω ότι έχουν συμπεριληφθεί όλα όσα ήθελαν οι ομάδες και εφόσον συμφωνείτε θα στείλαμε την απάντησή μας στον ε, Κλάους Χάινα Θα το δείτε και στους φακέλους σας κανονικά. Και αυτό που είπα στους συντονιστές θα ήθελα να το πω και εδώ. Δεν, ε, αυτό που έχουμε εδώ εμείς ως κείμενο σίγουρα δεν αντικατοπτρίζεται πλήρως λέξη-λέξη στο ψήφισμα. Αυτό που εμείς γράψαμε είναι μία παρέμβαση για την συνεδρίαση των, ε, για τη διάσκεψη των Προέδρων. Μετά θα γίνει μια συμπερίληψη όλων των απόψεων και αυτό το κείμενο θα πάει στην διάσκεψη των Προέδρων για να αποτελέσει το ψήφισμα. Οπότε μην απογοητεύεστε εάν δεν είδατε κάτι που έχει, να μην έχει συμπεριληφθεί, ακόμη και αυτοί που ήσασταν στην όλη συντακτική εργασία. Από την πλευρά μας επίσης έχει αποσταλεί σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια μια επιστολή σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όντως λάβαμε κάποιες ε, απαντήσεις από κάποια κοινοβούλια. Οι απαντήσεις αυτές ήταν στη γλώσσα του κάθε κοινοβουλίου βεβαίω, δικαίωμά του βέβαια. Απλώ τώρα θα πρέπει να περάσει κάποιο χρόνο για να τα μεταφράσουμε ώστε να είμαστε όλοι σε θέση να καταλάβουμε τι λένε τα, οι απαντήσει των κοινοβουλίων. Έχουμε την δανέζικη απάντηση στα δανέζικα, καταλαβαίνετε. Πρέπει να τα μεταφράσουμε για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Και στο τέλος της εβδομάδας νομίζω ότι θα μπορέσουμε έτσι να έχουμε έτσι ένα κείμενο συνεκτικό με όλες τις ε, ε, απαντήσεις και όταν θα έρχεται μια νέα απάντηση θα συμπληρώνεται. Αυτά για τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και όλες οι επιτροπές του ζήτησα εάν θέλουν να κάνουν κάποια παρέμβαση στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή SURE, παρακαλούμε να το κάνουν είτε με επιστολή, είτε μέσω μιας γνωμοδότησης. Υπάρχουν κάποιες γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής ε, Μεταφορών και της Επιτροπής Ανάπτυξης, οι οποίες ήδη έχουν εγκριθεί, μάλιστα πολύ άμεσα ώστε να μπορέσουμε να έχουμε την τελική εκδοχή των γνωμοδοτήσεών τους. Η Επιτροπή Βιομηχανίας και Έρευνας ε, ψήφισε, αλλά δεν έχει τελειοποιηθεί ακόμη η τελική εκδοχή του κειμένου. Οπότε σήμερα θα έχουμε αυτή την μη ε, τελική εκδοχή του κειμένου, σήμερα το απόγευμα. ώστε να έχουμε όταν θα συζητήσουμε με τον Επίτροπο για την έρευνα και την ε, ε, εκδοχή του κειμένου από την Επιτροπή. Επίσης, η Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων ψήφισε την, ε, την, θα ψηφίσει την Πέμπτη, συγγνώμη, και, και άλλη μια Επιτροπή θα ψηφίσει σήμερα, οπότε θα έχουμε άλλες δύο παρεμβάσεις. Να έχουμε, θα έχουμε δύο επίσημα κείμενα λοιπόν. Η Επιτροπή Πολιτισμού επίσης περιμένουμε και η Επιτροπή Γεωργίας θα περιμένουμε να έχουμε την ε, τελική εκδοχή και τη σωστή εκδοχή των κειμένων τους. Αυτά ε, για τις δικές μου ανακοινώσεις. Μην κοιτάτε εκείνο το ρολόι, δεν πάει καλά. Δεν πάει καθόλου καλά, ούτε το ένα ούτε το άλλο το ρολόι. Πάνε καλά. Δύο ρολόγια έχουμε και τα δύο πάνε πίσω. Δείτε το ρολόι σας ο καθένας για να ξέρουμε τι ώρα, τι ώρα είναι. Λοιπόν, είμαστε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Σημείο 4 λοιπόν. Για το σημείο 4 Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Επίτροπο, τον Επίτροπο Έτινγκερ. Χαίρομαι που βρήκατε σήμερα χρόνο να έρθετε στην Επιτροπή μας. Δεν είναι εύκολο να συνδυαστούν πάντα τα προγράμματα όλων. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Θα προχωρήσουμε όπως σας είπα από την αρχή. Θα Έχουμε πέντε λεπτά μια μικρή παρουσίαση από τον εισηγητή μας και μετά θα σας δώσουμε το λόγο για 10 λεπτά για να κάνετε την παρουσίασή σας, την παρέμβασή σας και μετά θα κάνουμε την ε, συζήτηση. Παρακαλώ, Σαλβαδόρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, Επίτροπε. Καλώς ήρθατε, συνάδελφοι. Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για την Επιτροπή μας, διότι προβλέπονται στο πρόγραμμα επισκέψεις από τρεις επιτρόπους και μάλιστα για τομείς ε, σημαντικότατους για μας, που αφορούν τις μελλοντικέ δημοσιονομικές προοπτικές, ιδιαίτερως για την έρευνα, τις μεταφορές και την ε, ενέργεια. Ξέρουμε ότι ούτως ή άλλως θα Έχουμε πάντοτε περισσότερε απαιτήσει για την εξωτερική μα δράση και τη χρηματοδότησή μα, αλλά ω προ την επίσκεψη του Επιτρόπου για την Ενέργεια. Ξέρουμε ότι θα έχει πολλά να λάβει υπόψη του Επιτροπό σε σχέση με τι μελλοντικέ δημοσιονομικέ προοπτικές. Θέλαμε λοιπόν να ξέρουμε την άποψή του, ε, τα, τις του, το πώ αντιλαμβάνεται την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κοινοβουλίου προκειμένου να κατανεμηθούν οι πόροι ε, βάσει των ερχόμενων των μελλοντικών δημοσιονομικών προοπτικών. Λόγω των νέων αρμοδιοτήτων του ε, βάση της συνθήκης της Λισαβόνας διαθέτουμε πλέον μια νέα νομική βάση. Νέα νομική βάση που θέτει συγκεκριμένους στόχους για την ενεργειακή μας πολιτική ιδιαίτερα φιλόδοξους. Το Κοινοβούλιο λοιπόν διαβλέπει την ανάγκη να αναλυθούν νέε δεσμεύσει, ε, ιδίω προ τι δαπάνε. Αυτό βάσει των σημερινών ε, προοπτικών δεν προβλέπεται ακριβώς. Ε, η Επιτροπή Σούρε προκειμένου να εξεύρει την, προστιθέμενη ευρωπαϊκή, την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία Πρέπει να λάβει υπόψη όλο τον ενεργειακό σχεδιασμό που χρειάζεται, την δημιουργία νέων υποδομών. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν πλέον σε κοινοτικό επίπεδο, διότι θεωρούμε ότι θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό κάτι τέτοιο. Και το να επικεντρωθούμε σε κοινοτική χρηματοδότηση, κοινοτικό προπολογισμό για όλε αυτέ τι πρωτοβουλίε είναι προτιμότερο από το να έχουμε 27 διαφορετικέ ενεργειακέ πρωτοβουλίε σε κάθε κράτο μέλο. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε την τοποθέτηση του Επιτρόπου που ασχολείται με τα θέματα ενέργεια σε αυτόν τον τομέα. Είναι προφανέ ότι θα χρειαστούμε νέα δημοσιονομικά κονδύλια, νέου πόρου που θα πρέπει προφανώς να ξεπεράσουν τα σημερινά όρια. Και εδώ έχουμε δύο διαφορετικές ε, δυνατότητες. Πρώτα απ' όλα, ως προς τα ζητήματα της ενέργειας ε, και ως προς τις ε, κύριες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να προβλέψουμε τάσεις ευθυγράμμισης, mainstreaming. και δύο ενεργειακές κατευθύνσεις κυρίως, βάσει των οποίων να μπορέσουμε να εξεύρουμε τα απαραίτητες, απαραίτητες γραμμές δαπανών κατά τη χρήση των κονδυλίων από τον προπολογισμό ή εκτός προπολογισμού. Κατά πρώτον κύριε Επίτροπε, θέλαμε να σας ρωτήσουμε τι κατά την άποψή σας είναι απαραίτητο να γίνει τα ερχόμενα χρόνια ως προς τους δημοσιονομικούς πόρους. Θεωρείτε ότι είναι δυνατόν οι επενδύσεις, οι ενεργειακές να κατανεμηθούν σε διαφορετικά κεφάλαια του σχεδίου προπολογισμού. Κάπου γίνεται λόγος για ένα εκατομμύριο ευρώ. Μάλλον ένα 3 ε, ευρώ, λέει ο για τον ε, ορίζοντα το 2020. Ως προς τις υποδομές, τις ενεργειακές και όλα τα άλλα κεφάλαια που έχουν σχέση με την ε, ενέργεια. Η Ευρωπαϊκή Επίτροπη ελπίζει να λάβει πόρους από ιδιωτικού φορεί Όμως μας μιλάει και για την ανάγκη να παρέμβουμε στο επίπεδο των ε, κρατικών φορέων. Τι εννοούμε λοιπόν με αυτό το 3 ευρώ. Τρίλιον euros λέει ο, ο μιλητής. Θεωρεί η Επιτροπή ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα ειδικό ταμείο για την ενέργεια, ένα ειδικό κονδύλι εκτός προπολογισμού που να μην περιλαμβάνεται απευθείας στις δημοσιονομικές προοπτικές και το οποίο να πρικοδοτείται από κοινοτικέ διαδικασίες και όχι ενδοκυβερνητικές ή διακυβερνητικές. Ε, βάσει των σημερινών δημοσιονομικών προοπτικών για τα ενεργειακά ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπονται 155 εκατομμύρια στο υπάρχον χαρτοφυλάκιο. Κατά την άποψή σας αυτό απαρκεί για να υλοποιηθούν οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες, δηλαδή οι διασυνδέσεις σε επίπεδο ενέργειας που ακόμη μας λείπουν. Ή πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια δημοσιονομική πιο εντατική για τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές. Και τέλος, το έλλειμμα ως προς την ενέργεια. Εδώ παραμένουν κάποιοι ενδιασμοί. Πιστεύετε, καθότι υπάρχουν και κάποιες μελέτες που εκπονήθηκαν από το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πιστεύετε ότι μπορούμε να φτάσουμε τα ποσοστά του 20%? Πιστεύετε ότι θα είναι αρκετό να αλλάξει η νομική βάση ή θα πρέπει να προβλέψουμε νέους δημοσιονομικούς πόρους. Για την ενεργειακή αποδοτικότητα δεν θα πρέπει να προβλέψουμε κάποιους υποχρεωτικούς στόχους. Επίσης κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερως και τους συναδέλφους της Επιτροπής Ήτρε. Για τις ευφυείς e τεχνολογίες θα πρέπει αυτά να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα SIP CIP ή να μετατραπούν εξ ολοκλήρου και να υπάρχουν υποδομές τελείως ανεξάρτητες σε σχέση με το ευρύτερο πρόγραμμα CIP. Ιδού, Πρόεδρε, πρώτες μου ερωτήσει για να ξεκινήσει όλη η συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Σαλβαντόρ. Ο κύριος Σότιγκερ, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμε κύριε εισηγητά, κυρίες και κύριες ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε ήδη εγκαίρως να συζητήσουμε για βασικά θέματα ε, διαρθρωτικά όσον αφορά την επόμενη περίοδο ε, και ιδίως ε, να συζητήσουμε τις έξυπνες και πολύ ουσιαστικές ερωτήσεις τις οποίες έχει θέσει ο εισηγητής. Θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση είναι μία πρώτη συζήτηση γιατί η Επιτροπή ακόμη προετοιμάζει το σχέδιό της και γίνονται συζητήσεις οι οποίες θα συνεχίσουν το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Οπότε ε, καταρχήν έχουμε να κάνουμε με μακροπρόθεσμες μα δημοσιονομικές ε, δομές ε, τις οποίες αξιολογούμε για να δούμε αν πρέπει να τις συνεχίσουμε ή όχι. Δεύτερον, επιμένουμε στο ειδικό πρόγραμμα ενάντια στην κρίση σαν συγκυριακό πρόγραμμα με τα μέσα και με τα προγράμματα τα οποία έχουν διατηρηθεί τεθεί από το Κοινοβούλιο για να δούμε εάν θα πρέπει να εκπνεύσουν μετά από τρία χρόνια ή αν θα πρέπει να συνεχιστούν και στην επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Τέλος, εξετάζουμε το νέο άρθρο 194, δηλαδή την τον εξευρωπαϊσμό της ενεργειακής πολιτικής με νέα βασικά σημεία ή με ε, ουσιαστικά βασικά σημεία τα οποία πρέπει ε, να καθορίσουμε για την ενέργεια. Και τέλος, στα τελευταία χρόνια είχαμε καταρτήσει α στόχους, δηλαδή μία αύξηση της αποδοτικότητας ενεργείας κατά 20%, ένα συγκεκριμένο ποσοστό ανανεωσίμων πηγών ενεργείας, οι οποίες επίσης θα πρέπει ε, ε, να, ε, οι οποίες έχουν επίσης περιληφθεί εις τον προϋπολογισμό. Δηλαδή είναι διάφορα προγράμματα τα οποία πρέπει ακόμη να καταστήσουμε πιο ουσιαστικά και να συμπληρώσουμε. Δηλαδή καταρχήν πρέπει να δούμε δούμε τι, ε, ε, ε, τι συνεπάγεται χρηματοδότηση από τον προπολογισμό και πού χρειάζονται ομόλογα τα οποία θα πρέπει να διοχετευτούν. Δηλαδή υπάρχει μία συνεργία μεταξύ της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, της αναπτύξεως, της βιωσιμότητος και της προστασίας του περιβάλλοντος διότι έχουμε το πρόγραμμα ε, το ενεργειακό για το 2020 το οποίο καθορίζει πέντε βασικά σημεία εκ των οποίων θα πρέπει να διατηρήσει κανείς μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Δηλαδή ε, ε, όποιος θα επενδύει ένα ευρώ την Ευρωπαϊκή Ένωση θα του θα έχει μεγαλύτερη απόδοση από ό,τι στα μεμονωμένα ε, κράτη-μέλη. Και γι' αυτό πιέζουμε βάσει της προεργασίας μας το Συμβούλιο χωρίς όμως να ζητάμε περισσότερες προσπάθειες ε, από τα κράτη-μέλη για να επιτύχουν ε, το 20% αυξήσεως της αποδοτικότητας στην επόμενη δεκαετία όπου αυτή δεν προχωρά σωστά. Αυτό που πρέπει να εξετάσουμε είναι πού και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι για, ε, τα, να προοδεύσουμε, δηλαδή ε, για τα κτίρια, για τα ιδιωτικά κτίρια αλλά και για τα δημόσια κτίρια, διότι στα διάφορα κράτη έχουμε διαφορετικές ε, εμπειρίες από την ανακαίνιση των οικοδομών και αντιλαμβάνομαι τα περιφερειακά ταμεία και τα ταμεία συνοχής θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν για την ενεργειακή αποδοτικότητα και την ανακαίνιση των κτηρίων σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη για τη βελτίωση των ιδιωτικών και δημοσίων κτηρίων και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει ένα βασικό θέμα που θα στηριχθεί από το Ταμείο Συνεχής. Δηλαδή δηλαδή να υπάρξει μία μετατόπιση της ευθύνης για την ε, ενεργειακή αποδοτικότητα και γι' αυτό προσβλέπω με την Επιτροπή σας σε έναν αποδοτικό διάλογο. Επίσης η εσωτερική αγορά θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, δηλαδή να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, την ε, ασφάλεια, τις ε, ανεκτές ανανεώσιμες πηγές ενεργείας, οποίε μπορούμε να πληρώσουμε, την ανταγωνιστικότητα, διότι αν δεν υπάρχουν υποδομές δεν θα τα καταφέρουμε. Πρέπει λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε προς ε, μη ε, ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ενεργειακό για το αέριο και το πετρέλαιο. Υπάρχουν όμως ορισμένα τιμία, σημεία της υποδομής τα οποία δεν έχουμε υπολογίσει επαρκώς ή που απαιτούν πάρα πολλά από τους ιδιώτες. Δηλαδή θα πρέπει να συμπεριλάβουμε ε, ορισμένες μεμονωμένες αγωγές οι οποίες ε, ε, δεν ε, συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στο σύστημα τα κράτη της Βαλτικής παραδείγματος χάρη και θα χρειαστεί επίσης αλληλεγγύη στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για του, τους interconnectors αλλά επίσης στο, ε, στο ενεργειακό πρόγραμμα θα πρέπει να κοιτάξουμε να αξιοποιήσουμε τις καλές εμπειρίες που έχουμε ε, με βάση ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος ε, για να μπορέσει μια σωστή ε, ε, υποδομή για τα επόμενα χρόνια. Πρέπει λοιπόν στον τομέα αυτό των επενδύσεων στην υποδομή να δούμε πώς θα τη θέσουμε στο επίκεντρο μίας χρηματοδοτικής προσπάθειας μέσω δανεισμού με, ε, νέες με άλλες διαρθρωτικές τράπεζες των κρατών μελών διότι ε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ε, συμμετοχή ε, όλων στη χρηματοδότηση αυτή. Επίσης όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη, την καινοτομία στον ενεργειακό τομέα διότι το πρόγραμμά μας ε, ε, είναι ουσιαστικό θα πρέπει να ακολουθήσουμε την ίδια τεχνολογική εξέλιξη να δούμε όμως που μπορεί να υπάρξει συγχρηματοδότηση ή με ε, πλειοψηφική χρηματοδότηση για να επέμβουμε και στη διοίκηση ε, των ε, επιχειρήσεων. Το ΙΤΡΕ, ξέρουμε ότι το ΙΤΡΕ είναι ένα αμφιλεγόμενο πρόγραμμα, το ξέρουμε. Αλλά πρέπει να αποδείξουμε με το ΙΤΡΕ ότι η Ευρώπη σε μεγάλα προγράμματα αναγνωρίζεται και από τους ομολόγους της όπως η Αμερική και η Κίνα και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε μία μακροπρόθεσμη δέσμευση στο τι αξίζει το Ίτρε κατά τρόπον ώστε να μην ε, συναγωνίζεται τα άλλα ερευνητικά ιδρύματα και όλα να είναι ισότιμα μέσα στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δηλαδή δεν ασχολείται μόνο το Ίτρε με την ενεργειακή έρευνα αλλά ασχολείται και θα προωθείται στα πλαίσια της συνεργασίας των κρατών μελών με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να δούμε ε, τι θα γίνει με αυτό το φιλόδοξο εγχείρημα διότι θα πρέπει να ε, βρούμε έναν ε, τρόπο με τον οποίο να προχωρήσουμε και να περιλάβουμε τα διάφορα προγράμματά μας στην επόμενη δημοσιονομική περίοδο και τέλος όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Η σχέση μας με, και, με, ε, και τη σχέση με τις τρίτες χώρες, η σχέση με την Τουρκία, με τη Ρωσία, με το χώρο της Κασπίας ε, μπορεί να προωθηθεί και να βελτιωθεί με κοινά προγράμματα ε, στα επόμενα χρόνια. Δηλαδή ε, υπάρχουν προγράμματα στα οποία η συγχρηματοδότηση θα είναι ευρωπαϊκή διότι το κράτος το οποίο είναι παραμεθόριο προς μία τρίτη χώρα δεν μπορεί να παραβλέψει ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή υπεραξία την οποία πρέπει να επιτύχουμε με αυτές τις συνεργασίες. Γι' αυτό και ε, θα πρέπει να υπάρξει μια προεργασία και ε, θα ήταν καλό το Μάιο ή τον Ιούνιο να κάνουμε μια συζήτηση με τον εισηγητή για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε τις συζητήσεις του φθινοπόρου για τον προπολογισμό. Τώρα ξεκινάμε μια συζήτηση και ε, ο κύριος ο... είναι ο εισηγητής για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την παρέμβασή του. Δύο πράγματα θα ήθελα να πω. Και θα ήθελα αν μπορεί ο Επίτροπος να σκεφτεί, να τα σκεφτεί λίγο το ελάχιστο και το μέγιστο. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε το ελάχιστο για να πετύχουμε το μέγιστο. Γιατί έχουμε νέες προσδοκίες, ας πούμε, για τις υποδομές. Πρέπει να σκεφτούμε πώς θα ελαχιστοποιήσουμε ε, την προσπάθεια για να επιτύχουμε τα μέγιστα αποτελέσματα. Ας πούμε, οι νέες φιλοδοξίες. Καλό θα ήταν να ακούσουμε την δική σας άποψη για το τι θεωρείτε ότι είναι οι νομικές συνέπειες της νέας συνθήκης. Και επίσης, το πακέτο για την αγορά ενέργειας που έχουμε αποφασίσει πριν από ένα χρόνο ε, και για τη διασυνοριακή συλλογή κτλ. Για τις διασυνοριακές συνδέσεις λοιπά. Θα ήθελα επίσης να μας πείτε δύο πράγματα για τις παλαιές φιλοδοξίες μας. Γιατί συνήθως μιλάμε για τις νέες, για τα μελλοντικά μας σχέδια. Ίσως ε, κάποια από τα παλαιά σχέδια τελικά να μην είναι τόσο σημαντικά πλέον. Οπότε θα, δεν ξέρω αν θα μπορούσατε βέβαια να πείτε κάτι τέτοιο χωρί δικηγόρο δίπλα σα, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν μπορείτε, νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε το θάρρο να μιλούμε όχι μόνο για το μέλλον, για τα μελλοντικά μα σχέδια, αλλά και πώ θα κάνουμε το phase out όλων όσων στο παρελθόν είχαμε ε, σχεδιάσει και τα οποία μπορεί να μην είναι πια επίκαιρα. Γιατί εκεί και εκεί έγκυται το ελάχιστο και το μέγιστο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Σε σχέση λοιπόν με αυτέ τι νέε φιλοδοξίε, τι γίνεται με τις παλαιές και πόσο θαραλέος μπορείτε να είστε ώστε να αποσύρετε κάποιες από τις παλαιές φιλοδοξίες. Επίσης για τις υποδομές. Περνούν σε μια νέα φάση με την νέα νομοθεσία που έχουμε για την αγορά ενέργειας. Γιατί νομίζω ότι αυτό ήταν μια, ένα σημαντικό τομέα όπου μπορούμε να έχουμε διασυνοριακές συνδέσεις και καλύτερα ευρωπαϊκό δίκτυο. Αλλά εσείς πώς μπορείτε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα αντικαταστήσουμε την εθνική χρηματοδότηση που θα μπορούσε να συμβαίνει σε άλλε περιπτώσει, ή την εμπορική χρηματοδότηση. Γιατί και εκεί πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα είναι επιπλέον. Πρέπει επίση να εξασφαλίσουμε ότι θα περιορίσουμε τη χρήση του. Γιατί αλλιώ ο κίνδυνο αντικατάσταση τη ιδιωτική και τη εμπορική χρηματοδότηση είναι μεγάλο. Οπότε σημαίνει ότι εμεί δεν θα έχουμε το ίδιο ε, αντιστάθμισμα. Και επίση για την ενεργειακή απόδοση. Είπατε ότι η ενεργειακή απόδοση έχει σχέση για τα κτίρια κτλ. Ε, το πιο φυσιολογικό είναι ότι τα κτίρια είναι όλα ένα τμήμα της, των ιδιωτικών επενδύσεων και των ανανεώσεων, γιατί όλο βλέπουμε να ανακαινίζονται κτίρια κτλ. Εσεί πώ μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι όταν θα δαπανίσουμε χρήματα και εφόσον το κάνουμε, ε, θα το κάνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να ε, έχουμε μια επιπρόσθετη αξία και να μην αντικαταστήσουμε αυτές τις επενδύσεις. Νομίζω, Πρόεδρε, ότι αυτός ο τομέας είναι πάρα πολύ ιδιαίτερος όταν μιλούμε για την ενέργεια, γιατί βασίζεται σε μια πολύ φυσιολογική, δομημένη εμπορική διαδικασία. Οπότε ό,τι κάνουμε μπορεί όντω να έχει σημαντικέ συνέπειε. Είτε στη χειρότερη περίπτωση θα αντικαταστήσουμε αυτό που υπάρχει τώρα, αλλιώ στην καλύτερη και αν είμαστε αποτελεσματικοί θα, θα κάνουμε κάτι επιπλέον των όσων γίνονται τώρα. Επίση, Πώς θα εξασφαλίσετε ότι μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα και την ανάπτυξη στα πλαίσια των κονδυλίων που έχουμε και σε ποιες θα είναι οι προτεραιότητες που θα λάβουν, ε, δεν θα λάβουν τόσο υψηλή θέση για σας. Ποιες είναι λοιπόν οι όχι και τόσο σημαντικές ε, προτεραιότητες ώστε να επιτύχουμε τις πολύ σημαντικές προτεραιότητες, να μειώσουμε την, ε, τις δαπάνες ώστε να μην αντικαταστήσουμε την ιδιωτική ή την εθνική χρηματοδότηση. Αυτά πρόεδρε, ευχαριστώ. Ja, Dank, ähm, Jetzt... Εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Κάλφιν έχει το λόγο. Thank you very much, uh, Madam. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε που Μα κάνατε αυτή την διεξοδική παρουσίαση για να αρχίσει η συζήτησή μα. Εκ μέρου τη δική μου τη ομάδα ήθελα να σα πω ότι σε γενικέ γραμμέ ε, στηρίζουμε τη στρατηγική που πρότεινατε για την ερχόμενη δεκαετία για την Ευρώπη. Στρατηγική που συζητήθηκε και στο Συμβούλιο αυτή την εβδομάδα. Οι σοσιαλιστέ μου λένε ότι. Λένε, μάλλον υποστηρίζουν ότι έχουμε δύο μέγιστε προκλήσει στην Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα να μειώσουμε την εξάρτηση από τα εισαγόμενα ρεκτά καύσιμα και έπειτα να περιορίσουμε την εκπομπή του διοξιδίου του άνθρακα, τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Εδώ έχουν προταθεί διάφορες λύσει και χαίρομαι ιδιαίτερω που βλέπουμε τις περισσότερες, πολλέ από αυτέ τουλάχιστον, στα στρατηγική που προτείνεται. Όμως, θα πρέπει να σκεφτούμε και πέρα από το 2020. Διότι όταν μιλάμε για εισαγωγή όλων αυτών που αναφέρετε και εσείς στρατηγική σα, τι εννοούμε. Θα πρέπει να υπάρχει μια τεράστια μεταλλαγή, μια πραγματική καμπή στη χρήση των ε, ενεργειακών υποδομών. Σε όλες τις υποδομές, τις μεταφορικές και τις ενεργειακές. Ε, και πάλι, νομίζω ότι αν ε, βλέπουμε πέρα από τον ορίζοντα του 2020, αν σκεφτούμε τι θέλουμε να πετύχουμε μέχρι το 2020, αλλά έχουμε κατά νου και πώς θέλουμε να διαρθρώσουμε γενικά το χώρο της ενέργειας, θα πρέπει να είμαστε πραγματικά διορατικοί. Νομίζω για παράδειγμα, ότι ο στόχο για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. το ποσοστό που έχουμε θέσει μπορεί να το πετύχουμε αρκετά εύκολα στο 2020, αλλά ίσως πρέπει να είμαστε αρκετά πιο φιλόδοξοι. Τα επιστημονικά πορίσματα λένε ότι μέχρι το 2050 θα πρέπει ίσως να στοχεύουμε 90% λιγότερη εξάρτηση. Για την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τα άλλα, νομίζω ότι δεν είμαστε ακόμη αρκετά φιλόδοξοι καθυστερούμε και ο στόχο που έχουμε θέσει δεν είναι υψηλό. Θα πρέπει και για την ενεργειακή απόδοση επίση να σκεφτούμε το ίδιο. Είναι πολύ απογοητευτικά τα αποτελέσματα που έχουμε θέσει ω στόχους για το 2020. Εδώ νομίζω ότι χρειάζονται δεσμευτικοί στόχοι και να σκεφτόμαστε πέρα από τον ορίζοντα του 2020, αν θέλουμε να πετύχουμε το 40% μέχρι το 2040. Εδώ δεν θα μιλήσω για την κοινή ενεργειακή αγορά, παρόλο που όπως είπατε έχει πάρα πολύ σημασία για τις επενδύσεις και τις κοινέ υποδομές, για την ενεργειακή όμως πολιτική και τις ε, προσπάθειες να διασυνδέσουμε τις ε, ευρωπαϊκές υποδομές με τα ευφύ δίκτυα, τις ευφύς λύσεις. Εκεί λοιπόν στη στρατηγική υπάρχει μια έλλειψη. Δεν βλέπω πώς θα γίνει μετάβαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην ενεργική πολιτική. Νομίζουμε ότι περίπου 50-100 εκατομμύρια πολίτε στην Ευρώπη καθημερινά αντιμετωπίζουν προβλήματα ενεργειακής ένδυα ή δυσκολίας να χρησιμοποιήσουν του ενεργειακού πόρου. Θα έλεγα λοιπόν ότι πρέπει και πάλι και σε αυτό το θέμα να σκεφτούμε και πέρα από τον οριζόντα του 2020. Και κάτι που μόλις είπε και ο συνάδελφος. Ε, έχουμε υπερβολικά πολλές προτεραιότητες στο ίδιο όμως επίπεδο στη στρατηγική. Και δεν κάνετε αρκετό λόγο για τη χρηματοδότηση, για, τα, για τους πόρους, τα κονδύλια. Αυτό που μόλις μας είπατε και αναφέρεται αυτό και ότι στρατηγική, είναι ότι θα υπάρξει ένα τρεις επενδύσεων ως το 2020. Δεν έλαβα όμω σαφή απάντηση στην. Ε, δεν λάβαμε σαφή απάντηση στην ερώτηση του του συναδέλφου. Πώ προβλέπετε ότι θα συγκεντρωθούν αυτά τα κρατικά, τα δημόσια κονδύλια. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αφήσουμε κατά μέρο τι ιδιωτικέ επενδύσει, όμω κάπω θα πρέπει να κάνουμε ελέγχο και για το δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2013. Και το βάρο που θα πρέπει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίω. Και κατά δεύτερον, εάν Θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Πώς θα διανεμηθεί, πώς θα γίνει η κατανομή μάλλον των δημόσιων δαπανών μεταξύ ευρωπαϊκού και κρατικού προπολογισμού. Μιλάτε για για upfront, upfront loading στην περίπτωση του προπολογισμού. Πώς θα γίνει αυτό και πότε θα ξεκινήσει προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας. Και επίσης για τα τελείως καινούργια χρηματοδοτικά μας μέσα. Μιλήσατε για τα ευρωμόλογα. Θα ήθελα περισσότερα σχόλια όμως και μιλήσατε για το σύστημα ανταλλαγής δικαιωμάτων εκπομπών. Ο φόρος για τον άνθρακα, για, το, για τις εκπομπές ή ο διαχωρισμός επενδύσεων στην ενέργεια σε ξεχωριστό κεφάλαιο ο εισηγητή μίλησε για άλλο κονδύλι. Εδώ ίσως θα πρέπει στο ίδιο κεφάλαιο να ξεχωρίσουμε τις κατηγορίες ώστε να είμαστε σαφεί στο τι εννοούμε όταν μιλάμε για ενέργεια. Αν χρησιμοποιήσουμε τα ιδρυθετικά κονδύλια, αυτό σημαίνει ότι αυτό θα γίνει βάρος άλλων προτεραιοτήτων σε συγκεκριμένε περιοχέ. Το ξέρω. πρέπει να είμαστε πολύ πειθαρχημένοι. Το ξέρω ότι όταν παθιάζεστε ξεπερνάτε λίγο το όριο το χρονικό, αλλά επειδή έχουμε πολλά ερωτήματα και κοιτάω και το ρολόι, ε, πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι. Αλεξάνδρ, ξέρω ότι θα αρχίσουν τα πέντε λεπτά να μετράνε δυστυχώς από σένα. Λυπάμαι, αλλά... Ε, συνήθως ο τρίτος την πληρώνει. Ευχαριστώ. Εντάξει, μην ανησυχεί. Εμεί ε, οι φιλελεύθεροι είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοια. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα α, να ξέρω ότι θα έχουμε πολλοί συνάδελφοι ερωτήματα και ήδη κάποιοι από αυτού που μίλησαν είπανε κάποια πράγματα. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που μάλλον δεν θα μπορέσω να περιμένω την απάντησή του από τον κύριο Επίτροπο γιατί πρέπει να παρουσιάσω ένα ερώτημα σε μια άλλη επιτροπή εκ μέρους τη ομάδα μου. Ε, είπατε ε, σωστά ο, και στην αρχή για την εξάρτηση της Ελλάδας από τους παρόχους ενέργειας εκτός Ευρώπης, Ρωσία, ε, Αλγερία, άλλα, άλλα κράτη, από αέριο. Ε, και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τη δική σας ε, ηγεσία προσπαθεί να εκπονήσει προτάσεις για το πώς μπορούμε να είμαστε ανεξάρτητοι από την ενέργεια και να έχουμε δική μας ενεργειακή απόδοση με, βλέμμα, με το βλέμμα μας το 2020 για να ε, ναι, επιτύχουμε και, την, και τους στόχους ενέργειας και του κλίματος. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εμπλακεί ενεργά σε όλη αυτή τη διαδικασία ώστε να υπάρχει ένα αυτόνομο ευρωπαϊκό δίκτυο. Ε, το είπατε και για μας ε, είναι πολύ σημαντικό ότι μέχρι το 2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δαπανίζει ένα τρισεκατομμύριο ε, ευρώ αυτό είναι πάρα πολύ περισσότερο από αυτά που, δίνουμε, που δίνει το ε, χρηματοδοτικό πλαίσιο, για να μην μιλήσω για το τι θα γίνει μέχρι τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερώτημα λοιπόν, πώς ακριβώς θα, θα χρηματοδοτηθεί αυτό το ποσό, ακόμη και αν μιλούμε για δάνεια. Με κάποιο τρόπο θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν αυτά τα δάνεια, να καταβληθούν, να πληρωθούν. Οπότε θα πέσουμε έξω στον προπολογισμό μας. Παρ' όλα αυτά, αυτό θα είναι σημαντικό και για αυτούς που θα αγοράσουν εκείνο το δάνειο. Οπότε μέχρι το 2020 εσείς πώς ακριβώς θεωρείτε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε στα χέρια μας αυτό το πόσο που χρειάζεται. Ευχαριστώ. Επόμενος, εκπρόσωπος των Πρασίνων. Thank you, Mrs. Chair. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ τα δύο λεπτά που μου άφησαν οι φιλελεύθεροι. Περίσευμα. Κρίμα, νόμιζα ότι θα με αφήνατε. Τέλος πάντων, προσπάθησα. Ε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Ε, κύριε Πίτροπε, ευχαριστούμε για την πρότασή σα για τη στατική ενέργεια, που είναι μια από τι μεγαλύτερε προκλήσει για την Ευρώπη. Το ζωτικό ζήτημα είναι ότι αν αρχίσουμε να μιλάμε για μεγάλε προκλήσει στον τομέα τη ενέργεια, θα πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε και για το ε, μακροπρόθεσμο όραμά μα από την Επιτροπή έχω ακούσει διάφορου επιτρόπου να μιλάνε για τέτοια θέματα, Όμω σα βεβαιωθούμε ότι εμεί ω Ευρώπη έχουμε συνέστηση του πού βρισκόμαστε σε σχέση με την ενέργεια και με ορίζοντα το 2050. Ένα από τα εμβληματικά μα σχέδια είναι η καλή χρήση των πόρων και ενεργειακή απόδοση. Αυτό ε, διέπει όλο μα το ενεργειακό πρόγραμμα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ σαφεί. Έχουμε ένα στόχο για τι κλιματικέ αλλαγέ. Αυτό θα πρέπει να μεταφραστεί σε εκπομπέ αερίων του θερμοκηπίου. Θα πρέπει να έχουμε μείωση 90% όλων των, αερίων, εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο 2050. Τι σημαίνει αυτό. Τεράστιε αλλαγέ για το ενεργειακό μα σύστημα. Πώ θα το πετύχουμε αυτό. Ο στόχο θα πρέπει να είναι το όραμα για το 2050 και πώ θα φτάσουμε εκεί. Βήμα 1 εξοικονόμηση ενέργειας, λιγότερη ενέργεια, λιγότερες εισαγωγέ, λιγότερη ενέργεια, λιγότερες ε, εναλλακτικέ και λιγότερο κόστο για του Ευρωπαίου πολίτε. Το νούμερο ένα λοιπόν θα πρέπει να είναι η εξοικονόμηση ενέργεια. Χωρί δεσμευτικού στόχου, καταλαβαίνω ότι η Επιτροπή ακόμη δεν το σκέφτεται. Να κάτι που θα έπρεπε να σκεφτούμε. Έπειτα για την εξοικονόμηση ενέργεια μακροπρόθεσμα. Βασική τομή για να το πετύχουμε αυτό είναι ο τομέα παραγωγή, ο τομέα των κτηρίων, τη στέγαση και των μεταφορών. Οι τομεί αυτοί είναι τομεί όπου θα πρέπει να γίνουν επενδύσει και να διασυνδεθούν αυτά με τον προπολογισμό σαφέστατα. Στέγαση και μεταφορέ. Εκεί θα πρέπει να γίνει πραγματική εξοικονόμηση, στις κεντρικές ευρωπαϊκές χώρες. Διασυνδέστε τα πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας με τις πολιτικές συνοχής. Να είμαστε σαφεί. Μιλάτε για mainstreaming και ευθυγράμμιση. Ξεκινήστε από αυτό για να έχουμε σαφή αποτελέσματα για τον προπολογισμό. Αυτό λοιπόν είναι ένα μέσο που μπορεί να γίνει εξοικονόμηση. Βήμα 2. Να αναπτυχθούν εναλλακτικέ λύσει. Πώ θα φτάσουμε στο μακροπρόθεσμο στόχο. Η βασική εναλλακτική είναι βεβαίω οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα στον τομέα τη παραγωγή ενέργεια. Εκεί πρέπει να πάμε κατευθείαν στι ανανεώσιμε πηγέ. Αυτή είναι η βιομηχανία του μέλλοντο. Όπω ήδη γίνεται στην Ισπανία, στη Δανία, στη Γερμανία για τον τομέα αυτό μπορούμε να θέσουμε στόχους για το 2050, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα. Ξέρω ότι υπάρχουν ομάδες και κόμματα που μιλούν για χαμηλές ε, εκπομπές άνθρακα, για λιγότερη χρήση του άνθρακα και σκέφτονται την πυρηνική ενέργεια ευσεβεί οι ε, φιλοδοξίες τους και υπόφητου, αλλά αν αρχίσουμε τώρα τη συζήτηση για την πυρηνική αντιπαραβαλόμενη με τι ανανεώσιμε, δεν θα καταλήξουμε εκεί που θέλουμε και θα καταλήξουμε στην περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα. Εάν θέλουμε λοιπόν να σκεφτούμε το μέλλον, ε, καταλήγουμε σε περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια, διότι και οι πυρηνικοί και οι ανανεώσιμε καταλήγουν σε αυτό. Εάν πρέπει λοιπόν να γίνουν επενδύσει κάπου τώρα, είναι στι υποδομέ παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια. Αν μιλάμε για υποδομέ, παρακαλούμε συγκεντρωθείτε στο ηλεκτρικό ρεύμα, στην ηλεκτρική ενέργεια όχι μόνο στα μεγάλα δίκτυα και στα μικρά και στα μικρότερα και στα ΕΦΗ. Εκεί πρέπει να γίνουν οι βασικέ επενδύσει. Εάν σκέφτεστε λοιπόν τι εναλλακτικέ σα λύσει, θα καταλάβετε ότι το βασικό ζήτημα είναι η ηλεκτρική ενέργεια. Και εναλλακτικέ λύσει χρειάζονται και για τον τομέα των μεταφορών. Διότι πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί και στι μεταφορέ. Εκεί είναι η μεγάλη δυσκολία. Έρευνα. Έρευνα είναι από τα βασικά ζητήματα που ε, τα βασικά στοιχεία που μα λείπουν. Όχι έρευνα βάσει των παλιών μα φιλοδοξιών όπω ΙΤΕΡ. Αυτό είναι μια ξεπερασμένη φιλοδοξία φιλοδοξία. Στον τομέα των μεταφορών πρέπει να έχουμε μεγάλε φιλοδοξίε. Και εκεί ε, πρέπει να έχουμε και οικονομικέ φιλοδοξίε. Εκεί βρίσκεται το μέλλον. Να μιλάμε για βιώσιμα βιοκάψιμα. Πρέπει να τα πετύχουμε όλα αυτά με ερευνητικά προγράμματα. Εκεί θα μπορέσουμε να πετύχουμε κέρδη για την οικονομία μα και θα βελτιώσουμε το μέλλον τη βιομηχανία και αυτό μπορούμε να το διασυνδέσουμε και με τη γεωργική μα ατζέντα. Εκεί θα πρέπει να γίνουν σωστοί συσχετισμοί και με τον προπολογισμό. Βήμα τρίτο να σκεφτούμε τη μεταβατική περίοδο. Μιλάμε για το 2050. Πώ θα πάμε ως εκεί. Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι η προμήθεια σε φυσικό αέριο. Μεγάλα προγράμματα όπω το Ναμπούκο. Κοιτάξτε τα δεδομένα που διαθέτουμε. Εάν επενδύσετε στην εξοικονόμηση που λέγαμε, η προμήθεια σε αέριο θα αυξηθεί λιγάκι ως το 2020 και μετά θα μειωθεί. Σαφώ. Θα ήμασταν λοιπόν ανόητοι αν επενδύαμε σε μεγάλα προγράμματα όπω το Ναμπούκο τώρα μόνον, γνωρίζοντα ότι μετά το 2020 οι εισαγωγέ του αερίου θα μειωνόντουσαν. Α σκεφτούμε και τα δεδομένα που διαθέτουμε τώρα όταν σκεφτόμαστε τη μεταβατική περίοδο. Το πιο σημαντικό είναι ότι ω Ευρώπη θα πρέπει να ενώσουμε τι εξωτερικού μα στόχου ω προ την ενέργεια. Λοιπόν, ε, συνοψίζω σύντομα. Στόχοι για το 2050, ε, μετάφραση σε βήματα τώρα. Ε, έρευνα, βιοκαύσιμα, μεταβατική περίοδο εναλλακτικέ λύσει, αλλά μην σκέφτεστε μόνο τα μεγάλα προγράμματα. Πρέπει να είμαστε έξυπνοι όταν σκεφτόμαστε. Wunderbar. Θαυμάσια. Νομίζω ότι σχεδόν τέλεια τα καταφέρατε. Και τώρα ε, για τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς ο Κόντρα Τσιμάνσκι. Κύριε Επίτροπε, δεν είναι πρώτη φορά που μας παρουσιάσατε ένα πολύ πλήρες πρόγραμμα για ε, δαπάνες και αυτό είναι τεκμηριωμένο διότι έχουμε πολύ ε, φιλόδοξους στόχους όσον αφορά την, το πρόβλημα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων την αποτελεσματικότητα του ηλεκτρικού την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς μας που όλα αυτά πρέπει να καταλήξουν σε χαμηλότερο κόστος, χαμηλότερες τιμές. Όσον αφορά τα προγράμματα. Έχουμε το Ναμπούκο και όχι μόνο θέλουμε να συνδέσουμε τον Βορρά με τον Νότο και όλα αυτά σημαίνουν ότι θα χρειαστούν πάρα πολλά χρήματα που αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν υφίστανται στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Επίσης μιλάμε εδώ για δημόσιο ε, χρήμα και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σοφά. Ως εκ τούτου θα πρέπει να ε, κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου όσον αφορά τις δαπάνες. Ο μόνος λόγος για τον οποίο θέλουμε να διοχετεύσουμε τέτοιες πιστώσεις ε, στην ε, ε, ενέργεια είναι για να επιτύχουμε ενεργειακή ασφάλεια και θα πρέπει να αυξήσουμε την ενεργειακή μας ασφάλεια γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να προκόψει και η οικονομία. Εάν όμως μιλάμε για ενεργειακή και ε, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια θα πρέπει να ασχοληθούμε με λεπτομέρειες, δηλαδή τη διαφοροποίηση. Η διαφοροποίηση η οποία θα πρέπει να προχωρήσει εις βάθος και να μην ασχοληθεί μόνο με ε, τις συνδέσεις αλλά να προχωρήσει και περαιτέρω. Περισσότερες πηγές. Όχι μόνο περισσότερες ε, προελεύσεις πηγές. Θα πρέπει λοιπόν να καταρτήσουμε διάφορα κριτήρια για να διαχειριστούμε τους περιορισμένους πόρους που διαθέτουμε. Είναι κριτήρια τα οποία θα βασίζονται σε αυτή την βαθύτερη διαφοροποίηση, περισσότερες ε, πηγές και όχι μόνο αυτό. Και αυτό με οδηγεί εις ε, την τελευταία μου ερώτηση. Ή στο πρόγραμμα υποδομών ε, θα υπάρξουν και άλλα κριτήρια κόστους πράγμα το οποίο πρέπει να ε, εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν μόνο ευρωπαϊκές αξίες και δεν θα υπάρχει μόνο διαφοροποίηση των πηγών μας αλλά και κάτι πιο χρήσιμο. Τώρα ο Μίγκελ Πόρτας. Ε, τα πέντε λεπτά του πράσινου συναδέλφου έκαναν περιττές όλες τις υπόλοιπες παρατηρήσεις, λίγο πολύ. Εγώ θα ήθελα δύο βασικά σχόλια να κάνω. Ή σχόλια, αν θέλετε. Πρώτα απ' όλα από αυτά που άκουσα υπάρχει μια σαφής αντίφαση μεταξύ των αριθμών και των, της έκφρασης των στόχων μας, ενώ είχαμε αρχικά στόχους πολύ σαφείς, μέσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους και κυρίως δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα μέσα χρηματοδότησης. Ως προς τα μέσα χρηματοδότησης λοιπόν και επειδή βρισκόμαστε ενώπιον μιας επιτροπής που Ω επιτοπλίστων συζητά τα θέματα αυτά, προπολογισμό, χρηματοδότησης, Δεν καταλαβαίνουμε πώς προτίθεστε να επιλύσετε αυτό το, αυτή την πτυχή του προβλήματος και με, μένα ε, μια επιβαρυντικό παράγοντα. Η στρατηγική χρηματοδότηση θα βασιστεί σε ε, εταιρικέ σχέσει δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Αυτέ οι σχέσει είναι το χειρότερο μέσο από την άποψη του δημόσιου χρέου. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να είμαστε πάρα πολύ σαφεί. Ποια είναι η άποψή σα, αυτό θέλω να ρωτήσω ξεκάθαρα. Ποια είναι η άποψή σα για τι εταιρικέ σχέσει δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Δεν είναι δυνατόν να ακούμε λόγους για την απόλυτη ανάγκη να μειωθούν τα χρέη και ταυτόχρονα να συνεχίζουμε να μιλάμε για εταιρικέ σχέσεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Δεύτερη παρατήρηση. Τα προβλήματα της ενεργειακής αποδοτικότητας. Δεν είναι δύσκολο κάποιοι στόχοι να επιτευθούν ως το 2020. Όμως, ως προς την απόδοση αυτή καθεαυτή, ξέρουμε ότι ποτέ δεν θα την πετύχουμε πλήρως. Και γιατί θα συμβεί αυτό. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι η απόδοση αντιθέτως από άλλους στόχους δεν είναι ευρωπαϊκός στόχος. Είναι ένας στόχος που εξαρτάται από τα κράτη, τα εθνικά κράτη επί της ουσίας. Θα ρωτήσω λοιπόν το εξή. Για πόσο καιρό ακόμη θα συνεχίζουμε να μην έχουμε πλέον τη δυνατότητα να ορίσουμε επιτακτικού στόχου στον τομέα αυτό τη ενεργειακή απόδοση. Έω πότε, κύριε Επίτροπε, θα αφήνουμε στα κράτη τη δυνατότητα να εκπληρώσουν όσο καλύτερα μπορούν έναν στόχο αύξηση της απόδοσης έως το 2020. Η ερώτηση αυτή είναι ζωτική σημασίας διότι έχει να κάνει με το πώς προσεγγίζουμε το πρόβλημα της απόδοσης της πόλης. Έχουμε ένα σύνολο μέσων τα οποία είναι διάσπαρτα, όπου τα κράτη και οι δημοτικές αρχές μπορούν να προσφύγουν, να ανατρέξουν, για να αυξήσουν την απόδοση, να ανακαινήσουν, να αναπαλαιώσουν και ούτω καθεξής. Τα μέσα αυτά όμως δεν συγκεντρώνονται σε ένα κεντρικό, σταθερό και σε γερά θεμέλια πρόγραμμα ευρωπαϊκό ώστε να υπάρχει η αυτή η αναδιάρθρωση των πόλεων. Εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε δυνατότητες απασχόλησης και για απασχόληση για εργαζομένους με προσόντα, όχι μόνο για εργάτες και με επιχειρηματική δράση, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη. Πείτε μου λοιπόν, πώς θέλετε να αυξηθεί η απόδοση μακροπρόθεσμα και ενώ υποστηρίζουμε ότι θέλουμε να ανανεώσουμε τις πόλεις μας και αυτό μόνο με ένα φεντέρ ε, ως ε, μέσο χρηματοδότησης δεν είναι λογικό, δεν βγάζει νόημα. Πείτε μας λοιπόν, σε αυτόν τον τομέα σκοπεύετε να θέσετε υψηλότερες φιλοδοξίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τελευταίος ομιλητής για την ΕΦΤΕ, η κυρία Τσαβέλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω δύο σχόλια. Το πρώτο είναι ότι είμαι βέβαιος ότι η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας έχει εκτιμήσει και συμπηλήσει τα δεδομένα που διαθέτει, οπότε καταλαβαίνουν πόσα κονδύλια διαθέτουν για τις ενεργειακές επενδύσεις και καταλαβαίνουν τι διαφορά υπάρχει, τι κενό, ώστε να εξευρεθούν τα κονδύλια και να, εκπληρωθεί να καλυφθεί αυτό το κενό. Από όσα άκουσα, η κάλυψη των κενών θα γίνει από κονδύλια εκτός του προπολογισμού τα οποία απαιτούνται για να αναπτυχθούν αυτέ οι τεράστιε υποδομέ, μεγάλε επενδύσει. Από πού θα έρθουν όμω αυτά τα κονδύλια, φαντάζομαι από τη συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ή από τον ιδιωτικό απλώ. Όμω, βάσει των όσων ακούσαμε από τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη ίδια, τον κύριο Μπαρόζο, εκείνο μα είπε ότι τα ευρωπαϊκά, το πρόγραμμα για τα ευρωπαϊκά ομολογά ίσως είναι ένα μέσο για να εξεύρουμε κονδύλια και να χρηματοδοτήσουμε τεράστια ευρωπαϊκά προγράμματα. Η ενέργεια είναι ένας τομέας όπου ακριβώς το ευρωπαϊκό πρόγραμμα των ε, ομολόγων, των bonds, θα είναι καθοριστική σημασία. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον Επίτροπο, πώς σκοπεύετε τα εταιρικά μόλογα να συνδυαστούν με τα ευρωπαϊκά ώστε να μπορέσουμε τελικά να αποσπάσουμε επενδύσεις για την ενέργεια. Η δική μου ερώτηση είναι κατευθύνεστε προς τα εκεί και σε ποιο στάδιο της διαδικασίας βρίσκεστε. Διότι πραγματικά νομίζω ότι εκεί το θέμα είναι ακριβώς πώς θα γίνει το μοίρασμα με αυτό το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα μόλογων. Μάλιστα, αυτά αναφέρονται και στην ε, δημοσιονομική ανακεφαλαίωση, την, την παρουσίαση την πρόσφατη της Επιτροπής για τον Προπολογισμό. Συμπεραίνουμε από όσα ακούσαμε ότι οι επενδύσεις στην ενέργεια είναι ιδιαίτερα δαπανηρές, διότι η Ευρώπη δεν έχει δικούς της πόρους ενεργειακούς, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα ή μέσο πρόθεσμα. Είδαμε τι συνέβη με τις πρόσφατες κρίσεις ε, σε γειτονικές χώρες και στην Αίγυπτο. Εάν υπάρξει λοιπόν ε, μια τέτοια λυσίδα γεγονότων, ιδίως στη Βόρεια Αφρική, θα συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι ο Νότιος Διάδρομος και η Κεντρική Ευρώπη θα αντιμετωπίσουν τεράστια προβλήματα. Τι κάνουμε λοιπόν. Πρέπει να δούμε εάν μπορούμε να καλυφθούμε από τους δικούς μας πόρους, τους ενεργειακούς. Το ερώτημα μου λοιπόν προς τον Επίτροπο είναι, χρηματοδοτούμε ή δίνουμε στο κίνητρα στις ιδιωτικές εταιρείε να κάνουν έρευνα, να εξορίξουν όπου χρειάζεται, να αποσπάσουν λύσεις. Μπορούμε να βρούμε νέους πόρους ενέργειας. Πολύ πρόσφατα άκουσα για κοιτάσματα φυσικού αερίου μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ. Υπολογίζεται ότι υπάρχει ένα τρεις κυβικών μέτρων τρία-τρει μέλλον κυβικών μέτρων στο κοίτασμα αυτό. Ε, το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξή. Θα δώσετε κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα, στι ιδιωτικέ εταιρείε, επίτροπε, ώστε τελικά με τις δικές μας ενεργειακέ πηγές να καλυπτώμεθα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αυτός ήταν ο γύρος των πολιτικών ομάδων. Ε, τώρα όμω υπάρχει ένας ε, μακρύς ε, κατάλογος ομιλητών που περιλαμβάνονται ιδίω φιλελεύθεροι συνενάδελφοι. Αλλά εγώ θα πάρω τρεις ομιλητές κατά ένα λεπτό, ε, Ήβας Βόλγουσλαβ Σλαβδικο-Λιμπεράτσχη και Γιάν Ούλριχτ. Κάθε φορά για ένα λεπτό και μετά ο Επίτροπος θα ε, πρέπει να κάνει τις απαντήσεις τους και μετά θα προχωρήσουμε στον κατάλογο των ομιλητών αν έχουμε ακόμη χρόνο. Διότι διαφορετικά εφόσον είναι, θα είναι ήδη 10 και 4 θα διαγράψουμε απλώς τους ε, συναδέλφους από τον κατάλογο των ομιλητών. Ράιμερ. Ε, φαντάζομαι δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αλλά θα ήθελα ε, αν υπάρχουν συνάδελφοι που είναι στον κατάλογο που ε, έχουν ερωτήσεις θα ήθελα η γραμματεία τουλάχιστον να μπορέσει να τις τα δώσει γραπτός ή στον Επίτροπο. Βέβαια είπε ο Επίτροπος ότι για όσους δεν μπορέσει να απαντήσει θα απαντήσει γραπτός οπότε αυτό δεν είναι πρόβλημα. Συνεχίζουμε λοιπόν ένα λεπτό ο Ήβαν. Ευχαριστώ. Έχω δύο ερωτήσεις κύριε Υπουργέ. Καταρχήν, αν κοιτάξετε τον προϋπολογισμό του 2011 δεν έχετε πολλά χρήματα. Είναι το 1 πέμπτον λιγότερο από το 2010 ε, και υπάρχουν χρήματα τα οποία αφαιρέθηκαν από τα διαρθρωτικά ταμεία και από τη γεωργία. Οπότε ε, τι σύστημα υπάρχει για να παρακολουθήσουμε την πορεία αυτών των πόρων διότι θα δοθούν τα χρήματα και ποιο θα είναι λοιπόν το σύστημα με το οποίο θα παρακολουθήσουμε τα προγράμματα αυτά, διότι μετά θα μας ρωτήσουν ποιο είναι η αποτελεσματικότητα αυτού του διαβήματος. Και το δεύτερο ερώτημα είναι πολύ συγκεκριμένο. Ένα από τα παραδείγματα ε, του δικτύου είναι Σουηδία-Λιθουανία και αντιλαμβάνουμε τώρα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προχωρήσει. Είναι ρεαλιστικό να προχωρήσει αυτό το εγχείρημα ή όχι. Και ο επόμενος είναι ο Μπόγκουσλαφ Λιμπεράτσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα πολύ σύντομο ερώτημα έχω για τον ε, Επίτροπο. Η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών. Θα μπορούσατε να μας πείτε δύο πράγματα παραπάνω γι' αυτό. Για το αέριο για άλλες πηγές επίσης ε, διαφοροποίηση με βάση την ε, γεωγραφική πτυχή και ακόμη και αν ε, αυτές οι πηγές βρεθούν θα μπορέσουν να μας ικανοποιήσουν στο μέλλον ο Γιάν Ουλριχτ ευχαριστώ ε, κύριε Επίτροπε δύο ερωτήματα το ένα έχει να κάνει με την αξιολόγηση των αρχών που διέπουν την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Μιλήσατε για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Πώς ακριβώς ε, αξιολογείτε την κατάσταση τώρα. Έχει λειτουργήσει το σύστημα τελικά ή όχι. Και δεύτερον, ξέρω ότι κάποια από τις ε, γενικές διευθύνσεις έχει υποστηρίξει την ιδέα μιας ε, σύμβασης για την ενέργεια κάτι που συζητείτε γενικώ. Εσεί έχετε σκεφτεί καθόλου κάποια ε, οικονομική, κάποιο οικονομικό κίνητρο για όσου θέλουν όντω να μειώσουν την ε, κατανάλωση διοξιδίου του άνθρακα. Ευχαριστώ. Ε, να δώσουμε το λόγο τώρα στον Επίτροπο για να απαντήσει. για το, το καθήκον μου τώρα είναι να κάνω προτάσεις για τον τομέα της ενέργειας για προγράμματα, για project, για ε, στόχους που θα θέσουμε στην επόμενη δημοσιονομική περίοδο για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τον εξευρωπαϊσμό. Αυτό θα είναι ένας μεγάλος κατάλογος από αυτό που θα μπορούσε να καλύψει ο ήδη υπάρχον προπολογισμό, αλλά τώρα θα ήταν λάθος να σας πω από την αρχή, να μην πω μάλλον σε πολύ φιλόδοξα προγράμματα που υπάρχουν. γιατί έχουμε ξεπεράσει με πηγές από άλλους τομείς όπως ας πούμε θέματα υποδομών, γεωργία κτλ. γιατί τότε τα κράτη-μέλη και εσείς θα αναρωτιέστε Πώ ακριβώ θα εξελιχθεί στο σύνολό του ο προπολογισμό. Όλοι έχουμε διάφορες εμπειρίες από τις τελευταίες ε, ε, εβδομάδες με απεργίες στα, στα κράτη-μέλη κλπ. Πρό το παρόν, εγώ είμαι πεπισμένο ότι θα μπορέσουμε να έχουμε εξευρωπαϊσμό της ενεργειακής πολιτικής και ολοκλήρωση της ενεργειακής πολιτικής ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιπλέον προστιθέμενη αξία, απόδοση για να μπορέσουμε να ε, επιτύχουμε τους στόχους μας. Απόδοση. Ένας ευρωβουλευτής είπε ότι η απόδοση προς το παρόν δεν έχει επιτευχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά στα κράτη-μέλη και στα κρατήδια. Αυτό ισχύει και για τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Ισχύει για τους περισσότερους στόχους. Μιλούμε όμως για προγράμματα κυρίως περιφερειακά, για προγράμματα τοπικά. Για το θέμα των ε, κτηρίων και της εξυγίανσής τους, είναι όντως αυτό ένα σημαντικό στόχος που έχουμε θέσει. Και η δική μου πεποίθηση είναι ότι η ε, σύγκληση του ε, προϋπολογισμού στα περισσότερα κράτη-μέλη νομίζω ότι θα λειτουργήσει έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε μειώσεις για τα δημόσια οικονομικά, για την εξυγίανση των ιδιωτικών και των δημοσίων κτηρίων. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε κίνητρα με τα διαρθωτικά προγράμματα, τότε και τα κρατημέλη και οι περιφέρειες και οι κοινότητες θα θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν. Και το θέμα είναι να μην μειωθούν τα κονδύλια που δίδονται, αλλά να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο και πρέπει να υπάρχει και ένα σκόπιμο κίνητρο. αυτό, αυτό προσπαθεί να κάνει ο προπολογισμό. Υπάρχουν τα συγκεκριμένα, οι συγκεκριμένοι στόχοι που έχουν τεθεί και σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο και θεωρούμε ότι μπορούν να, να επιτευχθούν. Ένα, το κόστος για την εξηγήνση ενός ενός κτηρίου θα φανεί, το κόστος θα φανεί τώρα αλλά το όφελος θα φανεί σε 10 χρόνια. Οπότε ας επενδύσουμε τώρα για να μπορέσουμε να έχουν τα παιδιά μας να υποφεληθούν από, από την εξυγίανση αυτή. Αυτό θα είναι η πρώτη περίπτωση μιας, ε, ε, της, ε, του ότι θα κάνουμε εμείς κάτι για να το βρει τελικά προστάτες η επόμενη γενιά. Αυτό μπορεί να ξεκινήσει από την εξυγένση των κτηρίων, για να μπορέσουν τα παιδιά μας να επωφεληθούν από καλύτερα ε, κτίρια και να ε, βοηθήσουμε και εμείς βεβαίως και στην εξοικονόμηση κονδύλιων αλλά και στην ε, αντιμετώπιση των κλιματικών προβλημάτων. Για το θέμα της έρευνας τώρα. δεν ε, θέλω να πιστεύω ότι είναι ανόητα αυτά που, αυτά που λέμε. Το ITER είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είχε και μεγάλη πλειοψηφία όταν υπευλήθη. Νομίζω ότι τώρα δεν μπορεί το Κοινοβούλιο να λέει ότι αυτή η πλειοψηφία ήταν ανόητη, ήταν χαζή. Ε, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό που λέτε. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να, κάνουμε, να λέμε κάτι τέτοιο, γιατί έχουμε ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Και το Ιντερ, το Ιντερ νομίζω ότι πρέπει μέχρι το τέλος να το φτάσουμε. Για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ε, πρότυπο για την ενεργειακή παραγωγή. Οι δημοκράτες πρέπει να δέχεστε τις πλειοψηφίες. Εγώ δέχομαι την πλειοψηφία που προκύπτει στο κοινοβούλιο. Τώρα, στο μέλλον, αν ακυρώσουμε το ΙΤΕΡ, δεν θα μας παίρνουν σοβαρά ούτε οι Κινέζοι, ούτε οι Ρώσοι, ούτε οι Αμερικανοί. Γιατί δεν θα είμαστε αξιόπιστοι σε κανένα επίπεδο πια. Είναι θέμα αξιοπιστίας το να ολοκληρώσουμε το ίτερ. Ξεπερνάει δηλαδή το θέμα της ε, πυρηνικής σύνταξης. Το θέμα δεν είναι να έχουμε ίτερ ή γενική έρευνα. Αυτό θα ήταν ελαφασμένο πρέπει να έχουμε τον διάδρομο για το ίτερ και μετά πρέπει να έχουμε έναν άλλο ε, διάδρομο ε, για υπόλοιπα, ανεξάρτητο από το ίτερ, για τα υπόλοιπα ε, project σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα για τις υποδομές. Νομίζω ότι τα δάνεια είναι σκόπιμα. Η έρευνα πρέπει να, έχει, πρέπει να είναι αντικείμενο, πρέπει να έχει συγκεκριμένους τομείς ε, συγκεκριμένου στόχου, συγγνώμη. Αλλά όταν μιλάμε για υποδομές, για διασυνδέσεις, για, αποθήκευση, για αποθήκευση και αν θέλουμε να επενδύσουμε σε όλα αυτά, τότε μιλούμε για ε, σύγκληση όλων αυτών των τομέων στον τομέα των υποδομών. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσω δανείων και ιδιωτών επενδυτών. Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει. Και πρέπει να πω και αυτό. Θα είναι και πιο φθηνό. Συν, ε, Τι ζητούν οι ε, τράπεζες τι ζητούν οι, ε, τα ταμεία, τι ζητούν οι, τα ιδιωτικοί το, φορείς. Και ο τόκος για το δάνειο αυτό θα είναι πιο μικρός από το, το επιτόκιο, συγγνώμη, θα είναι πιο μικρό, από το επιτόκιο που πληρώνουν τα κράτη-μέλη μας τώρα. Θέτω λοιπόν το ερώτημα, γιατί θα τεθεί. Έχουμε υποδομές για ε, μεταφορές, για ICT e και ενέργεια και για κτίρια. Νομίζω λοιπόν ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι στο τέλος ο λογαριασμό δεν θα είναι πιο μικρό. Νομίζω ότι αξίζει πάση περιπτώσει να το σκεφτούμε. Και στην ε, Κομισιόν αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή, το συζητούμε, το μελετούμε και θα δούμε τι θα προταθεί και από τα κράτη-μέλη. Για τι υποδομές προφανώς θα έχουμε και έναν κατάλογο προτεραιοτήτων. Και αυτόν προσπαθούμε να επεξεργαστούμε τα, τα, επιπλέον, ε, ε, τα επιπλέον κονδύλια δεν είναι από τώρα μέχρι το 2020. Μιλούμε για τον τομέα γενικώ ε, τι διάφορε συνιστώσει τη ενέργεια και την αποθήκευση και την απόδοση. Μπορεί να μιλούμε για πολύ μεγάλα ποσά. Και το, το μισό μπορεί να είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και το άλλο μισό κονδύλι που θα χρειαστεί να είναι αντικείμενο συγχρηματοδότησης με συγκεκριμένα κίνητρα. Γι' αυτό η δική μου πρόταση ήταν το μέσο πρόγραμμα που έχουμε στην, ε, στο οικονομικό μας πρόγραμμα να, μπορεί να είναι και εφαρμόσιμο. Έχουμε 2,4 δισεκατομμύρια για τις ε, υποδομές. 98% έχει εφαρμοστεί και έχει, έχει χρησιμοποιηθεί και έχει πάει και καλά. Αυτά τα 2,4 ε, ε, ε, δισεκατομμύρια μοιράστηκαν σε τρία χρόνια. Μιλούμε δηλαδή για πολύ μεγάλα ποσά, τα οποία βεβαίως είναι και, αποτελούν και ένα σημαντικό κίνητρο για τη συγχρηματοδότηση. Δηλαδή δεν έχουμε προγράμματα για να δημιουργήσουμε υπερβολικές δαπάνες. Μέχρι το 2015 θέλουμε να ε, έχουμε μονώσεις και στα νησιά διότι δεν είναι ε, δυνατόν να ε, δεν, μπορεί να υπάρχει απομόνωση μάλλον νησίδες απομόνωση στην Ευρώπη. Θα πρέπει να μην εξαρτώμαστε από τρίτα κράτη κανείς μέσα στην Ευρώπη και θα πρέπει να υπάρχουν δίκτυα διασύνδεση σε όλη την επικράτεια διότι πέρυσι πήραμε ορισμένες αποφάσεις. Κάθε χώρα θα πρέπει να αυξήσει τα αποθέματα του σε 30 ημέρες επάρκεια αερίου. Δεν είναι ιδεώδες αλλά ποτέ δεν θα έχουμε επάρκεια αερίου σε όλα τα κράτη-μέλη. Ε, θα πρέπει επίσης επιχειρήσεις να μπορούν να μεταφερθούν. Αν έχουμε σε κάθε όμως κράτος 30 ημερών επάρκεια αερίου μπορεί να υπάρχει αλληλοβοήθεια, αλληλεγγύη σε περίπτωση ανάγκης. Και αυτό θα πρέπει να γίνει και στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, στα δίκτυα διασυνδέσεως για την, ε, για την επάρκεια όλης της Ευρώπης και ε, θα πρέπει εκεί να εξετάσουμε το, ε, ε, τις, ε, τις προϋποθέσεις δανεισμού. Διότι όσον αφορά τα προγράμματα μας ε, θα, υποβάλουμε το δεύτερο τρίμηνο ένα ερωτηματολόγιο με εναλλακτικές λύσεις κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αποθήκευση ε, ηλεκτρικού και θα δούμε, ε, θα ρωτήσουμε μάλλον πώς μπορούμε να αποθηκεύσουμε το ηλεκτρικό ρεύμα διότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε το αέριο, το πετρέλαιο, τα, την πυρηνική ενέργεια, μπορούμε να παγώσουμε το ψωμί, αλλά δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε το ηλεκτρικό ρεύμα εκτός από το νερό. Πρέπει να δούμε εάν υπάρχουν δυνατότητες με την Ορβηγία, ένα εταιρικό κράτος ή στις Άλπεις με την Ελβετία ή στα Δυτικά Βαλκάνια να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αποταμιευτήρες ρεύματος δηλαδή σε συνεργασία με το πρόγραμμα Natura 2000. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Στην Αυστρία παραδείγματος χάρη η στην Αυστρία ε, μπορούν να ετοιμάσουν ε, αποταμιευτήρες ε, στο Καπρούν αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα δίκτυο στη υπόγειο και εκεί χρειάζεται μία διαδικασία αδειοδοτήσεως. Υπάρχουν άλλες δυνατότητες από την αποθήκευση άλλων προϊόντων όπως είναι το υδρογόνο ή η μπύρα παραδείγματο χάρη. Χρειάζονται άλλε δυνατότητε. Γι' αυτό ε, μίλησα για μεταφορέ όπου δεν επιτύχαμε πολλά με τα, ε, τις πηγές ενεργείας ε, από βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς. Αυτό ήταν κάτι που είχε εξεταστεί πριν από μερικά χρόνια αλλά δεν επιτύχαμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενεργείας θα πρέπει να γίνουν κάτι. Και ρωτώ τώρα, μπορείτε να φανταστείτε η Γαλλία, ένα κράτος το οποίο συμπαθώ πολύ, ε, πιστεύετε ότι θα είναι έτοιμη σε 40 χρόνια να χρησιμοποιεί μόνο ε, ανανεώσιμες ενεργείες με μηδέν διοξίδιο του άνθρακος ή η Πολωνία ότι δεν θα έχει διοξίδιο του άνθρακος και θα χρησιμοποιεί μόνο ανανεμώσεις με πηγές ενεργείας. Πρέπει να έχουμε λύσεις οι οποίες να είναι εφικτές για όλα τα κράτη-μέλη και γι' αυτό το είναι η δυνατότητα να έχουμε περισσότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος, να έχουμε ε, ένα μείγμα πετρελαίου με διοξίδιο του άνθρακος και ένα ε, ποσοστό αερίου με εκπομπές που θα συνδυαστούν. Είναι όμως ένα σχέδιο το οποίο επεξεργαζόμαστε και σε λίγους μήνες θα υποβάλουμε στο Κοινοβούλιο προς εξέταση από τους Ευρωβουλευτές. Ε, βεβαίως ε, είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω στις ε, επόμενες υπόλοιπες ερωτήσεις. Συζητάμε τα διάφορα θέματα και βρισκόμαστε εδώ στην αρχή μία συζητήσεως με τους συζητητέ. Εγώ λοιπόν στους επόμενους μήνες θα επανέλθω με τα θέματα αυτά και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Έτιγεν. Όντως σας ευχαριστούμε για όλες τις απαντήσεις που μας δώσατε και για την δυνατότητα ε, να απαντήσετε γραπτός όσα θέματα μείναν ακόμη σε κρεμότητα και προτού ξαναδώσω τον λόγο στο Σαλβαντόρ για να κλείσει το θέμα θα ήθελα να σας πω ότι όταν κοιτώ την, ε, τον κατάλογο μιλητών και παρακαλώ τους συναδέλφους να διατυπώσουν τις ερωτήσεις τους γραπτός γραπτός να τις δώσουν στη γραμματεία κατά τρόπον ώστε ε, να δοθούν εις τον εισηγητή ε, η Πιλάρ Καστίγιο και άλλοι τρεις οι οποίοι παρακαλούνται να συντάξουν γραπτός στην ερώτησή τους και να τη έχει το λόγο. Hm.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 σχόλια για όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν και διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα το Κοινοβούλιο σύντομα θα πρέπει να υποβάλει μια πρόταση ε, με συγκεκριμένα μέτρα. Θα πρέπει λοιπόν να τοποθετηθούν οι πολιτικέ ομάδε σε σχέση με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άκουσα με προσοχή αυτό που είπε ο Επίτροπο, ότι θα πρέπει να περιορίσουμε τον αριθμό προτεραιοτήτων αλλά θα πρέπει να είμαστε βέβαια για την επιλογή τους. Να είναι οι σωστές. Σιγά σιγά οι παλιές προτεραιότητες θα αντικατασταθούν από νέες. Αυτό είναι κάτι που μας βρίσκει όλους σύμφωνους ε, και ως προς το χρονοδιάγραμμα. Όλοι θέλουμε ενέργεια πιο ανταγωνιστική και πιο καθαρή, πιο πράσινη θα μπορούσε η ενεργειακή πολιτική να γίνει ένα μέσο για την ανάπτυξη της Ευρώπης και βεβαίως εδώ απαιτούνται σημαντικότατες επενδύσεις. Ιδιαίτερο στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για το 2020. αλλά και για την μεσοπρόθεσμη στρατηγική μας με τους τρεις στόχους μας γύρω από τα ποσοστά του 20%. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ενδιασμοί από κάποια κράτη-μέλη, διότι σαφώς υπάρχουν δημοσιονομικοί περιορισμοί και τα ποσά που προβλέπονται θα είναι ένα μεγάλο βάρος για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Πάντως, πάντοτε παραμένει μία διαφορά μεταξύ των φιλόδοξων στόχων που θέτουμε και των μέσων με τα οποία αποφασίζουμε να τους πρικοδοτήσουμε. Η κατάσταση του προπολογισμού στα κάτι μέλη είναι δυσχερής. Το γνωρίζει αυτό και ο Επίτροπος. Και ξέρουμε ότι κάποιοι ως σχηνοβάτες προσπαθούν να ξέρουν το σημείο ισορροπίας μεταξύ των αναγκών για δαπάνες και των δημοσιονομικών περιορισμών. Μελλοντικέ δημοσιονομικές προοπτικές θα πρέπει εδώ να αποτελέσουν αντικείμενο εντατικότατης μελέτης για όλους μας. Θα πρέπει να είμαστε πολύ δραστήριοι και βεβαίως βλέπουμε ότι επενδύσεις απαιτούνται στον ενεργειακό τομέα με δεσμεύσει κρατικές και δημόσιες στο, στο συγκεκριμένο τομέα. Και βεβαίως και, και η παρουσία της κοινότητας της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Οι επενδύσεις λοιπόν στην ενέργεια εξαρτώνται από τα κράτη-μέλη και από την διακυβερνητική συνεργασία. τα πράγματα δεν θα είναι απλά. Εάν θέλουμε ο κοινοτικό προπολογισμό να διδραματίσει έναν σαφή ρόλο, θα πρέπει να λυθούν και αποφάσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μένα αυτό είναι αποφασιστική σημασία. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσει όλη τη την επιρροή στον τομέα των επενδύσεων, τη ενέργεια. Το συζητούμε αυτό ε, στην Επιτροπή μα. Μιλάμε για τον αντίκτυπο των μελλοντικών δημοσιονομικών προοπτικών και δικαίω, πολύ σωστά, μα μιλούν οι συνάδελφοι για εξοικονόμηση ενέργεια. Η εξοικονόμηση ενέργεια είναι σε κάθε περίπτωση η καλύτερη πηγή ώστε να εξεύρουμε πόρους, να αντλήσουμε πόρους. Δεν χρειάζεται σε αυτή την περίπτωση καν να αποδεσμευτούν κονδύλια. Και μετά ως προς τις υποχρεώσεις μας. Νομίζω ότι ε, πολύ γίνεται λόγος για τις δαπάνες και τις υποχρεώσεις που βαρύνουν τον προπολογισμό για τον τομέα των μεταφορών. Θα πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην θεωρούμε τίποτε δεδομένο ως τον προπολογισμό εφόσον δεν ξέρουμε ακόμη τι μελλοντικέ δυνατότητε χρηματοδότηση θα έχουμε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα συγκεκριμένα. Θα πρέπει η δική μας η Επιτροπή να εξετάσει το θέμα αυτό. Να δει κατά πόσον οι υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων μπορεί να εξαρκούν ώστε να επιτευθούν όλοι αυτοί οι στόχοι που έχουμε θέσει. Και υπάρχει κι άλλο ένα στοιχείο Μιλάμε για το συσχετισμό μεταξύ πολιτικής συνοχής και διαρθωτικών πολιτικών, αλλά και ενεργειακής πολιτικής. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα ήδη θεωρητικό στην αντίληψή μας την ενοιολογική. Ο Επίτροπος προσπάθησε να μας ε, δώσει κάποιες Απαντήσει και είδαμε ότι οι ενεργειακέ αποφάσεις μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην περιφερειακή πολιτική. Τα κράτη-μέλη παίρνουν πολλά κονδύλια από τα θεραπευτικά ταμεία, από τα ταμεία συνοχής. Τα κράτη αυτά μέλη θα είναι τα ίδια που θα καλούνται να πραγματοποιήσουν όμως μαζικές επενδύσεις για την διασύνδεση λόγω χάρη των δικτύων. Αυτό είναι μια διάσταση την οποία θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Θέλουμε να διαφυλάξουμε την περιφερειακή μας πολιτική, την πολιτική συνοχής επίσης, αλλά σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποιος είναι ο ρόλος της ε, διαδοτικής πολιτικής στο μέλλον των υποδομών, στη διασύνδεση των δικτύων στον τομέα της ενεργείας. Τα διευθυντικά ταμεία και πολιτική συνοχής δεν μπορεί παρά να αποτελούν μια πηγή χρηματοδότησης για τα έργα αυτά, αλλά με την συγκατάθεση των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Τα διευθυντικά ταμεία Μπορούν να είναι λοιπόν μια πηγή χρηματοδότησης ε, για τα έργα αυτά που φέρουν τις υποδομές αλλά θα πρέπει να το συζητήσουμε και ελπίζουμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία να το ξανασυζητήσουμε με τον Επίτροπο Έτιγκερ. Και σε ό,τι αφορά το ΙΤΕΡ, νομίζω συμφωνεί η Επιτροπή μας ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε εδώ τη χρηματοδότηση. Όμως, να σκεφτόμαστε και το εξή. Χρηματοδοτούμε το ΙΤΕΡ με τα πλεονάσματα τα οποία αποσπάσαμε από τον προπολογισμό της Γεωργίας. Δεν θα διαμορφώσουμε έτσι μια χρηστή, μια υγιή πολιτική προπολογισμού και ενεργειακή για το μέλλον. Πρέπει να προσέξουμε. Ευχαριστώ, Σαλβαδόρ. Όντω, σε πολλά σημεία πρέπει να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά πώ όλα αυτά που μα είπε ο Επίτροπο Ότιγκερ και που είναι όντω πολύ καλέ ιδέε, πώ λοιπόν θα μπορέσουμε να τι εφαρμόσουμε ε, και να είμαστε και ε, Προσεκτική ως προς τον προϋπολογισμό. Νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται πολύ περισσότερη ε, πειθό η ιστορία αυτή και από εμά και από τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε λίγο ξεπεράσει το χρόνο, αλλά εντάξει. Να καλωσορίσουμε τον David Sullivan ο οποίος είναι γενικός γραμματέας της, ε, της Επιτροπής Εξωτερικών ε, της Υπηρεσίας συγγνώμη, Εξωτερικών Υποθέσεων είναι έτσι διοικητικός ε, διευθυντής έχει γενική γραμματή συνήθως αυτό είναι αν δείτε και τις αρμοδιότητες τους Το ίδιο συμβαίνει και στην ΟΚΕ και στην Επιτροπή των Περιφερειών. Υπάρχουν γενικοί γραμματείς, οι οποίοι γενικώ είναι διοικητικοί διευθυντές. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μισή ώρα τώρα για να συζητήσουμε με τον ίδιο για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων, η οποία έχει νέες αρμοδιότητες, νέα καθήκοντα, Έχουμε, υπάρχει προσωπικό από τα τρία θεσμικά όργανα σε αυτή τη νέα υπηρεσία. Υπάρχει μια πολιτική α, ε, ε, διευθύντρια, υπάρχει, ε, η οποία είναι και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αναπληρώτρια πρόεδρος της, αντιπρόεδρος της, των εξωτερικών υποθέσεων της Ένωσης. Θα μας πει λοιπόν ο κύριος Σάλιβαν πώς θα επηρεάσει η υπηρεσία του τα δημοσιονομικά μας πράγματα, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις, αν θα υπάρξουν ε, ε, αλλαγές στον ε, προϋπολογισμό σε σχέση και με άλλες υπηρεσίες και επίσης ποια είναι η επιρροή που έχει η δημιουργία αυτές, αυτής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων στα υπόλοι, στις υπόλοιπες 27 υπηρεσίες εξωτερικών δράσεων. Ε, είπαμε ότι η Ευρωπαϊκή αυτή υπηρεσία δεν θα είναι απλώς η 28η υπηρεσία εξωτερικών υποθέσεων, αλλά πρέπει να είναι αποτελεσματική, αποδοτική και πρέπει να δούμε ποιε είναι οι συνέργειε που μπορούν να γίνουν και κατά πόσο μπορούν να γίνουν εξοικονομήσει. Το ερώτημα αυτό το έχουμε θέσει πολλέ φορέ. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση. Αλλά παρόλα αυτά, εάν ο Ντέιβιντ ο Σάλιβαν μπορεί στα 10 λεπτά που έχει στη διάθεσή του να μας απαντήσει, θα το εκτιμούσαμε για να πάρουν το λόγο μετά και οι συνάδελφοι πολύ χρόνο δεν έχουμε, οπότε όποιος έχει ερώτημα προς την ε, ε, Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων, ήδη έχω τρεις, τέσσερις μάλλον στον κατάλογο, πέντε και θα μπορέσουμε νομίζω να απαντήσουμε στα ερωτήματα. Ε, κύριε Οσάλιβαν, έχετε 10 λεπτά για μια μικρή εισαγωγή. Well, thank you very Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία να σας παρουσιάσω την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ζητώ συγγνώμη αν ο τίτλος που κατέχω σας δημιουργεί κάποιες δυσκολίες. Είμαι επικεφαλής διευθυντής προσωπικού. Ε, Δυστυχώ αυτό που σημαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι είμαι υπεύθυνο για ό,τι δεν λειτουργεί και όχι για αυτά που λειτουργούν κανονικά. Από την στιγμή τη θέση σε ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα, και χάρη στη συνεργασία ιδιαίτερως του Κοινοβουλίου η κυρία Άστον προώθησε την άμεση λειτουργία της υπηρεσία αυτής. Αυτό προβλέπεται προβλεπόταν αρχικά στη σύμβαση, μετά στο μελλοντικό στο σύνταγμα το οποίο απορρίφθηκε και τελικά στη συνθήκη. Μια από τι βασικέ μα αρμοδιότητε είναι απλώ να αρχίσει να λειτουργεί αυτή η δομή. Όπω ξέρετε, επί της ουσίας προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε υπάρχοντες πόρους και αυτό προσπαθώ να το, θέλω να το, τονίσω. Τα συστατικά τη υπηρεσία εξωτερική δράση ήδη υπήρχαν και ήδη χρηματοδοτούνταν είτε από τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε του Συμβουλίου. Και αυτό βεβαίω είναι το προσωπικό που ε, ε, βρίσκεται στι Βρυξέλλε. Είναι από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ στο δίκτυο των αντιπροσωπιών σε περίπου 137 χώρε παγκοσμίω. Εκεί υπήρχαν πάλι τη Επιτροπή, αντιπροσωπείε τη Επιτροπή που από την 1η Δεκεμβρίου του 2009 άρχισαν να λειτουργούν και ω αντιπροσωπείε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβαν λοιπόν να εκπροσωπούν την εκάστοτε Προεδρία. Επιπλέον έχουμε δεσμευτεί να συμπεριλάβουμε σε αυτή τη νέα υπηρεσία μια συνιστόσα από τις διπλωματικές υπηρεσίες των κατομελών αυτό μέχρι το τέλος της μεταβατικής περίοδου του 2013 θα είναι ένα τρίτο και ένα τρίτο του προσωπικού θα αποτελείται ακριβώς από αυτό τι υπηρεσίε τη διπλωματική των κρατών με συμβόλαια προσωρινών εργαζομένων, των ΠΟΡΕΡ. Ε, αυτή τη στιγμή λοιπόν βρισκόμαστε στη διαδικασία τη συγκέντρωση αυτού του προσωπικού. Μια από τι βασικέ προκλήσει που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ότι όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε 7, 8, 9 διαφορετικά κτίρια στην πόλη των Βρυξελών. Ε, εδώ βλέπω ένα δύο πρόσωπα γνωστά που είχαν παρακολουθήσει τη συζήτηση στην Επιτροπή Προπολογισμών για να δουν κατά πόσο μπορούμε να βρούμε ένα κοινό κτίριο για να συγκεντρωθεί όλο αυτό το προσωπικό σε ένα μέρο και να αρχίσει να λειτουργεί κανονικά η υπηρεσία μα. Ποιο είναι τώρα το πρώτο ζήτημα. Ποια είναι η αξία αυτή τη υπηρεσία. Όπω είπατε, Πρόεδρε, δεν είμαστε η 28η διπλωματική υπηρεσία, αλλά θέλουμε να προσφέρουμε έργο της στην πολιτική εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για να δούμε τι θα γίνει με τις 27 διπλωματικές αντιπροσωπίες... των κρατών μελών στις τρίτες χώρες ή με τις προξενικές μας αντιπροσωπήσεις στις διάφορες πρωτεύουσες. Ο στόχος είναι να ενισχύσουμε τις σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των ε, μερών που μας αποτελούν, δηλαδή το προσωπικό της Επιτροπής με το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου. Κάποιες φορές ε, τα δύο αυτά σώματα θεσμικώς ήταν διαχωρισμένα. Δεν συνεργάζονταν αποτελεσματικά. Θέλουμε να πάψει λίγο αυτός ο διαχωρισμός, ο διαχωρισμός του μέσου CFSP και του όπως το ονομάζω εγώ, και από την άλλη της Επιτροπής. Θέλουμε να υπάρχει συνέπεια και ολοκλήρωση των διαφορών εργαλείων. Είτε αυτά είναι ο προϋπολογισμός του CFSP, είτε μιλάμε για επιχειρήσεις για τους πολίτες ή στρατιωτικές ή μιλάμε για κοινοτικά εργαλεία τα οποία πολύ καλά γνωρίζει το Κοινοβούλιο και τα οποία παραδοσιακά χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από αυτήν λοιπόν την άποψη ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματική, να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και να έχουμε επιτέλους μια κοινή διαχείριση των ε, εργαλείων, των μέσων, στα πλαίσια των πολιτικών που έχει σχεδιάσει η ε, Λεδιάστον ως ε, εκπρόσωπος και Υπουργός Εξωτερικών και προσπαθούμε εκεί να συνδυάσουμε την προοπτική της Επιτροπής και την άποψη του Συμβουλίου με την παρουσία της ΕΠΑ της Εκπροσώπου και την συνδρομή του Ευρωκοινοβουλίου σε πολιτικό επίπεδο όπως τα πράγματα έχουν συμφωνηθεί και προωθηθεί εδώ. Σε ό,τι αφορά τώρα το μελλοντικό μας προπολογισμό, νομίζω ο επίτροπο Πίμπαλκ θα σα μιλήσει αργότερα σήμερα το πρωί, για την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την αρχική τουλάχιστον άποψη, για την πρόθεση των εξωτερικών σχέσεων και το πώς θα χρηματοδοτηθούν από τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές. Υπό την εξουσία της ε, Άστον και εμείς ε, ως, εξωτερική υπηρεσία, ως υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, προσφέρουμε σε αυτή την ε, μελέτη. Θα δούμε τις ε, προτάσεις της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου μέχρι το καλοκαίρι για το πώς προβλέπεται να διαρθωθεί αυτή η μελλοντική χρηματοδότηση. Σήμερα δεν θα ήθελα να επιμείνω στο θέμα αυτό. Θα αφήσω τον Επίτροπο Πίμπαλξ να σας παρουσιάσει το πολιτικό όραμα της ε, Επιτροπής. Εκ των έσω κιόλα. Τώρα, ως προς το διοικητικά μας έξοδα στον προπολογισμό δεν είναι μεγάλο το επιπλέον κόστος. Ε, συμφωνήθηκε να μας δοθούν κάποιες περαιτέρω θέσεις, να ενισχύσουμε τη θέση κάποιων αντιπροσωπιών, τη δημιουργία της έδρας της υπηρεσίας. Ε, τα μέλη τη Επιτροπής Προπολογισμού θα το ξέρουν ότι κάποιοι χρειάστηκε να μετακινηθούν σε νέα κτίρια, εκεί υπήρξε ένα μικρό κόστο, αλλά σε γενικέ γραμμέ ενοποιούμε τι δαπάνε σε έναν κοινό προπολογισμό, τον προπολογισμό τη ΕΕΔ, η οποία θα υποβληθεί το 2012 ως ξεχωριστό μέρος του προπολογισμού. Ενοποιούμε λοιπόν δαπάνες που είτε βρίσκονταν στον προπολογισμό της Επιτροπής ήδη, είτε της Γενικής Γραμματέας του Συμβουλίου. Οπότε, δεν δημιουργούμε καθαρή επιβάρυνση, αν θέλετε, ε, στο τι επομίζονται οι φορολογούμενοι. Για τη δημοσιονομική αρχή προσπαθούμε μεταξύ κάποιων γεωγραφικών, την επικάλυψη μεταξύ γεωγραφικών αντιπροσωπιών μας στα ίδια σημεία να την εξαλείψουμε σε ό,τι αφορά το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου και των ε, υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσπαθούμε λοιπόν να ενώσουμε τις υπηρεσίες το προσωπικό τη δική μα τη υπηρεσία θα εκπροσωπεί πια αυτού που παλιά εργάζονταν στι εξωτερικέ υποθέσει του Συμβουλίου. Και βεβαίω η Λέδη Άστον θα προεδρεύει ίδια σε τέτοια συμβούλια. Άρα οι αναλασσόμενες προεδρίες είχαν ένα σημαντικό έργο που τώρα το έχουμε αναλάβει εμείς σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές υποθέσει και την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά. Το ίδιο και στις αντιπροσωπείες. Αυτό ήταν μια σημαντική σημαντική δουλειά που ανέλαβαν οι δικές μας ε, υπηρεσίες. Προσπαθούμε να συντονίσουμε το ρόλο μας σε τρίτες χώρες, κάτι που παλιά το διασφάλιζαν οι εναλλασσόμενες προεδρίες. Συντονιστικές συναντήσεις και ούτω καταξής, όλα αυτά διοργανώνται πλέον από τις αντροσωπήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκπροσωπούμε εμείς. Υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών και συντονισμό μεταξύ κρατών μελών που έχουν πρεσβείες επιτόπου όταν τι έχουν και τις αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου καλύπτονται ακριβώ τα βασικά στοιχεία που προηγουμένω τα διασφάλιζαν οι αναλωσόμενε προεδρίε. Αυτό είναι λίγο πολύ ο τρόπο που η ΕΕΔ έχει προσφέρει μεγαλύτερη συνέπεια και έχει εξορθολογήσει τη χρήση των πόρων. Δεν θα έλεγα ότι από οικονομικέ άποψει είναι τεράστια αυτή η αλλαγή. Ε, αν σκεφτούμε τα τεράστια ποσά τα οποία συζητάει η Επιτροπή σας, εδώ μιλάμε για πολύ περιορισμένα ποσά. Όμως, εδώ μιλάμε για ένα σημαντικό βήμα πρόοδου, όπως ή άλλως. Και ένα άλλο ζήτημα που θα πρέπει να απασχολήσει όλους μας είναι ποιες θα είναι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις όλων αυτών για τις εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες. Για την ώρα το ερώτημα αυτό παραμένει ανοιχτό. Δεν ε, ιδρυθήκαμε για να υποκαταστήσουμε τις διπλωματικές υπηρεσίες των δεν είμαστε αντικαταστάτες κανενός, κανενός διπλωμάτη. Από την άλλη όμως, εάν αποδείξουμε την αξία μας και ειλικρινώς νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε, τα κράτη-μέλη ίσως θέλουν να προσαρμόσουν την θεώρησή του των διπλωματικών υπηρεσιών και του διπλωματικού σώματος στη χώρα τους, λαμβάνοντας πλέον υπόψη την ύπαρξη της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μπορεί να στηρίζει ενδεχομένως ε, διοικητικώς ή με άλλα μέσα ε, τα κράτη-μέλη εκεί όπου υπάρχουν εκπροσωποί μα. Αυτέ είναι ορισμένε ιδέε, οι οποίε φαντάζομαι ότι μελλοντικά θα εξελιχθούν από μόνε του. Πάντω, σε καμία περίπτωση δεν έχουμε ήδη μια σειρά προτεραιοτήτων, ούτε έχουμε προγραμματίσει κάτι τέτοιο. Μόλι ιδρυθήκαμε, μόλι αρχίσαμε να λειτουργούμε, πρέπει να αποδείξουμε ότι κάνουμε καλή δουλειά και Είμαστε ευγνώμονε για την εμπιστοσύνη που μα έχουν δείξει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ε, πρόεδρε, θα σταματήσω εδώ, γιατί νομίζω ότι εξάντλησα τα 10 λεπτά, αλλά ευχαρίστω να απαντήσω στι ερωτήσει σα. Αυτή ήταν η αρχική παρουσίαση που είχα να κάνω για τι προκλήσει ίδρυση αυτού του νέου οργανισμού. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Σύντομο, σαφή και πλήρη ο κύριο Σάλιβαν. Οπότε από όλα αυτά που μας είπε μπορούμε να κρατήσουμε την ε, εξοικονόμηση που θέλει να επιδείχει. Θα το δούμε βέβαια αυτό, γιατί όταν μιλούμε για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της υπηρεσίας εξωτερικών δράσεων, πάντα λέμε ότι πρέπει να υπάρχει εξοικονόμηση χρημάτων. Θα το δούμε. Αυτό βέβαια θα πρέπει να το αποδείξει η υπηρεσία, όπως είπατε κι εσείς, θα σας παρακολουθούμε. Λοιπόν, στις 11 θα έρθει ο Επίτροπος Πίμπαλξ. Έχουμε 5-6 στους 6 ομιλητές στον κατάλογο, 7 1 λεπτό για τον καθένα, ώστε να υπάρξει ενδεχομένως και κάποια ε, απάντηση. Ναι, θα είμαι σύντομη, γιατί συχνά έχουμε μιλήσει για την υπηρεσία εξωτερικών δράσεων. Χαίρομαι που ανέλαβε τα καθήκοντα αυτά τη ενοποίηση η υπηρεσία. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει και σε όλε τι ε, υπηρεσίε τη ε, Κομισιόν. Η ΕΦΚΟ έχει πάρα πολλέ. Ε, πολύ, πολύ περισσότερες μάλλον αντιπροσωπίες στην Ευρώπη παρά η υπηρεσία εξωτερικών δράσεων. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η ενοποίηση θα είναι καλή και θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο το καθήκον αυτό, αλλά νομίζω ότι οι εσωτερικές δομές της υπηρεσίας εξωτερικών δράσεων θα πρέπει να έτσι συγκλίνουν, ε, έχουν πάρα πολλά ε, καθήκοντα και ούτως ή άλλως πολλά, πολλές φορές έχουμε ακούσει για διάφορες ε, περιπτώσεις κακοδιαχείρισης που συμβαίνουν στα κράτη-μέλη, οπότε καλό θα ήταν να είναι ένα παράδειγμα η υπηρεσία αυτή. Τώρα, Ποτέ δεν μιλούσαμε για τις ε, αρμοδιότητες αυτής της, υπηρεσία, υπηρεσίας, γιατί μονίμως μιλούσαμε για τον έλεγχο και όχι για τις αρμοδιότητες και αυτό είναι λάθος. Νομίζω ότι πρέπει τώρα να δούμε ότι αυτή η ε, υπηρεσία θα γίνει όντως ευρωπαϊκή, θα, έχει, ας πούμε, θα μπορεί να προσφέρει και προξενικές υπηρεσίες. Ίσως θα μπορούσε ο κύριος Σαλίβα να μας δώσει κάποια αριθμητικά στοιχεία Δηλαδή ποια είναι η προσφορά που φαντάζεται ότι θα υπάρχει προ τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να, δούμε, να έχουμε μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή υπηρεσία. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ο Γιώραν Φέρμ έχει το λόγο. Ε, ε, ευχαριστώ. Για την εξοικονόμηση που ακούστηκε για τα κράτη-μέλη, εντάξει, είναι πολύ σημαντικό, αλλά είναι δύσκολο αυτό προς το παρόν δεν είναι θέμα διοικητικό απλώ, είναι πολιτικό θέμα γιατί ε, ουσιαστικά δεν είναι απόλυτα ε, πεπισμένα τα κρατημέλη που μπορούν να, εμπιστευθούν να ε, αυτή την υπηρεσία. Δηλαδή πρέπει να εξασφαλίσετε και την ανεξαρτησία σας. Είναι πολιτικό θέμα λοιπόν. Έχω ένα ε, πιο συγκεκριμένο θέμα να θίξω. οι συμφωνίες, οι αμοιβέ συμφωνίες και, η, ε, και το ψήφισμα το οποίο επίσης θα, θα, πρέπει και επίσης θα πρέπει να μπουν κάποια αποθέματα, κάποια χρήματα στο αποθεματικό, βέβαια αυτό είναι λίγο μακροπρόθεσμο. Ερώτημα λοιπόν, πού είμαστε, έχουμε την, ε, το αποθεματικό για το προσωπικό. Η ύπατη εκπρόσωπος είπε ότι θα μας ενημερώσει για το, για το προσωπικό Βεβαίω, το θέμα είναι πολύ δύσκολο γιατί πρέπει να υπάρχει και ε, ισορροπία γεωγραφική και ισορροπία μεταξύ των φύλων. Τώρα πού είναι τα πράγματα, πώς έχει η κατάσταση. Έχουμε το παθηματικό για την ενσωμάτωση του πολιτικού προσωπικού για το εργαλείο, από το σχετικό εργαλείο στην ε, Κομισιόν για να αποφύγουμε μεγάλη κυριαρχία των στρατιωτικών υπαλλήλων. Αυτό πού βρίσκεται. Επίση, έχουμε το θέμα τη λογοδοσία, τη διαφάνεια κτλ. Πού είμαστε ως προς αυτό και το θέμα της ενσωμάτωσης των ειδικών απεσταλμένων. Ε, και σε αυτό που είμαστε, τι συμβαίνει. Και τέλος, είδα το οικονομικό πρόγραμμα για το 2012 και 2013. Υπάρχει αύξηση 4, 5, 7% κάθε χρόνο, δηλαδή για τα δύο αυτά χρόνια που απομένουν μέχρι το 2013. Πώς ακριβώς θα αντιμετωπίσετε αυτή την εξέλιξη των επιχειρησιακών δαπανών χωρίς να αυξήσετε το δικό σας το διοικητικό προπολογισμό. Δεν νομίζω ότι ακόμη και τα μέλη της δικής μου ομάδας μπορούν να, έτσι, να ξεπερνούν το χρόνο ε, ούσα εγώ παρούσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι έχουμε πολλά ερωτήματα για το πώς τελικά θα παρουσιάσουμε τα κέρδη, την εξοικονόμηση που θέλουμε να γίνει σε εθνικό επίπεδο ε, μέσω των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων, αλλά πόσο διπλωματική και πόσο ε, διστακτική θα είστε στην ε, διαδικασία αυτή. Γιατί δεν μιλούμε για επιχειρήσεις τώρα. Ε, μιλούμε για το τι θα γίνει μέχρι το 2020. Ε, επικοινωνείτε λέτε με την Κομισιόν για την εκπόνηση των προγραμμάτων και πώς όλο αυτό θα έχει επίπτωση στη δική σας δουλειά. Πώς ακριβώς θα έχετε ένα όραμα συνολικό το οποίο θα ξεπερνά τα βασικά. Ποιος δηλαδή θα κάνει τι στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής είναι η Φρανσίσκα Μπάνκ. Ευχαριστώ διότι ε, αναφέρθηκε ένα σημείο που θα ήθελα να τονίσω και ποια είναι ε, η διαφορά μεταξύ Γενικού Γραμματέως και ε, Διευθύνοντος Συμβούλου διότι η διπλωματία αυτή τη στιγμή είναι σε δύσκολη θέση και οι αποφάσεις λαμβάνονται στα γραφεία των Πρωθυπουργών οπότε πιστεύω ότι ότι θα πρέπει να σκεφτούμε ποια είναι η προστιθέμενη αξία από πλευράς ε, ε, ουσιαστικής και χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό στις διάφορες υπηρεσίες οπότε πιστεύω ότι πρέπει να παλέψουμε να ε, μπορέσουμε να αυξήσουμε το προσωπικό επίσης στις διάφορες υπηρεσίες υπάρχει το θέμα της αποδοτικότητας αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστέ. Δεν μπορούμε να ζητούμε σαν κοινοβούλιο να έχουμε περικοπές σε ένα, δύο, τρία χρόνια διότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης πρέπει να συνεχίσει. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω μπορείτε να αυξήσετε το προσωπικό το οποίο αυτή τη στιγμή περικόπτεται από τους διάφορους οργανισμούς. Ευχαριστώ, κύριος Έλλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να αναφερθώ περισσότερο στο 2020 και το 2025 περισσότερο από ότι οι προηγούμενοι ομιλητές που επικεντρώθηκαν στην τρέχουσα κατάσταση σχετικά με τις διατάξεις της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και την υλοποίησή τους. Λέγουμε συνέχεια ότι δεν έχουμε επαρκή χρηματοδότηση. Τώρα θα μπορέσουμε να έχουμε μία σαφή σαφέστερη ιδέα ποια είναι, ε, ποιο θα είναι το επίπεδο δαπανών στις ε, εξωτερικές δράσεις και ποιες είναι οι παγκόσμιες τάσεις προς το 2020-2025 όπου λέγεται ότι θα αυξάνεται η θέση της Ασίας και της Κίνας. Τι προβλέπετε εσείς για το 2020 για να μπορέσουμε να αναπροσαρμόσουμε τις τωρινές καλοκαιρινές διακοπές αντί σιγά σιγά ε, να βρεθούμε σε μια θέση που δεν θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους μελλοντικούς στόχους της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Και εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε επαρκή χρηματοδότηση και η κατάσταση δεν βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου. Αν μιλήσουμε ε, για τη Βόρειο Αφρική και τις εξελίξεις εκεί και την Μέση Ανατολή πιστεύω ότι η χρηματοδότησή μας δεν επαρκεί. Ο Μιγγέλ Πόρτας. Ευχαριστώ. Ε, καταρχήν θα ήθελα να πω το εξής. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη για ένα κτίριο όπου όλο το προσωπικό μπορεί να συναντάται και η δουλειά να γίνει πιο εύκολη. Αυτό το οποίο δεν μπορώ να αντιληφθώ είναι στα πλαίσια της, ε, ε, της περιστολής τι θα γίνει με τα κτίρια. Δηλαδή τι θα γίνει με ένα κτίριο το οποίο θα πρέπει να αποπληρώνεται επί τρία χρόνια που έχει ε, μεγάλο κόστος κατασκευής θα είναι αποτελεσματικό γιατί για να είμαι ειλικρινής πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε ε, να ε, δώσουμε ε, μια μεγαλύτερη αξία στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης εφόσον έχουμε συγχρόνως να αντιμετωπίσουμε τα προγράμματα περιστολής των εθνικών κρατών και των κυβερνήσεών τους. Επίσης αντιλαμβάνουμε ότι έχετε αμφιβολίες για το εάν πρόκειται ε, να αποτελέσει υπηρεσία ε, αυτή απλώς μία 28η διπλωματική ε, υπηρεσία. Πρέπει να έχουμε ένα σαφές πλαίσιο για την αντικατάσταση των διαφόρων λειτουργιών σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Όταν μιλάμε για τις εξωτερικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ενώσεως σκεφτόμαστε τη συνθήκη της Λισαβόνες και την προσπάθεια την οποία προσπαθούμε να κατατήσουμε κατά τρόπον ώστε ε, να εφαρμόσουμε και να αναβαθμίσουμε την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως διεθνώς διότι θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος ε, δωρητή στην, ε, ε, ε, στην Ευρώπη και συμβάλλει εις την ανάπτυξη πολλών χωρών. Όταν όμως μιλάμε για την εξωτερική αγορά και την εξωτερική δράση δεν μιλάμε για συντονισμένες προσπάθειες σκεφτώ όπως είναι παραδείγματος χάρη η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά σκεφτόμαστε ότι θα υπάρξει ε, μία υπηρεσία η οποία θα χρηματοδοτείται από άλλες ευρωπαϊκές πηγές και η υπηρεσία αυτή διπλωματικά θα συμβάλλει στην επιτυχία των προγραμμάτων με τον τρόπο που προανέφερα. Πρέπει λοιπόν να μιλάμε για κοινή ε, διαχείριση από όλες αυτές τις υπηρεσίες, να υπάρχει ένα μοναδικό γραφείο στις χώρες όπου όλες αυτές οι υπηρεσίες εκπροσωπούνται και να δημιουργήσουμε μία ε, ε, επιτροπή εργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, της, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, της Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσης. Ευχαριστώ. Κύριε Σάλιβαν, φαντάζομαι ότι μπορείτε να απαντήσετε, ε, διότι δεν νομίζω ότι θα μπορέσετε να απαντήσετε σε όλες ε, στο χρόνο τον οποίο έχετε, αλλά ξεκινήστε. Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω ούτε να αποφύγω να απαντήσω ούτε να σας απασχολήσω υπερβολικά οπότε παρακαλώ να, με, να μου κάνετε ένα σήμα αν νομίζετε ότι παρεκτρέπομαι χρονικά διότι πολλά θέματα μπορούν να χρειαστούν ώρες για να συζητηθούν εν πάση λεπτομερία σχετικά με την ερώτηση της κυρίας Γκρέσλε συμφωνώ απολύτως ότι χρειαζόμαστε ένα πολύ καλό ορισμό του, ε, του, ε, των καθηκόντων μας και της αποστολής μας. Έχουμε ε, ε κληρονομήσει μία σειρά ε, καθηκόντων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τις αντιπροσωπείες και ούτω καθεξής. Άρα ο πρώτος μου ρόλος είναι να εξασφαλίσω ότι θα υπάρχει μία συνέχεια και ότι θα εκτελούμε τα καθήκοντά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πράγμα όμως το οποίο δεν ε, μας εμποδίζει και αυτό είναι σαφές ε, και μας το έχει ξεκαθαρίσει η κυρία Άστον ότι δεν ε, πρέπει να καταρτήσουμε ένα κατάλογο προτεραιοτήτων βάσει των οποίων θα καθορίσουμε τι πρέπει να μας αποσχολήσει κατά προτεραιότητα τα επόμενα χρόνια και τι είναι υποδέστερο. Θα καταλάβετε ότι και πάλι εδώ προσπαθούμε να καταρτήσουμε μία οργάνωση, να εξασφαλίσουμε την συνέχεια και να κάνουμε έναν, μία προβολή προς το μέλλον, καλύπτοντας πάντοτε όλα μας τα καθήκοντα. Πρέπει όμως να σας πω ότι όλα αυτά τα θέματα από γεωγραφικής απόψεως και ισοτιμίας των φύλων η κάθε Άστερ έχει πει ότι πρόκειται για μία πρόκληση ιδίω η ισότητα των φίλον έχω προσπαθήσει να την εφαρμόσω κατά το χρόνο που ήμουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, είτε μιλάμε για την Επιτροπή είτε για το Συμβούλιο ή για τις εθνικές ε, υπηρεσίες προσπαθούμε να εξισορροπήσουμε μία μονόπλευρη αντιμετώπιση των φύλων και προσπαθούμε να βελτιώσουμε την προοπτική από, τους, από τη ε, σε σχέση με την κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα από τα οποία προερχόμαστε. Τώρα, ε, όσον αφορά τους προγραμματιστές της εξωτερικής δράσης που έχει έχει, έχουν απασχολήσει την Επιτροπή σας. Νομίζω ότι όσον αφορά το προπολογισμό και το προσωπικό νομίζω ότι επαρκούμε αλλά το ουσιαστικό ερώτημα είναι ότι πρέπει να δούμε ποιος είναι ο στόχος για το 2020 και πιστεύω ότι ο Επίτροπος Σπίλμπαξ θα σας πει τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι στη νέα γενιά και στα προγράμματα πρέπει να δούμε δούμε πώς ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις του 21ου αιώνα σε ένα χώρο από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό πώς θα μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε των προκλήσεων δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει σωστή κλίμακα όπως είπε ο πρόεδρος Μπαρόζο πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα ε, στα οποία όμως θα απεμπολίσουμε ορισμένα στοιχεία εθνική κυριαρχίας. Τι θα χρειάζεται λοιπόν, πώς θα χρησιμοποιήσουμε και ποια μέτρα για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις οι οποίες θα προκύψουν στην επόμενη, στα επόμενα χρόνια και θα πρέπει συγχρόνως να υπάρξει αξιολόγηση και μία διαδικασία αξιολογήσεως της μετατόπισης των προτεραιοτήτων διότι εγώ αυτό το οποίο θέλω να επιτύχω εις τη την υπηρεσία εξωτερικής δράσεως είναι να γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε τι μέλη γενέσαι. Εάν λοιπόν έχουμε ε, μία προοπτική πενταετή προπολογισμού θα δούμε ότι ναι μεν μας καλύπτει για τον πρώτο χρόνο, το δεύτερο χρόνο απέχουμε και τον τρίτο χρόνο ψαχνόμαστε. Πρέπει λοιπόν να προγραμματίσουμε σωστά τη χρηματοδότηση με κάποια όμως ευελιξία για να αντιμετωπίσουμε νέες κρίσεις εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να προσθέσουμε και να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση η οποία είναι ήδη διαθέσιμη από το, όσον αφορά την ερώτηση της κυρίας Μπραντνερ ε, για την ε, ε, διαχείριση κρίσεων πρέπει να πούμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν μας έχει απασχολήσει χρειαζόμαστε περισσότερες μελέτες και πρέπει να δούμε πώς θα το οργανώσουμε καλύτερα διότι μέχρι στιγμής απλώς έχουμε προσαρμόσει τις δομές αυτές ο σύστημα σύστημα. Θα επανέλθουμε στο Κοινοβούλιο επ' αυτού και στην, ε, ε, στην προσθήκη 10%, 10 αποδοτικότητος, κυρία Μπράντνερ, θα πρέπει να δούμε πού θα αναφερθεί. Δηλαδή αν πρόκειται για την ενεργειακή πολιτική, την πολιτική ασφαλείας ή άλλους τομείς όπου χρειαζόμαστε προσωπικό που δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή. Πώς δηλαδή θα αναπτυχθούν ε, τα κέρδη αποτελεσματικότητος ε, από το Συμβούλιο και την Επιτροπή με λιγότερη επικάλυψη. Ε, επίσης ε, θα ήθελα να σας πω ότι τελικά δεν υπάρχει περισσότερο κόστος με το να συγκεντρώσουμε τους υπαλλήλους σε ένα κτίριο διότι απλώς δεν θέλουμε όπως είμαστε τώρα διασπαρμένοι να υπάρχει συγκέντρωση με το ίδιο όμως ο κόστος και ε, όσον αφορά τη διπλωματική υπηρεσία θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει και επιπλέον προστιθέμενη αξία ε, για και αυτό να αποδειχθεί καλύτερα ιδίως στα πλαίσια της εναλλασσόμενης προεδρίας και άπαξ και γίνει αυτό όπως και άλλοι σχολίασαν θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνέργεια μεταξύ ημών και των εθνικών διπλωματικών ε, κάτι το οποίο ελπίζω ότι μακροπρόθεσμα θα επιτευχθεί. Ελπίζω λοιπόν ε, κυρία Πρόεδρε ότι παρόλο που δεν απάντησα σε όλα τα ερωτήματα δεν θέλω να υπερβώ το χρόνο μου είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον είναι ε, ένα επίτευγμα του Κοινοβουλίου ένα παιδί του Κοινοβουλίου στον τομέα αυτό και χαίρομαι που συμβάλλω έχουμε προκλήσεις και διοικητικές και πολιτικές θα τις αντιμετωπίσουμε από κοινού και η κυρία Άστον προσπαθεί να απαντήσει και ε, να ανταποκριθεί στις ερωτήσεις που θέσατε για να αποδείξει ότι είναι ένας τομέας όπου η Ευρώπη μπορεί να διαμορφώσει τον 21ο αιώνα και να μην διαμορφωθεί απλώς από άλλους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης και για την ε, ακριβέστατη και σύντομη απάντηση στα πολυάριθμα ερωτήματα που σας είχαν τοποθετηθεί. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ και όπως άκουσα ο Επίτροπος Πίμπαλς έχει ήδη έρθει, δεν ξέρω αν είναι έξω από την αίθουσα αλλά θα ήθελα να πω ένα πράγμα προτού του ζητήσω να έρθει. Αυτά τα οποία είπατε και είμαι βέβαιη ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία θα εμβαθύνουμε την επόμενη μια μισή ώρα. Εάν στις, ε, στην επόμενη δημοσιονομική ε, προοπτική χρειαστούμε ε, ορισμένες προοπτικές νέες ακόμη και για την εξωτερική υπηρεσία για να υπάρξει η ευελιξία που χρειαζόμαστε και χρειαστεί να παλέψουμε για όλα αυτά. Ελπίζουμε ότι θα συνεργαστείτε μαζί μας και θα είσαστε μαχητές στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ. Και τώρα θέλουμε να καλωσορίσουμε So, wir heißen äh, den Kommissar ganz herzlich willkommen. Να καλωσορίσουμε τον Επίτροπο. Μόλις έφτασε στις Βρυξέλλες. Και χαίρομαι που βρήκε και χρόνο να είναι εδώ στην Επιτροπή μας. Την επόμενη, λοιπόν, μια μισή ώρα θα μιλήσουμε για την πολιτική ανάπτυξης και την εξωτερική πολιτική. Ο Επίτροπος είναι εδώ και για την εξωτερική πολιτική και για την ανάπτυξη. Ο Επίτροπος ε, Πίμπαλξ είναι ο μόνος που ασχολείται με την ε, εξωτερική πολιτική και έχει σχέση με την ε, υπηρεσία εξωτερικών υποθέσεων, εξωτερικών δράσεων για την εκπόνηση των μελλοντικών δημοσιονομικών προοπτικών. Ως συνήθως, Θα ακούσουμε για πέντε λεπτά το Σαλβαδόρ και μετά ο Επίτροπος Πίμπαλξ θα πάρει τα δέκα λεπτά που του αναλογούν για να κάνει την ε, δήλωσή του. Μετά θα ακούσουμε τις ε, ομάδες. Θα σας δώσω τέσσερα λεπτά γιατί μετά θα έχουμε πάλι πρόβλημα για να χωρέσουν όσοι θέλουν να κάνουν ερωτήσεις στον Επίτροπο να μπορέσουμε λοιπόν να εξυπηρετήσουμε τους πάντες. Λοιπόν, Σαλβαδόρ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε τον Επίτροπο Πίμπαλξ που είναι βετεράνος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εφόσον έχει αναλάβει τόσο δύσκολα θέματα όπως τις ενέργειες στο παρελθόν. Και τώρα έχει επιφορτιστεί με την εξωτερική πολιτική, την πολιτική ανάπτυξη, θέματα που τραβάνε την προσοχή του κοινού ιδιαίτερω. Για τι ερχόμενε δημοσιονομικέ προοπτικέ, το θέμα των εξωτερικών ε, σχέσεων προφανώς θα αποτελέσει προτεραιότητα και για το Ευρωκοινοβούλιο και Ό,τι μορφή και να πάρουν τελικώ οι δημοσιονομικέ προοπτικέ, η εξωτερική πολιτική θα αποτελεί ένα κεφάλαιο ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα. Και εφόσον δεν καλύπτεται από τη στρατηγική 2020. Χρειάζεται λοιπόν εδώ να τοποθετηθούμε σαφώς και να υπογραμμίσουμε τη σημασία της πολιτικής αυτής για το ερχόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πρόκειται για ένα κεφάλαιο που δεν έχει ως τώρα χρηματοδοτηθεί επαρκώς. Μιλάμε για μια κατηγορία εξωτερικών σχέσεων σε όλες τις δημοσιονομικές προοπτικές που εγώ τουλάχιστον έχω γνωρίσει ως τώρα. Πιστεύω ότι το πρόβλημα της ε, χαμηλής χρηματοδότησης ως τώρα ήταν σοβαρό. Ε, το ζήτημα της ε, εξωτερικής, της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης μας το παρουσίασε με λαμπρό τρόπο ο Διευθυντής Προσωπικός Άλιβαν. Τώρα πρέπει να δούμε, κύριε Επίτροπε, πώς η εξοικονόμηση θα μας επιτρέψει να πετύχουμε αυτή η υπηρεσία στις εξωτερικές σχέσεις και πώς θα βελτιώσει τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλα μέρη του κόσμου. Πώ θα συσχετιστεί με την πολιτική συνοχή και πολιτική Εδώ πώς θα συνδυάσουμε τους στόχους και τα πολιτικά μας μέσα, ώστε να ανταποκρίνονται στα, στις πολιτικές δεσμεύσεις και τα πολιτικά μέσα που διαθέτουμε. Ιδίως για χώρες που είναι υποψήφιες για ένταξη μεσοπρόθεσμα. Νομίζουμε ότι οι σχέσεις μεταξύ της Ένωσης και των χωρών αυτών θα πρέπει να αλλάξουν ολοσχερός. Για να γίνει λοιπόν αυτό θα πρέπει να προβλέψουμε επίπεδα ανάπτυξης και οικονομικής αύξησης πολύ ανώτερα για τις χώρες αυτές και θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια διαφοροποιημένη προσέγγιση χάρη στην προσέγγιση που θα έχουμε στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων και αντιστρόφως για τις χώρες που έχουν καλύτερα αποτελέσματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, για τις ισχύουσες δημοσιονομικές προοπτικές, είναι σαφές ότι για να έχουμε περισσότερη αποτελεσματικότητα στην απονομή των κονδυλίων σε αυτόν τον τομέα των εξωτερικών ε, υποθέσεων και των εξωτερικών σχέσεων, είναι απαραίτητο τα προγράμματα με γεωγραφική διάσταση να συμβάλλουν περισσότερο και να ενισχύονται από το μέσο σταθερότητας. Ποια είναι η εξωτερική διάσταση, Επιτροπή, των εσωτερικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς θα συμπεριληφθούν στο ερχόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο με συγκεκριμένα μέσα που θα δημιουργηθούν επί τόπου ή θα συνδυάσουμε την εξωτερική διάσταση με τις υπάρχουσες ε, πολιτικές αναγεωγραφική περιοχή. Πιστεύετε ότι η εξωτερική διάσταση των ε, εσωτερικών πολιτικών της Ένωσης θα πρέπει να παραμένουν στην θέση που ήδη βρίσκονται στον προπολογισμό ή να αλλάξουν κατηγορία και θέση. Για το Ταμείο της Ανάπτυξης. Εδώ το Κοινοβούλιο έχει απαιτήσει αξί το όμω οι νέε δημοσιονομικέ συνθήκε δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα, πιστεύουμε. Και θα είναι ακόμη πιο δύσκολο να υλοποιηθεί, να λάβει σάρκα και ωστά η επιθυμία αυτή του Κοινοβουλίου. Ποιο θα είναι λοιπόν ο αντίκτυπο στι μελλοντικέ δημοσιονομικέ προοπτικέ. Και ακόμη μια ερώτηση προ τον Επίτροπο. Για τους απαραίτητους δημοσιονομικούς πόρους, τι όγκο θα φτάσουν οι πόροι αυτοί, ώστε να φέρουμε σε αίσιο πέρα την ε, πολιτική εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύετε ότι η πόροι μα ως τώρα ήταν επαρκή. δεν νομίζετε ότι θα έπρεπε να αυξηθεί το σύνολο των ε, πηγών και των πόρων. Και αν ισχύει αυτό, νομίζω ότι και οι υπόλοιποι επίτροποι που ασχολούνται με δαπάνε του προπολογισμού θα έχετε σκεφτεί και συζητήσει όλοι μαζί νέα μέσα χρηματοδότησης, νέα χρηματοδοτικά μέσα, όπως την ε, αποτελεσματικότερη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. φαντάζομαι ότι όλο και περισσότερο επιβαρύνουμε την τράπεζα αυτή με απαιτήσει και οι διάφοροι επίτροποι που έχουν παρελάσει στην Επιτροπή μας θα έχουν ακούσει αυτά. Πώς διαβλέπετε λοιπόν εσεί αυτή τη διασύνδεση της τράπεζας με την εξωτερική πολιτική. Το μόνο μέσο που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή είναι η ευελιξία. Ω τώρα έχουμε λάβει χαμηλή χρηματοδότηση τη εξωτερική πολιτική μέσω της εντατικής χρήση του μέσου της ευελιξίας. Αυτό ήταν αναπόφευκτο τώρα. Και ακόμη μια ερώτηση, που μας, ε, ένα θέμα που μας είναι προσφυλές. Πώς η γενική σας διεύθυνση θα βοηθήσει την αναχέτηση των ε, αρνητικών συνεπειών από τις κλιματικές αλλαγές και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Έχει δεσμευτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλει ένα εκατομμύριο ευρώ από τώρα στο 2012 για το σκοπό αυτό. Τι ακριβώς θα γίνει η δέσμευση αυτή θα διατηρηθεί μακροπρόθεσμα και αν ναι, πώς θέλετε αυτό να συμπεριληφθεί σε μια διάρθρωση δημοσιονομικών προοπτικών πιο περιοριστική από τη σήμερα. Και άλλη μια σειρά ερωτήσεων. Ο Επίτροπος έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Σιγητά, αξιότιμα μέλη, Όντω, ο εισηγητή έθεσε πολύ σημαντικά ερωτήματα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα περισσότερα. Ελπίζω όμω να μπορέσω να απαντήσω πιο λεπτομερώ και, και στι ερωταπαντήσει. Το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να το δούμε στο νέο θεσμικό του πλαίσιο. Η, συνθήκη τη Λισαβόνα θέτει ένα νέο, ένα νέο πλαίσιο για τι εξωτερικέ δράσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θέτει και του στόχου. Το νέο μα θεσμικό ε, πλαίσιο είναι η δημιουργία τη υπηρεσία εξωτερικών δράσεων, δίνοντα την Ευρωπαϊκή Ένωση την ικανότητα να έχει ευρωπαϊκή προσέγγιση προς τις εξωτερικές δράσεις. Αυτό δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την, την δυνατότητα να έχει στενότερη σχέση μεταξύ πολιτικών προτεραιοτήτων, διακυβέρνησης των ε, σχέσεων μας με τις υπόλοιπες χώρες και θέτει το πλαίσιο για την βοήθεια που θα δίνουμε. Επίσης, οι, το, το, οι δαπάνες μετά το 2013 θα πρέπει να συνάδουν με τις ε, προτεραιότητες της στρατηγικής 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, το δίκτυο με τις διεθνείς συμβάσεις ε, με τους εταίρους σε όλο τον κόσμο δίνει ένα εξαιρετικό δυναμικό για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, οικονομία κλίμακος και ορατότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την, ε, τον, απαραίτητο, τον απαραίτητο τρόπο για να αντιμετωπίσει τις ε, προκλήσεις που είναι οι κλιματικές αλλαγές και η μείωση της φτώχειας. Επίσης, έχει τη δυνατότητα και την αξιοπιστία που είναι αναντικατάστατες όταν μιλούμε για ανθρώπινα δικαιώματα, ε, παρατήρηση εκλογών, ε, διακυβέρνηση και διαχείριση κρίσεων. Είναι, ε, έχει λοιπόν τη δυνατότητα να καλύψει ανάγκες που έχουν να κάνουν με την ανθρωπιστική βοήθεια σε παγκόσμιο επίπεδο, ταυτόχρονα και σεβόμενοι τα όσα, δίνονται στην, τα όσα ε, θεσπίζονται σε διεθνεί ε, συμβάσει. Επίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει την εξωτερική αυτή υπηρεσία με αποτελεσματικό τρόπο, να την διευκολύνει ώστε να, να επιτύχει τι ε, προτεραιότητέ τη σε συνάφεια πάντα με, το παγκόσμιο οικονομικό, με την παγκόσμια οικονομική και πολιτική σημασία που έχουν όλα αυτά. Πρέπει στενά να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη, του στρατηγικού εταίρου και, και τι διεθνεί φορεί για τις ε, δημοσιονομικές ε, ε, προοπτικές μας μπορούμε να έχουμε βοήθεια και προς τις γειτονικές χώρες. Οι προσπάθειές μας ξεπερνούν την περιφερειακή ενσωμάτωση και την αντιμετώπιση της φτώχειας και πρέπει να επέμβουμε μαζί με στρατηγικούς εταίρους ώστε στο μέλλον να μπορέσουμε να λύσουμε παγκόσμιες κρίσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διατηρήσει ένα πολιτικό, μια μακροχρόνια πολιτική δράση για τις εξωτερικές υποθέσεις συμπεριλαμβάνοντας και θέματα ασφάλεια, ώστε να, εξασφαλίσουμε την συνέχεια στις εξωτερικές δράσεις. Η οστατική μα στοχοθέτηση μετά το 2013 θα πρέπει να υποστηρίζει την επίτευξη έξι βασικών στόχων. Ε, μία ατζέντα αντιμετώπιση τη φτώχεια, που είναι ολοκληρωμένη και επικεντρώνεται στην ε, βιώσιμη ανάπτυξη στι αναπτυσσόμενες χώρε. Μία ειδική σχέση με τι ε, όμορε χώρε, με τον στόχο δημιουργίας ενός χώρου σταθερότητας και ευημερίας και, προετοιμάζοντας και προετοιμασίας των, ε, των υποψηφίων χωρών για ένταξη οι νέες διατάξεις της ε, συνθήκης για την ε, ανθρωπιστική ανάγκη για την προστασία θα πρέπει να συμπληρωθούν και από τα νομικά εργαλεία. Μία ατζέντα που θα αφορά την ε, Τι ε, αμοιβέ σχέσει μεταξύ βιομηχανοποιημένων χωρών και των αναδειωμένων οικονομιών ε, σε συνάφεια με του στρατηγικού εταίρους. Επίση, η μοντέρνα και αποτελεσματικά εργαλεία θα πρέπει να υπάρξουν ώστε να αντιμετωπιστούν οι κρίσει και ψηφίσματα. Και η ευρωπαϊκή ηγεσία θα πρέπει να είναι σημαντική ώστε να αντιμετωπίσει προκλήσει όπω κλιματικέ αλλαγέ, βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία των παγκόσμιων δημοσίων αγαθών η συνθήκη τη Λισαβόνα έχει δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την εντολή να επιταχύνει το ρόλο τη, να ενισχύσει το ρόλο τη ω παγκόσμιο παίκτη. Αυτό λοιπόν το υψηλό επίπεδο προσδοκιών θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στο επίπεδο χρηματοδότηση για τι εξωτερικέ δράσει. Παρ' όλα αυτά, Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι η Κομισιόν τώρα μελετά όλες τις πτυχές του νέου δημοσιονομικού πλαισίου και γι' αυτό προς το παρόν είναι πολύ νωρί για να σα δώσω οποιαδήποτε ε, αριθμητικά στοιχεία η βασική αρχή, οι βασικές αρχές που πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ορίζουν τις, ε, τις δημοσιονομικές μας στο μέλλον αναφέρονται στο, στην αναθεώρηση για τον προβολισμό και τη σχετική ανακοίνωση του Οκτωβρίου. Ε, πρέπει να έχουμε τρεις βασικούς στόχους. Να έχουμε αποτελέσματα, να προσπαθήσουμε να έχουμε ε, μόχλευση σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο και να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Εάν θέλουμε να επικεντρωθούμε στα αποτελέσματα, θα πρέπει να ε, ε, ελέγξουμε ε, τις επιπτώσεις των δράσεων και των προτεραιοτήτων μας. Όσο πιο ψηλά είναι οι επιπτώσεις των προτεραιοτήτων μας, τόσο πιο, ψηλά, πιο ψηλή θα είναι και η αποτελεσματικότητά μας. Επίσης, προσπαθούμε να, να κερδίσουμε και σε αποτελεσματικότητα, τονίζοντας περισσότερο την οικονομική μόχλευση και την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών πόρων και στην πολιτική μόχλευση. Επίσης, πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία ισορροπία μεταξύ προβλεψιμότητας και ευελιξίας. Και θα πρέπει να δούμε το θέμα της αιρεσιμότητας ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όλα αυτά θα συνάδουν και θα, συμπληρώνονται από καλή διακυβέρνηση. Επίση, πρέπει να έχουμε μεγαλύτερο περιθώριο για απλούστευση και για streamlining στην, σε ό,τι αφορά τα εξωτερικά εργαλεία αυτή η αρχή θα πρέπει να χρωματίζει την ε, ε, προσέγγιση μας για τον τίτλο για, την εξωτερική, τις εξωτερικές δράσεις και θα επικεντρωθώ σε τέσσερις δομές που πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να ε, αφορούν τον, που αποτελούν μάλλον τον, το μεγαλύτερο όγκο των, των κονδυλίων για τις εξωτερικές δράσεις έχοντας υπόψη και τους, και τους στόχους της ε, της χιλιετίας και το 0,7% που θέλουμε να επιτύχουμε μέχρι το 2015 πρέπει να έχουμε γενική ε, αύξηση των, ε, των κονδυλίων για την αναπτυξιακή βοήθεια. Εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει το ρόλο που της αναλογεί. Μία πιο διαφοροποιημένη προσέγγιση σύμφωνα με την ανάπτυξη και το επίπεδο ανάπτυξης των χωρών και των γεωπολιτικών αλλά και οικονομικών θέσεων θα μας επιτρέψει να επικεντρωθούμε σε ευρωπαϊκό, ε, ευρωπαϊκό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την αμοιβαία ε, αναγνώριση συμφωνιών με Κίνα, ε, Ινδία και άλλες χώρες καθώς επίσης και πιο φτωχές χώρες ή πιο ευαίσθητες. Αυτοί, αυτές οι αρχές της διαφοροποιημένης προσέγγισης θα πρέπει να ε, ενσωματωθούν ε, στι μελλοντικέ νομοθετικέ προτάσει και στην αρχιτεκτονική των μελλοντικών εργαλείων μας. Αυτό συνεχίζει να μελετάτε. Η Κομισιόν έχει επαναλάβει την πρόταση για το EDF ε, για λόγους πολιτικής λογοδοσίας και δημοκρατικού ελέγχου για την περίοδο πέρα από το 2013. Αυτά τα επιχειρήματα είναι, παραμένουν, παραμένουν ενισχύ. Ε, θεωρώ ότι είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παίξει σημαντικό ρόλο στη συνεργασία με τι ε, ε, χώρες ΑΚΕ. του λεχθέντο, στην συζήτηση που γίνεται για τον προπολογισμό, θα πρέπει χωρίς αμφιβολία να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίε που μας τίθενται από την δύσκολη οικονομική κατάσταση τώρα, που αφορούν το γενικό επίπεδο κονδυλίων για την ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, πέραν των, της γεωγραφικής συνεργασίας, η, θεματική, η εκπόνηση θεματικών προγραμμάτων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο θα μπορέσουν να στηρίξουν τη στρατηγική και την ορατότητα των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορέσουν να υποστηρίξουν συγκεκριμένους τομείς και θα μπορέσουν να θίξουν συγκεκριμένες προτεραιότητες που δεν καλύπτονται προς το παρόν ε, επαρκώς από γεωγραφικά εργαλεία. Θεωρούμε ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία στο να διατηρήσουμε τα παρόντα θεματικά προγράμματα, αλλά υπάρχει δυναμικό για να στοχοθετήσουμε ε, το πλαίσιο επικεντρώνοντάς το σε οριζόντιες, παγκόσμιες και διεθνικές δράσεις σε τομείς όπως η βιώσιμη ενέργεια, ε, ασφάλεια τροφίμων, ε, κλιματικές αλλαγές, μετανάστευση για να πω μερικά. Επίσης θα πρέπει να μελετήσουμε το αν ένα θεματικό πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που έχουν να κάνουν την, ευαλω... την ε, ε, ευαλωτότητα ευαισθησία των χωρών μπορεί να αντιμετωπιστεί. Επίσης μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε τέτοια προγράμματα και να, ε, έχουμε, να μπορέσουμε να επιτύχουμε δράσεις υψηλής αποτελεσματικότητας. Επίσης, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών πρέπει να βελτιωθούν, ενισχύοντας την συνεργασία συνεργασία, σε κοινά προγράμματα μπορούμε να ε, κάνουμε μεγάλη πρόοδο στο να, αντιμετωπίσουμε, να ε, βελτιώσουμε ε, την ορατότητα των δράσεων τη υπηρεσία εξωτερικών δράσεων. Επίσης, σε ό,τι αφορά τη μόχλευση, στην πράσινη βίβλο που δημοσιεύθηκε το φθινόπωρο, η στοχοθέτηση μιλά για, την, για την καλύτερη κατανομή δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων. Η αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αποτελέσει τον καταλήτη. Για να μπορέσουμε λοιπόν να έχουμε μόχλευση και να πολλαπλασιάσουμε τους πόρους μας πρέπει να έχουμε μια καλή εταιρική σχέση συμπεριλαμβανομένης και της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρική Τράπεζας, ε, Επενδύσεων συγγνώμη, αλλά και άλλων εταίρων. Η χρήση καινοτόμων εργαλείων ε, όπως α πούμε τα δάνεια ή η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για Συνεργασία και Ανάπτυξη θα μπορέσουν να υποστηρίξουν αυτό το στόχο μα. Η πολιτική δέσμευση, Πρόεδρε, τρία λεπτά αν μου δώσετε ακόμη. Εντάξει, ωραία. Τρία λεπτά. Η πολιτική δέσμευση λοιπόν έναντι των υποψηφίων χωρών, των πιθανών υποψηφίων και των όμορων χωρών βασίζεται στη συνθήκη και έχει επιβεβαιωθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η, η οικονομική βοήθεια σε αυτές τις χώρες είναι άμεση συνέπεια αυτής της πολιτικής δέσμευσης. Αλλά ε, είναι και επένδυση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σταθερότητα στην, στους, στην ε, γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένω, είναι στο, προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δομή για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής διεύρυνσης ορίζεται σαφώς. Ξεκινώντας με την ε, σταθεροποίηση και την, και την διαδικασία ένταξης, η χρήση των εργαλείων αυτών έχει αποδείξει την χρησιμότητά της ώστε να βοηθήσει τις, και να καθοδηγήσει τις χώρες τις επιλέξιμες στην ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του πολιτικού διαλόγου και των διαπραγματεύσεων. Ε, τα εργαλεία αυτά, για τον τομέα αυτό, έχουμε το προενταξιακό εργαλείο, το οποίο θα συνεχίσει να προετοιμάζει τις ε, υποψήφιες χώρες για την ένταξη το Ευρωπαϊκό ε, Εργαλείο ε, Εταιρική ε, Σχέση και Γειτονία θα πρέπει να συνεχίσει να μιλά για την ολοκλήρωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δημιουργία ενό Ευρωπαϊκού χώρου ευημερία και καλή γειτονία στα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι, οικονομικοί πόροι τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μπορούν να καλύψουν του πολιτικού τη στόχου. Θα πρέπει επίση να δοθεί σημασία στη δυνατότητα προοδευτική διαφοροποίηση μεταξύ κρατών ε, Όπω επίση και αυτό πρέπει να συμβεί και στην, ε, στον τομέα τη αναπτυξιακή βοήθεια. Τώρα για τι φυσικέ και τις ανθρωπογενείς καταστροφέ που ε, ενισχύονται από την πίεση των πολιτών. Η ανάγκη που υπάρχει για την ανθρωπιστική βοήθεια στους πιο ευαίσθητους πληθυσμούς του θα αυξηθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ανθρωπιστικής βοήθειας και επομένως είναι σημαντικός παίκτη στην ε, στην παγκόσμια σκακέρα. Η ε, ενίσχυση λοιπόν των δραστηριοτήτων αυτών θα βοηθήσει μέσω μεγαλύτερη ευελιξία. Πρέπει να υπάρξουν περισσότερε προσπάθειε για να δούμε πώ θα βελτιώσουμε το εργαλείο ε, ε, ευελιξία και, και το αποθεματικό που υπάρχει για τι επίγουσε ανάγκε. Επίση θα πρέπει να δούμε κατά πόσο το τελευταίο θα μπορέσει να ενισχυθεί με μια πολυετή διάσταση. Θα πρέπει να υπάρχουν απαραίτητα, τα απαραίτητα κονδύλια ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προβλέψιμες ή προβλεπόμενες καταστάσεις στα επόμενα χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης πρέπει να εξοπλιστεί καλύτερα για να βελτιώσει την παρέμβασή της σε κρίσεις και σε μεταβατικές περιόδους. Οι υποχρεώσει από την συνθήκη για την αντιμετώπιση ε, των κρίσεων και την ε, εγκαθίδρυση τη ειρήνη είναι ένας βασικός στόχος των εξωτερικών δράσεων που καθορίζει και τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ένα τρόπος για να, αντιμετωπίσουμε, για να εξελίξουμε τα εργαλεία μας περισσότερο είναι να τα ανασχεδιάσουμε. Το εργαλείο για την σταθερότητα ε, επιτρέποντας ευέλικτε παρεμβάσεις με ε, συγκεκριμένη διασύνδεση με την ε, εγκαθίδρυση της ειρήνης. Αυτό μπορεί να γίνει και για την ανθρωπιστική βοήθεια και να και να διευκολύνει την ανοικοδόμηση των χωρών αυτών. Το CFSP και το CSDP επίσης θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Αυτό θα ανοίξει το δρόμο για πιο μακροπρόθεσμες ε, ε, παρεμβάσεις, ειδικά ε, σε ό,τι αφορά την ανοικοδόμηση. Επίσης πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσο η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των εργαλείων για την ε, σταθερότητα μπορεί να ενσωματωθεί στο μελλοντικό εργαλείο για την ε, ανάπτυξη, ίσω μέσω ενό συγκεκριμένου προγράμματο για τι ευαίσθητε χώρε. Χαίρομαι που το Κοινοβούλιο έχει τονίσει την ανάγκη για περαιτέρω ευελιξία. Αυτό είναι ένα τομέα ιδιαίτερη σημασία για τι εξωτερικέ δράσει και δεδομένη τη περιπλοκότητά του και τη αλλαγή που ε, υπάρχει στι συνθήκε, και αυτό αναφέρεται και στην κοινοποίηση της ε, ε, Κομισιόν, μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη ή θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να μην υπονομεύουμε την ε, προβλεψιμότητα για την απόδοση κονδυλίων για μεγάλες καταστροφές. Μεγάλες μεταφορές ποσών ή μεταφορές περιθωρίων θα ήταν ε, χρήσιμε όπως επίσης θα ήταν και η δυνατότητα ε, δεσμευμένων ε, κονδυλίων για ένα χρόνο να μπορεί να μεταφερθούν σε μετέπειτα χρόνια. Όπως ας πούμε η προκαταβολή των υποχρεώσεων των, του προϋπολογισμού. Αυτά, Πρόεδρε, από μένα θα σταματήσω εδώ και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Είμαστε ευέλικτοι και ε, αυτό ζητάμε και από το Συμβούλιο στις επόμενες δημοσιονομικές διαπραγματεύσεις. Αυτό εμείς το επιδεικνύουμε τώρα. Όλοι οι ομιλητές θα χρειαστεί να περιοριστούν σε τέσσερα λεπτά και έτσι θα καλύψουμε το χρόνο. Ο κύριος Κασουλίδης για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Πρώτα απ' όλα είναι σαφές ότι οι εξωτερικές σχέσεις θα έχουν πλέον δικό τους, ε, δική τους γραμμή στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Επίσης φαίνεται να μην υπάρχει άμεσος συσχετισμός μεταξύ της εξωτερικής μας πολιτικής και της στρατηγικής για το 2020. Άρα οι σχέσεις αυτές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν και το τι γίνεται στις εσωτερικές πολιτικές υπόθηκε ξεκάθαρα κατά τη συζήτηση για τη στρατηγική του 2020 ότι ό,τι ευθυγράμμιση γίνει μεταξύ πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και αυτής της στρατηγικής εκεί θα πρέπει τα ίδια να ισχύουν και για τη διάσταση των εξωτερικών σχέσεων. Όμω δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκλειστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση για άλλε προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω οι εξωτερικέ σχέσει. Το άλλο ζήτημα είναι η πείρα μας από το ισχύον πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτή μας έδειξε ότι από εξ αρχής οι οροφές ήταν πολύ περιοριστικές. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε εσφαλμένη εκτίμηση αρχικά σε σχέση με τις ανάγκες αυτής, τη της του κεφαλαίου. Θα πρέπει να, αυτού του τίτλου μάλλον. Θα πρέπει να είμαστε Βέβαια, ότι δεν θα συμβεί το ίδιο και στο ερχόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όπως και σε άλλους τίτλους πρέπει να έχουμε τον απαραίτητο βαθμό ευελιξίας Και αυτό ισχύει περισσότερο από άλλου τομείς για τις εξωτερικές ακριβώς σχέσεις με μεταβαλλόμενες ανάγκες και προτεραιότητες. Αυτές διασυνδέονται και με το μεταβαλλόμενο πολιτικό σκηνικό διεθνώ κρίσεις, ε, κατεπίγουσες ανάγκες. Αυτά απαιτούν διαφορετικές παρεμβάσεις κάθε φορά. Αλλά θα πρέπει να δοθεί έμφαση θα πρέπει να δοθεί έμφαση ακριβώ στον παράγοντα τη ευελιξία. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό θα το διαθέτουμε. Το ποσό που έχει προβλεφθεί για τι κατεπήγουσε ανάγκε έχει αποδειχθεί ότι δεν ήταν αρκετό καθόλου ε, ε, αρκετό για αυτές τις, για την κάλυψη των αναγκών για τις νέες ανάγκες χρηματοδότησης σε αυτόν τον τομέα, είδαμε τι συνέβη πρόσφατα με τα συνοδευτικά μέτρα που πρότεινε το Συμβούλιο. Για την μπανάνα εδώ θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι όλα αυτά θα διασφαλίζονται κατά τρόπο ώστε να μην υποφέρουν όμως αναλόγως άλλοι τομείς. Το Κοινοβούλιο πρόσφατα επέβαλε έτοιμα το ε, Ταμείο για την Ανάπτυξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριληφθεί στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια στη χρήση του. Και να βεβαιωθούμε και για το δημοκρατικό έλεγχο που ασκούμε. Τώρα, θα λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτήν την τοποθέτηση στην επόμενη πρότασή τη για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα υπάρχει αύξηση στην ε, διακυβερνητική χρηματοδότηση με το μέσο σταθερότητας και το καθεξής. Άρα η ανάγκη συντονισμού είναι περισσότερο από ποτέ μεγάλη. Αναγνωρίζεται ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διεθνές πολιτικό προσκήνιο δεν συνάδει με τα κονδύλια που προβλέπει για τη διεθνή βοήθεια. Όπω τα κονδύλια που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Παλαιστίνη. Εκεί δεν θέλουμε να διαδραματίσουμε σοβαρό ρόλο για την ανάπτυξη τη περιοχή αυτή. Τι μέτρα μπορούν να προβλεφθούν ώστε να αυξήσουμε και την αποτελεσματικότητα και την προβολή της παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί, προκειμένου να βελτιωθεί ακριβώς το κύρος της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τώρα ο Τάις Μπέρμαν τέσσερα λεπτά για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, η άποψη της Επιτροπής Ανάπτυξης, όπου ήμουν εισηγητής για το ζήτημα ακριβώ του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, υπήρξε σαφής. Εδώ θα επικεντρωθώ στο θεμελιώδες ζήτημα του τι διαβλέπουμε για το μέλλον της ερχόμενης επταετίας για την εξέλιξη ακριβώς των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαφές ότι υπάρχουν τρεις μεγάλες προτεραιότητες στις εξωτερικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για τις εσωτερικές της πολιτικές ισχύουν τα ίδια. Πρέπει να εργαστούμε στην κατεύθυνση της ειρήνης σε ένα κόσμο που να βασίζεται στο διάλογο και τις πολυμερείς συμφωνίες. Χρειαζόμαστε ε, μια τάξη που να βασίζεται στα δικαιώματα των πολιτών, ανδρών και γυναικών, ευάλωτων ομάδων όπω των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες και μια νέα τάξη που να βασίζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό για τους σπόρους, το περιβάλλον και την ε, αποκατάσταση της βιοποικιλότητας που έχουμε χάσει, δηλαδή προστασία από τις κλιματικές αλλαγές. Αυτά τα τρία βασικά ζητήματα, ειρήνη, δικαιώματα και βιωσιμότητα, αηφορία δηλαδή, είναι αυτά που θα πρέπει να μας οδηγούν στο σχεδιασμό των πολιτικών. Υπό αυτήν την οπτική γωνία, το Ευρωκοινοβούλιο, μάλλον η Ευρωπαϊκή το Ευρωκοινοβούλιο έχει να δραματίσει εδώ καθοριστικό ρόλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του πολίτε τη. Όμω, ποια είναι η θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση ω τώρα. Κατά την άποψή μου, είναι ένα 28ο δωρητή. Με πολύ ωραίε, αξιέπαινε εξωτερικέ δράσει, αλλά ποια είναι προστιθέμενη αξία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια θα μπορούσε. Αυτό βασίζεται στην, στο πόσο στενέ ε, είναι οι σχέσει συνεργασία μα ε, εντό Ένωση και το πολιτικό κύρο και την επιρροή που μπορεί να έχουμε. Χρειάζεται ένα συντονισμό και ένα υπεύθυνο συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, χωρί να επιζητούμε να είμαστε 28 δωρητή όπω όλοι οι άλλοι. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να επικεντρωθούν στο τι ε, κάνουν καλύτερα και πώ το πετυχαίνουν αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει να καθοδηγήσει τι κοινέ του προσπάθειε και προγράμματα που κάποιε φορέ ξεπερνούν τα όρια του ενό κράτου μέλου προγράμματα τα οποία μπορεί να τα φέρει πέρα καλύτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του ενδεχόμενου πολιτικού τη κύρου, τη ενδεχόμενη πολιτική τη επιρροή. Αυτό οδηγεί κατά την άποψή μου στην εξή δομή. Τα κράτη-μέλη ε, ε, επικεντρώνονται στι περιφέρειε, περιοχέ και τα θέματα που έχουν τη μεγαλύτερη εμπειρογνωμοσύνη και που είναι οι καλύτεροι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντονίζει τα προγράμματα των κρατομελών για να διασφαλίσει ότι οι διάφορε περιοχέ και όλα τα θέματα λαμβάνονται υπόψη και καλύπτονται και η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση είναι προφανώ ζωτική σημασία. Μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και την προβολή της πολιτικής αυτής εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αφήνει και περιθώριο ώστε οι τρεις αυτοί παράγοντες να ε, μπορέσουν να επικεντρωθούν στο εξή μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει έμφαση στις επενδύσεις, στη δημοκρατία, τον εκδημοκρατισμό, τα δικαιώματα των πολιτών, το κρατος δικαίου και τα προγράμματα για μεγάλες υποδομές, τα μεγάλα έργα υποδομών που δεν θα μπορούσαν μόνο τους να αναλάβουν τα κράτη-μέλη. Πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην υγεία και την εκπαίδευση, διατηρώντα το στόχο του 20% για τις δαπάνες σε αυτούς τους τομείς. Επίσης, πρέπει να επενδύσουμε σε έργα μεγάλης εμβέλειας, όπως την ε, ε, ενίσχυση των ασφαλιστικών πολιτικών για να παραμένουμε και λίγο εντό πραγματικότητας. Έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να είμαστε σοβαροί, μεγάλοι παράγοντες και σε άλλα ζητήματα χρηματοδότηση, όπω οι μικροπιστώσεις. Μπορούμε λοιπόν να συμβάλλουμε και σε άλλες περιπτώσεις όπως η ανακούφιση από φυσικές καταστροφές. Εδώ χρειάζεται αυτόνομο μέσο χρηματοδότησης διότι πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια δεν διασυνδέεται με τις πολιτικές επιλογές των μεν και των δε, αλλά είναι αμερόληπτη και ουδέτερη. Είναι πολύ σημαντικό η επιλογή αυτή να γίνει ευθύ εξ αρχής. Θα παραμείνω σε αυτά, διότι αυτέ είναι οι βασικέ μου παρατηρήσει. Θέλω να κάνω πολύ περισσότερε, αλλά ίσω μπορέσω να επανέλθω αργότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Γκέρενς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά τις δημοσιονομικές προοπτικές των επομένων ετών, το βασικό είναι το επίπεδο φιλοδοξίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πρέπει να δούμε αν θέλουμε να είμαστε μία οικονομική και εμπορική ε, Δύναμη, εάν θέλουμε να συνεργαστούμε με τις ε, ε, πιο φτωχές χώρες και ε, ε, να μπορέσουμε να τις βοηθήσουμε ε, να αναπτυχθούν και αυτό είναι ο στόχος της αναπτυξιακής βοήθειας. Πρέπει να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας. Έγινε μια μελέτη λοιπόν και είδαμε ότι από το 1980 στο 2011 το ΑΕΠ του, το διεθνές αυξήθηκε σε, ε, δε, κατά 19 δισεκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων ένα μόνο πήγε εις ε, τις φτωχές χώρες και όλα τα υπόλοιπα ανακατανέμηθηκαν μεταξύ των πλουσίων χωρών. Άρα εάν δεν υπάρχει εστίαση δεν μπορούμε να ε, κάνουμε πρόγραμμα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η παγκοσμιοποίηση μειώνει της ε, ε, μειώνει μεν τον ανταγωνισμό εξωτερικά αλλά την αυξάνει εσωτερικά διότι υπάρχουν χώρες οι οποίες ε, όπως η Ινδία και η Κίνα που δεν χρειάζονται καμία βοήθεια το πρόβλημά τους δεν είναι η δημιουργία πλούτου αυτήν την έχουν εξασφαλίσει αλλά μια σωστή κατανομή στο εσωτερικό και είναι και τους ευθύνη να απαντήσουν σε αυτό. Αλλά στην Αφρική, το Νότιο Σουδάν, ο Νίγηρας, η Μπουρκίνα Φάσο και άλλες ε, έχουν ε, ελάχιστο ΑΕΠ και πρέπει να βοηθηθούν. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε πολιτικές οι οποίες είναι δαπανηρές ή φτηνές. Αυτές οι οποίες δεν ε, κοστίζουν χρήματα, στις οποίες ανάφερα, είναι ε, ο πολιτικός διάλογος με τους Κινέζους, τους Ινδούς, να τους πούμε ότι δεν πρέπει εμείς να λύσουμε τα προβλήματά τους, είναι η μεγαλύτερη χρηματοδότηση στον κόσμο, άρα δεν χρειάζονται βοήθεια χρηματοδοτική. Αλλά ε, είμαστε υπέρ 0,7% ε, που έχει συμφωνηθεί διαθεσμικά. Ε, γιατί λοιπόν θα σπάσουμε αυτή την πολιτική τη στιγμή που έχουμε ακόμη τέσσερα χρόνια μέχρι να επιτύχουμε το στόχο για τον οποίο έχει δεσμευτεί η Ευρώπη. Τι μέτρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχει μια καλή δυνατότητα αρκεί να υπάρχει σωστή διακυβέρνηση αλλά συγχρόνως πρέπει να υπάρξει ε, μία αξιολόγηση του κινδύνου για να ξέρουμε ε, πόσο μπορεί να, τι θα γίνει αν υπάρξει κάποιο λάθος για να ξέρουμε ότι είναι έτοιμος ο μηχανισμός να αντεπεξέλθουμε. Έχουμε λοιπόν διάφορα ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσουμε. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο πρέπει να σας πω ότι η πολιτική μου ομάδα είναι υπέρ. Αλλά υπάρχουν συναφή ερωτήματα ε, σχετικά με ε, την χρήση του Αναπτυξιακού Ταμείου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που δεν έχουν ανταπαντηθεί. Δηλαδή θα αυξηθεί το ποσό που είναι διαθέσιμο διότι τώρα έχουμε το πλαφόν, το ανώτατο επίπεδο συγχύ ε, τη συνδρομή των κρατών ή το αναπτυξιακό ταμείο. Εάν όμως ε, ε, το αφαιρέσουμε από τους φόρους του ταμείου τότε θα είμαστε σε αντίφαση με όλες τις άλλες πολιτικές και επίσης πρέπει να δούμε εάν θα υπάρχει συνεργασία μεταξύ χωρών και, και Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Χρειάζεται αυτή η συμμετοχή, είναι ένα πρώτο που μπορούμε να αναπαράγουμε και αλλού και όσον αφορά την ευελιξία υπερθεματίζουμε. Θα είχα πολλά να σας πω ακόμη αλλά σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο και θα χρειαστεί να σταματήσω. Ευχαριστώ. Η Φρανσίσκα Μπράντερ τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι συνήθως στην ΑΦΕΤ με τον κύριο Πίμπαλξ. Έχουμε διάφορες ελλείψεις. Έχουμε πολλές ελλείψεις και το έχουμε εντοπίσει αυτό και για ε, όσα σχόλια έκαναν οι συνάδελφοι, την ανάγκη συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε τι γίνεται στις περιπτώσεις που κανεί αναποθέτει τι ελπίδες σε μια χώρα, όπως με την Τινησία και τη Γαλλία. Δεν ξέρω τι πετύχαμε εκεί. Α, νομίζω ότι αυτό που μας λείπει είναι ένα πραγματικό μέσο για την αναδιάρθρωση. Εδώ έχουμε ανθρωπιστική βοήθεια μεν, Έχουμε γενικότερα αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά δεν, μας, δεν έχουμε το ενδιάμεσο. Αυτό μας λείπει, ο ενδιάμεσος κρίκος. Θα πρέπει λοιπόν να πάρουμε ίσως κάτι από το μέσο σταθερότητας, από την αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά για την ώρα δεν αρκεί αυτό που έχουμε. Δεν θα έπρεπε να είναι εργαλείο αυτό αυτό αλλά εδώ χρειάζεται περισσότερη ευελιξία. Το χρειαζόμαστε. Και για το μέσο σταθερότητας θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντό λίγων μηνών, όχι να χρειάζονται χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο λίγο πιο ευέλικτο για την ε, ανάκαμψη, για στα πλαίσια του οποιοδήποτε μέσου προτιμήσουμε. Θα πρέπει να μην υπάρχει ιδιαίτερη πίεση για το μέσο σταθερότητας. Αυτό που μας λείπει είναι ένα πραγματικό μέσο που να αφορά τις αναδυόμενες χώρες πέρα από την επίσημη αναπτυξική βοήθεια. Εάν δεν θέλουμε λοιπόν να υπάρξουν κακές χρήσεις του, της αναπτυξικής βοήθειας πρέπει να προβλέψουμε ένα ειδικό μέσο. Δεν μπορεί αυτή, αυτός ο διάβλος να συντελεί στη βελτίωση των σχέσεών μας με τις αναδυόμενες χώρες. Και για τα ανθρωπιστικά δικαιώματα, το ευρωπαϊκό μέσο για τα δημοκρατικά δικαιώματα είναι ένα ποσό πολύ χαμηλό αυτό που του αποδίδεται. Βλέπουμε ότι έπρεπε να έχουμε χρησιμοποιήσει πολύ περισσότερα τα τελευταία χρόνια, γιατί είναι ένα μέσο που επιτρέπεται συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και του φορεί τη, χωρί αναγκαίο την συμφωνία του κυρίαρχου κράτου, του επισήμου κράτου. Αυτό λοιπόν θα συντελούσε σημαντικά στην πρόθεση των δημοκρατικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να αυξήσουμε τα σχετικά κονδύλια. Και για το μέσο σταθερότητα νομίζω ότι πρέπει λίγο να αποσαφηνίσουμε την εντολή από την άποψη την πολιτική. Δηλαδή, να υπάρχει διατησία και διαμεσολάβηση, να πηγαίνουμε στις ε, θερμές περιοχές, να προσφέρουμε και την πείρα και την εμπρογνωμοσύνη μας, αλλά πραγματικά να επικεντρωθούμε εκεί. Όχι να γίνει ένα εργαλείο που να έχει τόσο ευρία εντολή που τελικά να κάνει τίποτα και όλα μαζί να επικεντρώνεται στη διαμεσολάβηση, την βραχυπρόθεσμη πρόληψη κρίσεων και εκεί πάλι να υπάρχει ευελιξία. Πέραν αυτού, Νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε στην άσκηση των δικαιωμάτων δημοκρατικού ελέγχου, εφόσον θέλουμε ευελιξία. Οπωσδήποτε και εμεί θα πούμε ναι στην ευελιξία, αλλά μόνο αν υπάρχει δημοκρατικό έλεγχο. Αυτά τα δικαιώματα πρέπει να διασφαλιστούν. Αυτό έχει απασχολήσει τη συζήτηση μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπή ω τώρα. Και συμφωνώ και για τι παρατηρήσει για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη. Εφόσον καλυφθεί, βεβαίω θα πρέπει να ε, ξεπεράσει τα όρια των όσων είχαμε τώρα. Και μια τελευταία παρατήρηση για την άμεση στήριξη του προπολογισμού. Νομίζουμε ότι εάν υπάρξει τέτοια στήριξη άμεση για τον προπολογισμό, θα πρέπει στο μέλλον να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα ζητήματα και να υπάρχουν οργανώσει ε, τη κοινωνία των πολιτών που να μπορούν να ελέγχουν, ανεξάρτητοι οργανισμοί που να ελέγχουν πώ δαπανήθηκαν τα χρήματα αυτά, όπω στην Αφρική. Δεν έχουν δαπανηθεί σωστά τα κονδύλια. Ακόμη και στην άμεση στήριξη του προπολογισμού και ιδίω από ό,τι φαίνεται από του δείκτε των χωρών. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για τους τίτλους αυτούς που συζητούμε, θέλω να αναφέρω τρία πράγματα. Ποια είναι, ποιο είναι το όρομα και ποια η φιλοδοξία που έχει ο Επίτροπος για, ε, ε, για τον τομέα του. Μπορεί να μας δώσει κάποιες λεπτομέρειες. Επίσης, λογοδοσία, διαφάνεια ε, και φορολογική πειθαρχία. Ε, και επίσης ε, ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ε, μιλήσαμε πολύ σήμερα το πρωί για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων που θέτει ερωτήματα και για τους τρεις αυτούς τομείς και υπάρχουν πάρα πολλές έτσι πάρα πολλοί περιορισμοί ακόμη. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ε, προβλήματα. Πρώτον για, το, για τη χρηματοδότηση. Όσο εγώ ασχολούμαι με την Επιτροπή Προπολογισμού, τα κονδύλια που πάντα υπήρχαν ήταν λιγότερα από τις πολιτικές φιλοδοξίες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ανάπτυξη και στην επιρροή. Δεύτερον, προβλεψιμότητα. Είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα πρέπει να απαντά άμεσα και με συμπόνια σε κρίσεις όπως εξελίσσονται και εξελίσσονται όλο και πιο τακτικά πλέον, αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία. Ταυτόχρονα, ο τίτλος αυτός πάντα ε, τύχανε κριτικής από το ελεγκτικό συνέδριο λόγω έλλειψης ακρίβειας ε, και αποτελεσμάτων. Συμφωνώ λοιπόν ε, με αυτό που είπαν πολλοί συνάδελφοι ότι ναι, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει πολλή δουλειά που μπορεί να γίνει ακόμη. Ε, πρέπει να αναθεωρήσουμε λίγο την ε, διαδικασία και το πώς θα εξελιχθεί. Γενικώ, το 6% του προπολογισμού είναι ένα λογικό ποσοστό σε ό,τι αφορά την ποσότητα, αλλά θα ήθελα διαβεβαιώσεις σε ό,τι αφορά την ε, ποιότητα. Ευχαριστώ. Äh, η ποιότητα, η ποσότητα πάντα πρέπει να πηγαίνει χέρι-χέρι με την ποιότητα γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε το τι χρειαζόμαστε για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Δεν βλέπω κανέναν άλλον από την ΚΟΕ, δεν βλέπω κανέναν από την EFD, άρα να πάρουμε τον κύριο Έλλης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα συγκεκριμένο θέμα έχω να θέσω για τους έξι στόχους κλειδιά που έθεσε ο ε, Επίτροπος για τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές. Ναι, να παλύψουμε τη φτώχεια, ειδική σχέση με τις ε, γειτονικές χώρες. Αυτά ούτως ή άλλως είναι ε, πράγματα που συνεχίζουν να υφίστανται. Για τις βιομηχανοποιημένες χώρες είπε κάτι για στρατηγική σκέψη ο Επίτροπος. Εμένα πάντα με ανησυχούσε το γεγονός ότι έχουμε στρατηγικέ εταιρικέ σχέσεις ε, ακούμε πολλά από υψηλά ειστάμενους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εδώ, ε, αλλά δεν δεν ακούμε ποτέ για στρατηγική. Ακούμε μόνο για στρατηγικέ εταιρικέ σχέσει. Ε, εντάξει, επιλέγουμε εταιρικέ σχέσει με αυτέ τι χώρε επειδή είναι στρατηγικέ, αλλά τι ακριβώ σημαίνει αυτό ποτέ δεν έχουμε καταλάβει. Τι ακριβώ σημαίνει στρατηγική εταιρική σχέση και τι σημαίνει μακροπρόθεσμη στρατηγική για τι εξωτερικέ δράσει. So, Ωραία. Κοιτάω γύρω-γύρω να δω αν υπάρχει κάποιος που να θέλει να θέσει κάποιο ερώτημα. Ο Σάρλ και ο Γιώραν και μετά θα δώσουμε το λόγο στον Επίτροπο για να απαντήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ακούσαμε και κάποιες αδηγικές ανησυχίες από τον συνάδελφο για το συντονισμό μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, κρατών μελών για την ανταπτυξιακή βοήθεια. Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα που υπα, υφίστανται. Ε, για παράδειγμα, έχουμε τη συζήτηση, άλλο το μεγαλύτερο, κομμάτι της συζήτησης ε, σχετίζεται με, τους, με, τις, ε, με τις ε, γειτονικές χώρες. Την ενίσχυση για την προένταξη και τα λοιπά. Το πρωτεξιακό εργαλείο είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα αυτό. Υπάρχουν προβλήματα, να, τι να σας πω, Αίγυπτος, Γεωργία, Αρμενία, Αζερβαϊτζάν, Λευκορωσία, Μέση Ανατολή. Προφανώς αυτός ο τομέας των γειτονικών χωρών είναι πολύ ευαίσθητος και αν θέλουμε να επηρεάσουμε τα πράγματα πρέπει να έχουμε μεγάλη περισσότερους πόρους. Γίνεται επίσης συζήτηση για τη συνεργασία με πιο αναπτυγμένους χώρες, πολλοί το είπαν αυτό. Ε, γίνεται συζήτηση για τη χρηματοδότηση των ε, κλιματολογικών αλλαγών κτλ, κρίση, ε, διαχείριση καταστροφών κτλ. Όταν μιλούσαμε με τον κύριο Σάλιβαν, το είπα και πριν, Κοίταξα το χρηματοδοτικό πρόγραμμα για το 2012-2013, βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα, το γνωρίζω, αλλά έχουμε μία αύξηση επιπέδων όπως 5% για το 2012, 7% για το 2013 ε, που προβλέπεται από την Κομισιόν και τίποτα που να λέ, μιλάει για ανάπτυξη για μετά το 2013. Ερώτημα λοιπόν προς τον Επίτροπο. Πώς το βλέπετε υπάρχουν τομείς που να μπορούμε να μειώσουμε την προσπάθειά μας, υπάρχουν τομείς που να μπορούμε να ε, αυξήσουμε την ευρωπαϊκή ε, ε, προστιθέμενη αξία, υπάρχουν κρατημέλη που να μπορούν να προσθέσουν στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να είναι και τα ίδια αυτάρκη, γιατί ήδη υπάρχουν προβλήματα. Κάθε φορά έχουμε προβλήματα, κάθε φορά μιλούμε για τον τίτλο 4 και τώρα θα έχουμε ακόμη περισσότερα προβλήματα προβλήματα γιατί χρειάζεται πολύ περισσότερη ανάπτυξη. Η δική σας πρόθεση ποια είναι. Είναι σαφές το πρόβλημα, είναι υπαρκτό του να, να ε, συντεριαστούν οι προθέσεις με τους στόχους. Βλέπω ότι ε, πολλαπλασιάζονται οι συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο. Να δώσουμε το λόγο στο Σαρ πρώτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε να κάνω και εγώ τρία σχόλια. Πρώτα απ' όλα για την Κίνα, την Βραζιλία και την Ινδία. Εδώ πρέπει να προβλέψουμε ένα FES phasing out. Δηλαδή, οι χώρες αυτές μπορεί να φροντίσουν να έχουν μια τριμερή συνεργασία ε, και βορρά νότου νότου και ε, η Κίνα να γίνει αυτή που θα δορίζει και θα υποφελείται βεβαίως από τις επενδύσεις της βοήθειας αυτής. Ε, τώρα για το συντονισμό των 28 φορέων της Επιτροπής και των εθνικών κρατών μελών. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να βλέπουμε τι δημοσιονομικέ προοπτικέ και υπό την οπτική γωνία τη αύξηση που προβλέπεται έω το 2015. Τεράστιοι όγκοι θα εκταμιευθούν. Γιατί λοιπόν να μην έχουμε κοινό προγραμματισμό μεταξύ επιτροπή και ορισμένων κρατών μελών. Αυτό θα έπρεπε να γίνεται έφεξή, Τίποτε δεν θα ήταν αρκετό επιχείρημα για να μην κατευθυνθούμε σε μια τέτοια επιλογή. Πολλές φορές υπάρχουν κοινέ επιλογές μεταξύ κατωμέλων και των δικών σας υπηρεσιών. Μας το είπε και η κυρία Γιώργη από την Ευρωπαϊκή Γεώργαν, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπουμε να υπάρχουν ε, απαιτήσει και βάσει συνθήκη να υπάρχει συντονισμό καλύτερο μεταξύ ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικών Πολιτικών. Συντονισμό λοιπόν και στο επίπεδο του προπολογισμού. Αυτό προκρίνουμε. Τώρα ο Ε, Ευχαριστώ. Έχω δύο ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα έχει σχέση με την αναπτυξιακή συνεργασία και με την συνοχή, διότι πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές, γιατί ναι μεν είμαστε σημαντικοί ως Ευρωπαϊκή Ένωση για την αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά πρέπει να μπορούμε να ανανεωνόμαστε. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα προγράμματα σαν μέρος της αναπτυξιακής συνεργασίας. Έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο ε, να εμβαθύνει γιατί πιστεύω ότι ε, θα μπορούσαμε ε, στον τομέα αυτό να λειτουργήσουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης πέραν αυτού σχετικά με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν ε, σχετικά με τα προγράμματα αυτά και το τι μπορούμε να κάνουμε ως συνεργασίες με τη Ρωσία παραδείγματος χάρη που αντιμετωπίζουμε προβλήματα διότι τα προγράμματα αυτά έχουν σχέση με την αναπτυξιακή συνεργασία με τις ανάπτυξη χώρες. Θα μπορέσουμε και στα προγράμματα αυτά να συμπεριλάβουμε τα ε, εντόπια ε, προγράμματα διότι τα διαφορετικά πρόκειται για παρεμφερή θέματα. Ωραία, τώρα ο Ράιμαρντ Μπέγκε και μετά θα απαντήσει ο Επίτροπος. Ευχαριστώ, θέλω απλώ να συμπληρώσω αυτά που ελέγχθησαν διότι αυτά που είπαν οι συνάδελφοι είναι μία ευκαιρία να κάνουμε μία πολύ διεξοδική ανάλυση των μέσων που χρησιμοποιούνται, δηλαδή ε, ε, ενίσχυση από τον προϋπολογισμό. Ε, παρόλο που βλέπω ότι η Αναπτυξιακή Επιτροπή έχει προβλέψει μια κάποια χρηματοδότηση για εκπαίδευση και ανατροφή και θα ήθελα να ξέρω αν όλο το θέμα το οποίο είχαμε ξεκινήσει πριν από τρία χρόνια μέσω ενός ταμείου που όμως δεν είχε στρατηγικές επιπτώσεις ε, διεθνώς ή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως μπορεί ε, να αναθεωρηθεί κατά τρόπον ώστε να χρησιμοποιηθεί σύντομα. Θα ήθελα λοιπόν να έχω κάποια σχόλια επί του θέματος από τον Επίτροπο. Επίσης μιλάμε για αναπτυξιακή βοήθεια και βλέπουμε ότι σε ορισμένα κράτη έχουμε βελτιώσει σε σχέση με την προηγούμενη εικόνα που είχαμε και μπορούμε ε, ίσως να αναθεωρήσουμε αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πόσο ε, ε, πώς αντιμετωπίζει την χρηματοδότηση ε, των ορισμένων προγραμμάτων χωρίς να έχει εξετάσει τις κοινωνικές επιπτώσεις. Δεν θα πρέπει να προχωρήσει έτσι η Επιτροπή και γι' αυτό βλέπουμε στη σελίδα 15 της συνόψεως του πώληση Department D όπου ε, βλέπουμε ότι ε, στην ε, αναπτυξιακή βοήθεια υπάρχουν και άλλα, άλλες δυνατότητες τις οποίες χρειαζόμαστε. Πρέπει λοιπόν να δούμε εάν τα περιθώρια που υπάρχουν στις διάφορες κατηγορίες επαρκούν, αν χρειαζόμαστε νέες δυνατότητες μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης για να μην χρειάζεται να αντιδρούμε πάντοτε κατά περίπτωση το οποίο δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων. Έχουμε δηλαδή ε, εδώ ανάγκη για ε, ένα νέο πλωστάσιο που θα μας επιτρέψει να αντιδρούμε πιο αποτελεσματικά και πιο γρήγορα. Ωραία. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος Πίμπαλς τώρα παρακαλώ να απαντήσει. Έχετε λίγο περισσότερο χρόνο διότι όλοι ήταν πολύ πειθαρχημένοι και μπορείτε τώρα να μιλήσετε άνετα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω από τις πιο συγκεκριμένε ε, απαντήσεις και μετά θα θίξω τα ευρύτερα ζητήματα που έθιξαν οι βουλευτές για τη διαχείριση της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσφατα το συζητήσαμε στην Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών, βασιζόμενη στην έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου, για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ανάπτυξη και τα ανάλογα κονδύλια. Εδώ πρέπει να πω ότι το ποσοστό σφάλματος για το Ταμείο αυτό είναι 2% και 25% το ποσοστό επιτυχίας. Άρα πρέπει να πω ότι πετυχαίνουμε ακριβώς ό,τι και με τις εσωτερικές μας πολιτικές ε, και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η τάση, η θετική τάση. Έπειτα για τη διαφάνεια. Όλα μας τα προγράμματα είναι εξαιρετικά διαφανή. Πρόσβαση υπάρχει στο διαδίκτυο για όλους, όπως αναφέρθηκε στη συζήτηση. μπορεί ο καθένας να πάει και να, στην ιστοσελίδα και να συμβουλευτεί ό,τι θέλει. Επίση, υπάρχει μια πρωτοβουλία για τη διαφάνεια τη βοήθεια από την πλευρά τη Επιτροπή. Οπότε, είμαστε εκτεθειμένοι σε κάθε είδου κριτική και σχόλιο. Αυτό είναι κάτι που το φροντίζουμε, μην ανησυχείτε. Και για τους ε, εταίρους μας ε, στην βοήθεια πρόσφατα ε, επίκυνται επίσημες ανακοινώσει και νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο τα πάμε πάρα πολύ καλά. Τώρα για τις γενικές μας ανάγκες. Εάν κοιτάξουμε πώς είναι διεθνώς η κατάσταση σήμερα, ας πάρουμε το επιτυχές δημοψήφισμα στο Νότιο Σουδάν. Δεν θα ήταν αυτό δυνατό χωρίς τη δική μας οικονομική στήριξη. ή λόγου χάρη να υπάρξει ειρήνευση στη Σομαλία. Ε, ε, ε, ούτε αυτό θα ήταν δυνατό χωρίς τη δική μας την παρέμβαση. Κάποιοι είναι ιδιαίτερα επικριτικοί ακριβώ γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτελεί έργο. Επίση, είμαστε ε, σαφώ από του μεγαλύτερου δωρητέ στην αναπτυξιακή βοήθεια, ακόμη και αν είμαστε στα επίπεδα του 0,5% ακόμη. Κάνουμε πολλά σε πολλέ χώρε για τη στέγαση, για την εκπαίδευση. Χώρε ε, ε, τείνουν να πετύχουν του στόχου τη χιλιετία γιατί εμεί τα χρηματοδοτούμε. Πρέπει λοιπόν να επενέσω την αναπτυξιακή μας πολιτική. Είναι πολύ ισχυρή εδώ η πολιτική μας και σε συγκεκριμένε καταστάσει που προέκυψαν από το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο. Τώρα, με κάθε σεβασμό για τι συζητήσει σα για το δημοσιονομικό πλαίσιο και τι δυσκολίε του προπολογισμού, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ καλά εξοπλισμένη με εύρωστε δυνατότητε απόκριση. Εμεί είμαστε σταθεροί, άλλοι έχουν ε, ε σκαμπανεβάσματα. Όμω όχι, εμείς είμαστε σταθεροί και πολλές φορές βασιζόμαστε στις μεμονωμένες δράσεις βεβαίως των 100 μελών, όμως στη Νέα Υόρκη πρόσφατη σύνοδος βασίστηκε στην παρέμβαση του, ε, της, ε, στην παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε πλέον προκοδότηση με ένα δις για τέτοιες ε, πρωτοβουλίες. Είναι πολλά τα παραδείγματα που θα μπορούσα να αναφέρω εδώ και για τα πιο συγκεκριμένα ζητήματα που τέθηκαν για τη στρατηγική του 2020. Πιστεύω σαφώς ότι δεν θα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός των μέσων της εξωτερικής πολιτικής ε, με μεταξύ των αρμοδιοτήτων των διαφόρων επιτρόπων. Υπήρξα επίτροπο ενέργεια. Βλέπω τι γίνεται τώρα με τα κονδύλια τη εξωτερική πολιτική που μπορεί να αφορούν την ενέργεια. Όμω, συμφωνώ ότι όλε αυτέ οι πτυχέ πρέπει να συμπεριληφθούν ε, σε μια κοινή προσέγγιση. Και εγώ πιστεύω ότι η εξωτερική πολιτική πρέπει να ε, καλύπτεται εδώ όπω και προ την άσκηση του δημοκρατικού ελέγχου. Για την ευελιξία είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας βαθμός ευελιξίας και συντονισμός μαζί με έλεγχο. Αυτό θα πει δημοκρατικός έλεγχος νομίζω. Αυτού του είδους η άσκηση ελέγχου θα επιτρέψει να δούμε κατά πόσον υπάρχει αποτελεσματικότητα μέσω της διαφάνειας. Τώρα, για τον προπολογισμό του ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, είπατε θέση μου, είναι θέμα ελέγχου. Τα πάει καλά το Ταμείο αυτό. Και λειτουργεί για αρκετό διάστημα. Αλλά θα έπρεπε βεβαίω το όλο σύστημα να επιτρέπει έλεγχο και από το Κοινοβούλιο. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι λένε ότι μπορούν να υπάρχουν αντιρρήσει, ε, αδιαφάνειε. Σαφώ έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα δημοκρατικού ελέγχου. Ω επίτροπο, πάντοτε μου αρέσει ο έλεγχο είναι δύσκολο μένα, αλλά αν περάσει κανεί τη δοκιμασία του ελέγχου, είναι πολύ πιο ισχυρό μετά. Διότι καλύπτεται. Δεν είναι πλέον εκτεθειμένο ω μεμονωμένο πολιτικό παράγοντα. Για οποιοδήποτε σφάλμα ή παράβλεψη μπορεί να συμβεί. Θέλουμε λοιπόν ισχυρότατο έλεγχο ή δυνατόν για τον επιτόπια επιρροή που μπορεί να ασκήσουμε. Νομίζω η νέα μας, το νέο μας αρχιτεκτόνημα μπορεί να μας το επιτρέψει αυτό. Διότι αν δούμε την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κάθε πρόγραμμα από μόνο του είναι πολύ καλό. Το θέμα είναι τι γενικώ πετυχαίνουμε με τη στρατηγική μας προς μια συγκεκριμένη χώρα και τι επιρροή, τι αποτέλεσμα πετυχαίνουμε τελικά με αυτό το νέο αρχιτεκτόνημα που είναι πολύ ισχυρό και καλύπτει πάρα πολλούς διαφορετικούς τομείς θα έχουμε πλέον και την ισχυρή παρουσία της Αντιπροέδρου και με την ΤΕΦΚΟΜ μπορούμε να είμαστε πολύ συνεπείς, σαφείς και να αναλαμβάνουμε και τις ευθύνε μας σε συγκεκριμένες πολιτικές ε, καταστάσεις ε, όπως προκύπτουν στην πραγματικότητα. Είναι λοιπόν σημαντικό λογικό αυτό και αν δούμε τι πρόσφατε απαντήσει τη επιτροπή, είμαστε όλο ένα περισσότερο απαντούμε στο πώ απαντούμε, πώς επιτυγχάνουμε αποτελέσματα. Τι πέτυχαν οι δράσεις μας για την ειρήνη και τη σταθερότητα, τι πέτυχαν για συγκεκριμένες ε, ε, υποθέσεις. Έχουμε πετύχει πολλά και νομίζω σοβαρά αποτελέσματα. Θα σκεφτώ πολύ προσεκτικά τα σχόλιά σας, διότι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι είναι η Ένωση, κύριε Μπέρμαν, ένας 28ος δωρητής. Όμως είναι σημαντικά τα κονδύλια που αποδίδουμε και έχουμε και ολοκληρωμένες ε, πολιτικές. Προσπαθούμε λοιπόν να υπερκαλύψουμε, να γίνουμε πιο σημαντικοί από του 27 δωρητέ εμεί ω 28. Αυτό πολλέ φορέ συμπεριλαμβάνει μέχρι και δικαιώματα εργασιακά, βιώσιμη ανάπτυξη. ε, αξιοπρεπού βίου. Νομίζω ότι τα επιδιώκουμε όλα αυτά. Πρέπει πραγματικά να προβλέψουμε περισσότερα κονδύλια για την ανάπτυξη. Πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο σε συγκεκριμένους στόχους και για να τον αντίκτυπο στην καλή διακυβέρνηση πρέπει βεβαίως να το εξακολουθήσουμε αυτό. Τώρα, το μέσο σταθερότητας είναι πραγματικά ένα μέσο που θα πρέπει να γίνει ένα μέσο ταχείας απόκρισης σε συγκεκριμένες καταστάσεις που προκύπτουν και ξεπερνούν τα όρια της απλής ανθρωπιστικής βοήθειας. Θα πρέπει να επαναδιατυπώσουμε την εντολή και να την περιχαρακώσουμε, αν μπορώ να το πω έτσι. Υπάρχουν μέσα αναπτυξιακή βοήθεια προ αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν αποδίδουν τα απαιτούμενα τα αποτελέσματα. Θα πρέπει λοιπόν πολιτικώ να αναλάβουμε κάποιε ευθύνε για το ECI συν και κάποια από τα ερωτήματα που τέθηκαν για τι στρατηγικέ εταιρικέ σχέσει νομίζω ότι η Κίνα, η Ινδία ή η Βραζιλία είναι διαφορετικές από χώρες με μέσα εισοδήματα, από άλλες χώρες με μέσα εισοδήματα. Όμω το βλέπω και δύσκολο να προσφέρουμε εμεί βοήθεια σε χώρε που οι προσφέρουν βοήθεια σε τρίτες χώρε. Ναι, μπορούμε να συνεργαστούμε και στην ανάπτυξη, αλλά εδώ έχουμε μια σαφή συμφωνία θα πρέπει να τους πούμε κάντε εσείς αυτά για να κάνουμε εμείς τα άλλα. Αυτό θα ήταν στρατηγική σχέση. Για τους, απο... για τους άνθρακα λόγω χάρη Εκεί χρειάζονται συγκεκριμένα τεχνολογικά μέσα. Θα μπορούσαμε να έχουμε κοινά συμφέροντα. Ή για την ανταλλαγή φοιτητών. Αυτό είναι στρατηγική σημασία και για μα και θα έπρεπε να, υπάρξει στήριξη, να υπάρχει στήριξη από χρηματοδοτικά μέσα, αλλά αυτό δεν είναι κλασική αναπτυξιακή στήριξη. Θα μπορούσε να καλύπτεται από ένα μέσο ICI-SIN ή κάποιο άλλο νέο μέσο. Θα μα πει κάποιο γιατί δίνεται αναπτυξιακή βοήθεια στην Κίνα. Όχι, γιατί είναι προ το δικό μα όφελο η συνεργασία με την Κίνα για συγκεκριμένε προτεραιότητε. Είπατε εκπρόσωπο αυτή τη στιγμή συζητά τι θεωρήσει με τα κράτη-μέλη και το πώ βλέπουν τι στατηγικέ μα αυτέ σχέσει. Όπω με τη Ρωσία. Είναι ένα στατηγικό εταίρο η Ρωσία. Πρέπει να βρούμε σημεία ε, συνεννόηση με τη Ρωσία και έχουμε κάθε συμφέρον να συνεργαστούμε μαζί τη. Αλλά αυτό δεν είναι αναπτυξιακή βοήθεια, ούτε αναπτυξιακή συνεργασία. Για τον προπολογισμό το είπε ότι απαιτείται έλεγχος, περισσότερος έλεγχος, αυστηρότερος, αυστηρή εφαρμογή των κανόνων και αποτίμηση με συγκεκριμένους δείκτες Βλέπουμε τι ευθύνε βαρύνουν τι χώρε όταν μιλάμε για εκταμείευση κονδυλίων από τον προπολογισμό. Βλέπουμε τι γίνεται με τα προγράμματα ανακούφιση από τη φτώχεια ή με τα προγράμματα για την ανάκαμψη. Πρέπει λοιπόν εδώ να τα λάβουμε όλα αυτά σαφώς υπόψη μας από πολιτικές άποψεις. Ε, μιλάμε για ένα μέσο που θα μπορούσε να χρησιμοποιείται όταν μπορεί να προσφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα και εγγυήσεις. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι, ε, ότι το χρησιμοποιούμε σε χώρες δημοκρατικές που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Τινησία που κάποιο ανέφερε. Εκεί δώσαμε στήριξη στο λαό της χώρας. Όμως... Ε, αναγκάζομαι να τηρώ αμυντική στάση διότι μπορώ να σας πω ότι παρακολουθήσαμε πώς ε, δαπανήθηκαν τα χρήματα, αλλά υπάρχουν και πολιτικά πρόοπτα και αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Για τον δημοκρατικό έλεγχο θα επανέλθω. Ναι, πρέπει να είμαστε συνεπείς με τη συνθήκη, προφανώς. για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Υπάρχει ένα πράσινο βιβλίο, μια πράσινη βίβλος τέλο πάντων ακριβώς για αυτό το θέμα. Από την δική μου την προοπτική τι βλέπω. Όταν υποσχόμαστε σε μια κυβέρνηση λόγω χάρη στήριξη των απολογισμού, είναι σημαντικό να λειτουργούμε ω Ένωση των 27. Αυτό είναι ένα τομέα όπου πραγματικά θα μπορούσα να δω κοινοτική προστιθέμενη αξία. Εκεί έχουμε τις σοβαρότερες επενδύσεις. Βιώσιμη ενέργεια ή γεωργία και επισητιστική ασφάλεια. Εκεί υπάρχουν ανάγκες. Θα μπορούσαμε λοιπόν στρατηγικώς να παρεμβαίνουμε σε τομείς όπου τα κράτη-μέλη θα είχαν λιγότερη προβολή αν παρενέβαιναν. Πρέπει λοιπόν πάντοτε να το έχουμε, να το λαμβάνουμε αυτό υπόψη. για τους δρόμους είναι καθοριστική σημασία για την IT και την ε, ανάκαψη της χώρας αυτής. Δεν μπορούμε όμως να έχουμε τα αποτελέσματα τώρα, πρέπει να περιμένουμε μια διετία. Και εκεί θα φανεί όλη μας η προβολή και η αξία των αποτελεσμάτων μας. Αυτό θα μας προσφέρει προβολή. Αλλά κάποιος μπορεί να λάβει και τη δύσκολη δουλειά του να πει στο Συμβούλιο. Ε, τα κράτη με ζητούν με ένα από εδώ και από εκεί περικοπέ, αλλά το ζήτημα είναι το γενικότερό μα αρχιτεκτόνιμα. Τώρα το είμαστε αποτελεσματικοί. Ξέρετε ότι ο στόχος είναι το 0,7% του ΑΕΦ για την ανάπτυξη. Τελικά απαιτούνται περισσότερα κονδύλια συνήθω. Όμω δεν μιλούμε για επιβάρυνση των φορολογουμένων εδώ. Χρειαζόμαστε μια κοινή πλατφόρμα ώστε να έρχονται επενδύσει μέσα στι χώρε. Και πηγαίνουν εκεί που, υπάρχουν, που υπάρχει καλή διακυβέρνηση, σεβασμό του θεσμικού πλαισίου και κάποια στήριξη στις γραμμέ τι πιστοτικές. και εξερεύνηση νέων δυνατοτήτων. Εκεί δεν υπήρξαμε πολύ αποτελεσματική. Κίνα κίνδία στήριξαν εταιρείε που πήγαν στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Εδώ υπάρχουν δυνατότητε ανάπτυξη, μιλάμε και για δύσκολε χώρε, αλλά πρέπει κανεί να σκεφτεί πώ μπορεί να εμπλέξει περισσότερο τον ιδιωτικό τομέα στι χώρε αυτέ. Διότι οι συγκεκριμένε επενδύσει βοηθούν αυτέ τι χώρε να βελτιώσουν την φορολογική του δίκηση ή να σέβονται περισσότερο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε λοιπόν εδώ κάποια προσπάθεια, αλλά δεν είναι και τόσο απλή μαθηματική η παρέμβασή μας. Τώρα για αύξηση ή μείωση μιλήσατε. Εδώ αγωνιζόμαστε για τις εξωτερικές σχέσεις, όπως για όλους τους τομείς που χρειάζονται χρηματοδότηση. Θα ήταν άδικο να πω ότι δεν χρειαζόμαστε περισσότερου πόρους. Οι ανάγκες και τα κατεπήγοντα σε σχέση με τη δημοκρατία έχουν αυξηθεί. Ε, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι ανάγκες έχουν αυξηθεί. Πόσα μπορούμε να σας δώσουμε, αυτό είναι θέμα εξισορρόπησης του τι θα μπορούσαμε να δαπανίσουμε για την εξωτερική πολιτική και πώς θα μπορούσαμε να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα για την Ινδία και άλλες χώρες και τον κοινό προγραμματισμό. Μιλήσαμε για το πώς συντονιζόμαστε με τα κράτη-μέλη και τις, ε, νομίζω ότι συνολικά οι εξωτερικές σχέσεις των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν βελτιωθεί. Χθες, λόγου χάρη, ο Βρετανός υπουργό που επισκέφθηκε τη Σομαλία μου είπε εγώ θα αφήσω τα θέματα της εκπαίδευσης της Σομαλίας σε εσάς γιατί έχετε αναλάβει. Κάποιες φορές να έχουμε υπόψη ότι τα κράτη-μέλη παίρνουν πολύ σοβαρά τι δικέ μα προσπάθειε ω Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί πετυχαίνουμε και καλά αποτελέσματα. Μα σέβονται λοιπόν και σε ορισμένου τομεί είμαστε και πιο ισχυροί. για την ε, νέε ιδέε για την ενέργεια. Νομίζω ότι αυτό είναι πραγματική προτεραιότητα. Χωρί παροχή ενέργεια δεν υπάρχει ανάπτυξη. Εάν δείτε τι ευρωπαϊκέ χώρε, όπου υπήρξαν σοβαρέ επενδύσει στην ενέργεια από τι κυβερνήσει ω επιτοπλίστων, που ιδιωτικοποιήθηκαν και ε, τελικά μιλάμε για ιδιωτικέ εταιρείε, όπου, λοιπόν, όπου υπήρχε στήριξη για προγράμματα καθαρή ενέργεια, υπήρξε πρόοδο το να έχουμε αποψήλωση των τροπικών δασών ή πυρκαγιέ. είναι κάτι που δεν το θέλουμε για τι αναπτυσσόμενε χώρε. Εκεί χρειάζονται στήριξη και είναι έτοιμε χώρε αυτέ να υιοθετήσουν καθαρότερε λύσει για την ενέργεια. Για τον κύριο Μπέγκε, για την επιστημιστική ασφάλεια. Θα υπάρχουν και θετικέ ειδήσει εδώ και αρνητικέ. Οι καλέ είναι ότι κατά την κρίση παρεμβήκαμε και βοηθήσαμε κάποιε χώρε να ξεπεράσουν την κρίση. Το κακό νέο βέβαια είναι ότι προσπαθήσαμε να κατανείμουν ανάλογα με τι ανάγκε των κρατών, αλλά χάθηκαν πολλά κονδύλια επειδή ξεκίναγαν από διαφορετικά θεσμικά όργανα. Τι θέλουμε, απλώς να περιορίσουμε τον αντίκτυπο από την αύξηση των τιμών. Έχουμε όμως μακροπρόθεσμη στρατηγική για την επιστημιστική ασφάλεια και το μέσο διευκόλυνση για τα τρόφιμα ε, είναι μια προσπάθεια που θα πρέπει να εξακολουθήσει. Αλλά δεν πρέπει να κάνουμε παντού την, ε, μια κοινή προσπάθεια. Δεν μπορούμε. Θα ήταν αδύνατο να είμαστε παρόντε παντού. Όλοι τα θεσμικά όργανα συμφωνούν, Επιτροπή, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο. Δεν είναι δυνατόν. Χρειάζεται και συγκεκριμένη εμπειρογνωμοσύνη και να ληφθούν υπόψη και διοικητικέ δαπάνε που χρειάζονται περικοπή. Πολλέ φορέ από τα προγράμματά μα το 50% είναι έλεγχοι. Οπότε πολλά χάνονται γιατί βρισκόμαστε σε πολλού τομεί ε, παρόντε ταυτόχρονα. Δεν μπορούμε να τα περιορίσουμε. Στην εξωτερική πολιτική λοιπόν πρέπει να έχουμε σαφώ σχεδιασμένε στρατηγικέ. Στην ανάπτυξη είμαστε παρόντε. Με του στρατηγικού μα εταίρου, με την ύπατη εκπρόσωπο έχουμε έντονη δράση τη. Εκφράζεται και συνεχώ και πρέπει όμω να καταφέρει να εμπλέξει και τα κράτη-μέλη τα οποία συνηθίζουν να ενδιαφέρονται ιδιαίτερω για ένα συγκεκριμένο στατικικό εταίρο. Ε, Όμω έχουμε τα πράσινα βιβλία. Ε, τα κρατημέλη πρέπει να σέβονται τη στατική αυτή την κοινή και είπατε εκπρόσωπο θέλει στήριξη για αυτή την στρατηγική. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε, κινούμαστε και βλέπω εδώ να υπάρχουν ε, πραγματικές αλλαγές. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία Σημειώνουμε όλα σας τα σχόλια, όλες σας τις προτάσεις. Νομίζω ότι αυτή είναι μόνο η αρχή της συζήτησης. Δεν τέλειωσε τίποτα εδώ. Αύριο θα συζητήσουμε στο κολέγιο των Επιτρόπων. Θα τους αναφέρω λοιπόν και τις δικές σας θέσεις από τη σημερινή συζήτηση. Ähm, λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Επίτροπε διότι δεν απαντήσατε ίσως σε όλες τις ερωτήσεις όπως μας είπατε ότι ίσως δεν απαντήσατε επαρκώς την ερώτηση του James Ellis αλλά έχουμε πάντοτε την ε, δυνατότητα σε ορισμένα θέματα να υπάρξει μία γραπτή απάντηση. Ε, είχατε πολλές ερωτήσεις τις οποίες απαντήσατε και αντιληφθήκατε ότι υπάρχει μία μεγάλη Υπότιτλοι AUTHORWAVE στήριξη δηλαδή ότι ε, τα κράτη-μέλη ε, διαφημίζουν περισσότερο την πολιτική σας από ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και είναι πολύ πιο εμφανή τα αποτελέσματα αλλά όσον αφορά τα μέσα μας είπατε ότι έχετε υποκαταστήσει τα μέτρα μπορείτε να μας πείτε σε ποια μέτρα έχετε επέμβει γιατί θα μπορέσετε έτσι να μας βοηθήσετε όχι τόσο πολύ για να έχουμε κάτι μέχρι τον Ιούνιο αλλά όταν ε, θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση για τον όγκο του προπολογισμού μας αυτές οι πληροφορίες θα είναι πάρα πολύ χρήσιμες να τις έχουμε γραπτός. Τώρα υπάρχει ακόμη η σύνοψη του Σαλβαντόρ Γκαρίγκα και ελπίζω ότι αυτό θα το πετύχουμε μέχρι ότου τελειώσει η ώρα της Επιτροπής μας. Πρόεδρε, πολύ σύντομα να κάνω κι εγώ μια περίληψη των προτάσεων που μας έκανε ο κύριος Πίμπαλξ. Νομίζω ότι όντως υπάρχει συνένεση στην Επιτροπή αυτή ότι οι εξωτερικές δράσεις είναι πολύ ιδιαίτερες, ειδικά στα, υπό το φως της κρίσης που έχει ε, επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τα υπάρχοντα προβλήματα, όπως ας πούμε την χρόνια υποχρηματοδότηση στις εξωτερικές σχέσεις, καθώς επίσης και το γεγονός ότι οι δεσμεύσεις δεν ε, ε, αντικατοπτρίζουν αυτά που είχαμε φανταστεί ειδικά αν δείτε την ε, κρίση που υπάρχει στην άλλη πλευρά της Μεσογείου. Πρέπει να έχουμε ασφαλείς μορφές χρηματοδότησης. Αυτή λοιπόν η ιδιαιτερότητα των εξωτερικών δράσεων ε, νομίζω ότι είναι αντιληπτή από όλους στην Επιτροπή. Είναι σημαντικό να υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος. Το είπε ο Επιτρόπος Ανάπτυξης το είπε και ο συνάδελφος κ. Μπέρμαν, μας έδωσε και αριθμητικά στοιχεία για την κακοδιαχείριση και την μη χρηστή ε, χρήση των κονδυλίων. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα που πρέπει να το έχουν υπόψη όλα τα κρατημέλη και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Ανεξάρτητα από την στρατηγική για το 2020, πρέπει να υπάρξει μια σύνδεση μεταξύ της αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών και των στόχων ε, του τομέα της ενέργειας παρόλα αυτά υπάρχει μια έτσι, πολύ περιορισμένη σχέση μεταξύ της στρατηγικής 2020 και των εξωτερικών δράσεων. Χρειάζεται διαφοροποίηση, μια διαφοροποιημένη προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική στα επόμενα χρόνια. Και ο συνάδελφος κύριος Ashworth είπε ε, σαφώς ότι οι ποσότητες των κονδυλίων μπορεί να είναι μεν επαρκείς, αλλά είναι δύσκολο πολλές φορές να ε, αιτιολογήσουμε το υψηλό επίπεδο που αυτές έχουν. Είναι σημαντικό λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει διαφάνεια, γιατί προς το παρόν δεν υπάρχει και τόση. Υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους χάνουμε το, το όραμα, χάνουμε την, ε, τη διαφάνεια που θα έπρεπε να υπάρχει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πρέπει να μπει στο μικροσκόπιο αν θέλουμε να ε, αξιολογήσουμε την ε, ανάπτυξη όλων αυτών των δράσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό πρέπει να γίνει σε όλους τους τομείς. Κυρίως γιατί η προστιθέμενη αξία δεν προκύπτει μόνο από συγκεκριμένε δράσεις στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων, αλλά υπάρχουν και εσωτερικά προγράμματα που μπορούν να ε, που μπορούν να δώσουν αποτελέσματα, ας πούμε προγράμματα για τη μετανάστευση, προσπάθεια ε, αύξηση των εσόδων υπάρχουν πολιτικές, ε, υπάρχουν πολιτικές σε κοινωτικό επίπεδο ε, που έχουν και επίπτωση στις εξωτερικές δράσεις. Σε σχέση τώρα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, το οποίο μπαίνει στον προπολογισμό, ε, νομίζω ότι αυτή η ιδέα θα γίνει σιγά σιγά αποδεκτή. Βέβαια είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις στο ανώτατα επίπεδα το, του προπολογισμού που δίδεται στις εξωτερικές δράσεις. Και για την ευρωπαϊκή, εξωτερική, για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, το ξέχασα και νομίζω ότι πρέπει να το πω γιατί είναι σημαντικό. Το Ηνωμένο Βασίλειο είπε ότι θα αποσυρθεί από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει ξεκινήσει να ασχολείται. Θα αφαιρέσει δηλαδή, θα αποσυρθεί το, η εθνική αντιπροσωπεία του Ηνωμένου Βασιλείου από το συγκεκριμένο πρόγραμμα γιατί το ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια κράτη-μέλη λοιπόν εκχωρούν την αρμοδιότητα ε, του να συμμετάσχουν σε συγκεκριμένα προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν αυτό γίνει κανόνας, θα πρέπει αυτοί οι τομεί να έχουν τους απαραίτητου τους πόρους. Σε κοινοτικό επίπεδο μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Είναι λοιπόν σημαντικό να δούμε ότι ένα πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από 27 εθνικά αντίστοιχα προγράμματα. Δεν μπορούν λοιπόν να αποσύρονται με τέτοιο τρόπο τα κονδύλια από το ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, ένα άλλο που είπε ο Επίτροπος είχε να κάνει με την ε, επιρροή της ε, Επιτροπής ΣΥΟΡ και τις ε, επιπτώσεις που αυτή θα έχει στις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές. Είπε ότι στο μέλλον θα χρειάζεται μια πολυετής προσέγγιση σε αντίθεση με τα όσα συμβαίνουν τώρα. Σημειώνουμε την πρόταση αυτή και θα το δούμε στο ιστορικό της Επιτροπής μας. Σίγουρα θα εξασφαλίσουμε μέσω αυτής της πρότασης καλύτερο συντονισμό των πολιτικών που σχετίζονται με τις εξωτερικές ε, υποθέσεις, με πολιτικές που σχετίζονται με εσωτερικές υποθέσεις, γιατί είναι καλός, καλή ιδέα να μην υπάρχει αυτός ο κατακαιρματισμός και να υπάρχει μια πιο ενιαία προσέγγιση. Τίθεται το ερώτημα εάν οι εξωτερικές πολιτικές θα πρέπει να αποτελούν τμήμα Τη αναπτυξιακή πολιτική που υπάρχει στο εσωτερικό επίπεδο ή αν θα πρέπει να παραμείνουν εξωτερικές πολιτικέ. πολιτικές. Έχουμε το ICI-SIN, το οποίο χρησιμοποιείται στην αναπτυξιακή πολιτική, θα χρησιμοποιείται μάλλον στην αναπτυξιακή πολιτική στο μέλλον, στις σχέσει μας με τρίτε χώρες, ειδικά με αναπτυσσόμενε χώρε. Κάποιοι συνάδελφοι θεωρούν ότι πρέπει να αλλάξουμε τα τάκ για τις χώρες ε, που, των χώρε τις αναπτυσσόμενες χώρες που έχουν ε, μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορέσει να επιτύχει τους αναπτυξιακούς της στόχους για αυτούς τους, ε, για αυτά, για αυτούς τους τομείς, νομίζω ότι θα είναι σημαντικό για, όλους τους, για όλες τις χώρες. Ευχαριστώ. Hier wieder δεν λειτουργούσε το μικρόφωνο της Προέδρου και έτσι δεν ακούσαμε το σχόλιο